Euh, Αγαπητοί συνάδελφοι, η ώρα είναι αρκετά πρωινή. Σας εύχομαι καλή σας μέρα. Καλώς ήρθατε στην συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής μας Επιτροπής. Σημείο πρώτο της ημερήσιας διάταξης σας προτείνω να εγκριθεί η ημερήσια διάταξη χωρίς καμία τροποποίηση. Σημείο 2 της ημερήσιας διάταξης, ανακοινώσεις της Προέδρου, θα ήθελα να σας ενημερώσω για κάποια σημεία. Πρώτον, να σε επενθυμίσω ότι σήμερα το απόγευμα, από τις 3 το μεσημέρι και μετά, θα έχουμε μία ανοιχτή διάσκεψη των Προέδρων, δημόσια για όλα τα μέλη, παρουσία του Χέρμαν Βαν Ρομπέι, προκειμένου να ενημερωθούμε για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της προηγούμενης εβδομάδας, και για πρώτη φορά επιτρέπεται στις κοινοβουλευτικές επιτροπές να συνεδριάσουν από τις 3 το μεσημέρι και μετά. Χωρίς δηλαδή τροποποίηση, έτσι λοιπόν και εμείς θα συνεδριάσουμε σήμερα το απόγευμα χωρίς καμία τροποποίηση. Θα ξεκινήσουμε δηλαδή στις 3 το μεσημέρι με μια κοινή δημόσια ακρόαση με, το, με την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξη Πέθρου όσον αφορά τις εργασιακές και κοινωνικές συνθήκες στον τομέα της γεωργίας θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Αντιπρόεδρο Τόμας Μαν, ο οποίος αποδέχθηκε να προεδρεύσει τις προεδρίες της ε, ακρόασης αυτής. Δεύτερη τώρα ανακοίνωση. Η Ιώνα Καμαρσούγιου, μετά από πάρα πολλά χρόνια εργασίας ιδιαίτερα επαγγελματική στα πλαίσια τη ε, κοινοβουλευτική μα επιτροπή ω ε, εθνικό εμπειρογνώμονα, αποσπασμένο πρόκειται να φύγει από την υπηρεσία αυτή τη κοινοβουλευτική μα επιτροπή. Λυπούμαθε πάρα πολύ για την αποχώρηση αυτή και λίγο αργότερα στις 12.30 συγκεκριμένα το μεσημέρι μπροστά από την αίθουσα αυτή μπορούμε να πιούμε ένα αποχαιρετιστήριο ποτό. Και σε αντάλλαγμα θα έχουμε τον Ζώταν Πετών, ο οποίος θα εργαστεί στα πλαίσια της γραμματείας της Κοινοβουλευτικής μας Επιτροπής. Ήδη έχει ξεκινήσει από την 1η Μαρτίου να εργάζεται για την Επιτροπή μας και είμαι σίγουρος ότι στα πλαίσια της Επιτροπής μας θα καταφέρει να αναπτύξει ακόμα περισσότερο τα διαπραγματευτικά επαγγελματικά του ταλέντα και να αναπτύξει όλο και περισσότερο τις ανθρώπινες σχέσεις στα πλαίσια ενός συλλογικού πνεύματος. Όλα αυτά στο πλαίσιο της γραμματείας της Επιτροπής μας. Σημείο 3 της ημερήσιας η διάσκεψη της ε, Επιτροπής Παρακολούθησης από την Επιτροπή Προεπολογισμών για την Ανεργία των Νέων θα γίνει στις 21 Μαρτίου από τις 12.30 έως τις 2 ε, το μεσημέρι στην αίθουσα 3Ε3 του άλλου κτηρίου. Όλα τα μέλη της Επιτροπής μας είναι προσκεκλημένα να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση αυτή και δεδομένου του θέματος που διάλεξε τελικά η Επιτροπή Προϋπολογισμών ελπίζω ότι θα έχουμε πολλά μέλη από τη δική μας την Επιτροπή. Ιδίως τα μέλη της Επιτροπής μας τα οποία ασχολούνται με την ανεργία των νέων. Ελπίζω ότι θα καταφέρουν να συμμετάσχουν σε αυτή τη συνεδρίαση. Δυστυχώς εγώ δεν θα μπορέσω να παραστώ γιατί θα είμαι στο Παρίσι. Επαφή μου όμως σε εσά προκειμένου να είστε εκεί πέρα παρόντες. Τέταρτη ανακοίνωση. Ένα νέο σημείο στο οποίο θα αναφέρομαι πλέον συνεχώς από εδώ και πέρα στα πλαίσια των ανακοινώσεων. Ουσιαστικά θα ήθελα να ενημερώνω την ολομέλεια της Επιτροπής μας όσον αφορά το κόστος της δερμηνίας. Στην τελευταία συνάντηση των συντονιστών είχα πει ότι η μη χρησιμοποίηση της δερμηνίας ενώ είχε ζητηθεί η καθυστερημένη ακύρωση έχει ένα κόστος για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μία γλώσσα κοστίζει στις Βρυξέλλες περίπου 880 ευρώ. Και ξέρετε ότι στις αποστολές το κόστος αυτό είναι ακόμα υψηλότερο. Για τις συνεδριάσεις που γίνονται μεταξύ συγητών, σχεδόν εισηγητών ή κάποιες άλλες άτυπες συνεδριάσεις, ζητάτε από τους βουλευτές να περιορίσουν τα αιτήματα διερμηνίας, εκτός και να αυτή απαιτείται, και να ενημερώνουν ε, ταχύτατα αμέσω τη γραμματεία σε περίπτωση που δεν θα καταφέρουν να συμμετάσχουν στη δεδομένη αυτή συνεδρίαση. Η κάθε φορά που η συνεδρίαση αυτή πρέπει να ακυρωθεί στα πλαίσια της διαφάνειας είπε ότι από εδώ και εξή στην αρχή κάθε, διερμη... κάθε συνεδρίασης επιτροπής μας κάθε περίπτωση διερμηνίας που δεν χρησιμοποιείται ή ακυρώνεται θα αποτελεί αντικείμενο ανακοίνωσης ενημέρωσης από μένα. Πρέπει να σας πω ότι από τις 4 έως 8 Μαρτίου είχαμε περιπτώσεις ε, διερμηνίας που δεν χρησιμοποιήθηκε, ιδίως όσον αφορά τις, ε, τη συνεδρίαση των σκιωδών εισηγητών για τους αποσπασμένους εργαζομένους, όπου ακυρώθηκε τελικά, μάλλον δεν χρησιμοποιήθηκε διερμηνία στα πολωνικά, μολονότι είχε ζητηθεί, γιατί εν τέλει ακυρώθηκε η συνεδρίαση αυτή. 880 ευρώ χάθηκαν έτσι. Επίση, στη συνεδρίαση με τον Επίτροπο Αντόρ είχε προβλεφθεί διερμηνία στα αγγλικά, τα γαλλικά, τα ουγγρικά και τα γερμανικά. Η συνεδρίαση αναβλήθηκε και εν τέλει έλαβε χώρα χωρίς διερμηνία. Και πάλι 880 ευρώ επί 3, επί 4 λέει Πρόεδρο, τέλο, ο τριμερής διάλογος για την ευθύνη του κράτους σημαία. Πάλι και εκεί πέρα κάποια μέλη είχαν ζητήσει δερμηνία στα γαλλικά και εν τέλει δεν εμφανίστηκαν. Επομένως δεν χρησιμοποιήθηκε πάλι γαλλική δερμηνία. 880 ευρώ. Η γραμματεία έχει συντάξει έναν κατάλογο ιδιαίτερα συμπαθητικό βέβαια που δεν κατονομάζει εκεί τους βουλευτές. Από εδώ και πέρα θα ζητήσω από τη γραμματεία να κατονομάζει και τους βουλευτές που ζητάνε και δεν χρησιμοποιούν διερμηνία, δεν εμφανίζονται τελικά. Πέμπτο σημείο συνακοινώσει. Ξέρετε ότι η συνεδρίαση της Επιτροπής μας μεταδίδεται μέσω του διαδικτύου. Αν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις για τις ανακοινώσεις αυτές, περνάμε στο σημείο 3 της ημερήσιας διάταξης, όπου θα συζητήσουμε τις τρεις συμβαστικές τροπολογίες για την έκθεση, για το σχέδιο γνωμοδότησης μάλλον, Τη κυρία Σουγκουρανό όσον αφορά την ετήσια έκθεση σχετικά με την πολιτική ανταγωνισμού. Πρόκειται για μια γνωμοδότηση όπου αρχικά είχαν κατατεθεί 23 τροπολογίες. Η τροπολογία αυτή απευθύνεται προς την Επιτροπή ΕΚΟΝ όπου η συγητής είναι ο Αντολίν Σάντσες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Uh, Όπως ε, είπατε, έχουμε πολλές τροπολογίες. Ευχαριστώ θερμά τους συντάκτες των τροπολογιών. Δύσκολο ήταν να καταλήξουμε συμβαστικές τροπολογίες, αλλά τελικά ε, καταφέραμε να συντάξουμε τρεις συμβαστικές τροπολογίες για τις παραγράφους 5, 6 και 17, ε, τις οποίες θα υποστηρίξει και το ΕΛΚ. Για τις τροπολογίες 4 και 7, μία παρατήρηση. Συμφωνώ απόλυτα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να έχει ένα ολόκληρο κεφάλαιο για τα αποτελέσματα της πολιτικής ανταγωνισμού στην απασχόληση. Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με την τροπολογία 13, αλλά μπορούμε να δεχτούμε την 14. Επίσης, αποσύρω τις δικές μου τροπολογίε 12 και 17. Με δύο λόγια λοιπόν, αυτή είναι η θέση του ΕΛΚΑ, κυρία Πρόεδρε, σε ό,τι αφορά την γνωμοδότηση για το θέμα αυτό κυρία Στάινρουκ. Ευχαριστώ. Εκ των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών και του συναδέλφου Λούντβιχ που δυστυχώς απουσιάζει, συμφωνούμε με τις ε, συμβαστικές τροπολογίες και ευχαριστώ θερμά τον ε, συντάκτη της γνωμοδότησης για την ε, συνεργασία που είχαμε. Θέλει άλλος κανείς το λόγο παρακαλώ. εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κυρία Γουόνς. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ στο πλαίσια της συζήτησης για την ετήσια έκθεση για τον ανταγωνισμό. Έχω κάποιες προτάσεις. Ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη έχουν συμφωνήσει για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική του 2020 για ανάπτυξη που θα περικλείγεται, θα αποκλεί και θα είναι ευφύης και βιώσιμη και πιστεύω ότι αν ε, ε, υλοποιήσουμε τους στόχους του 2020 θα έχουμε σημαντική θετική επιρροή στην ανταγωνιστικότητα χωρίς κόστος για το φορολογούμενο. Η πολιτική ανταγωνισμού δεν εξασφαλίζει μόνο τη σωστή συμπεριφορά των εταιριών, αλλά καθορίζει και το κατάλληλο πλαίσιο για τις κυβερνήσεις ώστε να αξιοποιήσουν τις ε, ελάχιστα, ελάχιστα δημόσια έσοδα και να τα χρησιμοποιήσουν στις πιο αποτελεσματικές, ε, στους πιο αποτελεσματικούς τομείς. Έτσι θα αντιμετωπιστούν ε, οι οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις με τον καλύτερο τρόπο. Πέρυσι ανακοινώσαμε ότι θα ξεχρονίσει τον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων και θα διευκολύνει τη χορήγηση ενισχύσεων που είναι σωστά στοχοθετημένε, σχεδιασμένε και εντοπίζουν τι αδυναμίες αγορά και του κοινού στόχου, όπω είναι η έρευνα, η πράσινη οικονομία και η σωστή ενίσχυση που δεν θα στρεβλώνει την αγορά. Τώρα, σε ό,τι αφορά μερικέ τροπολογίε του σχεδίου γνωμοδότηση. Οι κανόνες κρατικών ενισχύσεων ήδη προβλέπουν δυνατότητα ε, συνδρομής προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ένα στόχο του εξυγχρονισμού των κρατικών ενισχύσεων είναι η ενίσχυση αυτή να συμβάλλει στην υλοποίηση των στόχων ε, για το 2020. Και πολλά μέτρα τη αγορά εργασία εκπίπτουν ε, το πεδίο εφαρμογή αυτών των στόχων. Τα κράτη-μέλη έχουν τη διακριτική ευχαίρεια να κρίνουν κατά πόσο θεωρούνται αυτά τα μέτρα ω ενισχύσει. Θα μπορούσε να είναι ε, μέτρα που δεν θα είναι ενίσχυση αλλά θα είναι συμβατή ενίσχυση ή θα προσπαθούν να συμφιλειώσουν, να λάβουν καλύτερη υπόψη το θέμα και τη σχέση προσφοράς και ζήτησης. Επίσης, σε ένα σημείο η διατύπωση δεν είναι πολύ σαφής, αλλά στον κανονισμό για τις ε, συλλογικές εξαιρέσεις ε, ήδη προβλέπουμε κάποιους κανόνες για τέτοιου είδους ενισχύσεις. Σε ό,τι φορά τις τροπολογίες, η τροπολογία 8 το πακέτο μας ό,τι αφορά τι κρατικές ενισχύσεις είναι πλήρες. Σε ό,τι αφορά το άρθρο 14 της συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα τέλη του 2011 ενέκρινε μία ανακοίνωση ό,τι αφορά το πλαίσιο ποιότητα για τις κοινοφελείς υπηρεσίες τη Ευρωπαϊκή Ένωσης. Το πακέτο SEE e αφήνει μεγάλο περιθώριο λίγο λοιπόν, στα κράτη-μέλη για να ε, τελειοποιήσουν και να, εξο... και να εξυγχρονίσουν αυτές τις ενισχύσει. Για παράδειγμα, η κοινωνική, κοινωνική στέγαση εκπίπτει και μάλιστα χωρίς ε, ανώτατο όριο για το ποσό. Για να είναι μια τέτοια ενίσχυση SJE θα πρέπει να πληρεί τι κοινωνικέ ε, κοινωνικές ανάγκες, να αφορά κυρίως από όρους πολίτες και λιγότερο προνομιούχων ε, στρωμάτων της κοινωνίας που δεν μπορούν να αγοράσουν ε, μια οικία με τους όρους αγοράς. Έτσι θα αντιμετωπιστούν τα προβλήματα σε ό,τι φορά τις κοινωνικές αιστείες. Και μπορούν φυσικά τα κράτη-μέλη να κοινοποιήσουν τα προβλήματα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να γίνει μια συζήτηση. Σε ό,τι αφορά τι ιδιωτικοποίησει, είμαστε ουδέτεροι σε ό,τι αφορά την ιδιοκτησία, την κυριότητα των εταιριών. Οι διαδικασίε ιδιωτικοποίηση όμω ίσω περιλαμβάνουν κάποια θέματα κρατικών ενισχύσεων. Εν τη αυτή περίπτωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να ενημερώνεται και να αναμειγνύεται σε πρόωρο στάδιο. Σε ό,τι αφορά τι τροπολογίε 18, 19 και 20, οι κανόνε κρατικών ενισχύσεων είναι υπέρ τη μετάβαση σε μια οικονομία με χαμηλή χρήση άνθρακα και ιδιαίτερε κατευθυντήριε γραμμέ για τι περιβαλλοντικέ ενισχύσει και τον κανονισμό για τι ομαδικέ εξαιρέσει ό,τι αφορά τι κρατικέ ενισχύσει, αλλά και τι ε, Κατευθυντήριε γραμμέ ε, για το περιβάλλον και την ενέργεια. Δεν υπάρχει ανάγκη εδώ εξαίρεση, γιατί οι κανόνε ε, δίνουν ε, μεγάλε ευκαιρίε για κρατική υποστήριξη. Οι κανόνε κρατικών ενισχύσεων ήδη στηρίζουν την έρευνα και τι επενδύσει στην έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη. Οι κατευθυντήρια γραμμέ και, και ο κανονισμό για τι ομαδικέ εξαιρέσει στηρίζουν κάποιο σχέδιο έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη. Οπότε κρίνουμε ότι δεν χρειάζεται εκεί πέρα περαιτέρω εξαιρέσει. Και τέλος, για την τροπολογία 22, για την ε, πιθανή παραβίαση δικαίου ανταγωνισμού όταν ε, ε, το κράτος μέλος αρνείται να πωλήσει ένα εργοστάσιο που θα κλείσει. Δεν ξέρουμε αν το κλείσιμο δημιουργεί στρέβλωση ανταγωνισμού σε αντίθεση με την πώληση. Ε, αν μια εταιρεία θέλει να κλείσει ένα εργοστάσιο και έχει προηγουμένως συμφωνήσει ε, με άλλες εταιρείες για το κλείσιμο και το προτιμά από, το, από την πώληση, τότε ίσως όντως δημιουργηθεί στρέβλωση του ανταγωνισμού. Σε, εν τη αυτή περιπτώσει θα δικαιούνται να παρεμβαίνουν είτε οι κρατικές ρυθμιστικές αρχές είτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η εταιρεία που κλείνει το εργοστάσιο φυσικά θα πρέπει να έχει δεσπο, δεσπόζουσα θέση και το κλείσιμο να ισοδυναμεί με κατάχρηση δημόσιας, δε, δεσπόζουσας θέσης. Επίσης θα πρέπει να δούμε αν η περιο, ο περιορισμός παραγωγής από το κλείσιμο ενός εργοστασίου βλάπτει τους καταναλωτές και να εξεταστεί η κατάλληλη πολιτική. Σε μερικές περιπτώσεις ίσως το κλείσιμο ε, δημιουργεί έλλειψη στην προσφορά ε, κάτι που πλήττει του καταναλωτέ, ιδιαίτερα όταν δεν υπάρχει αντιστάθμισμα από άλλε εταιρείε που μπορούν να καλύψουν αυτή την. Ε, το κενό τη ζήτηση που δημιουργήθηκε. Το κενό τη προσφορά, συγγνώμη, που δημιουργήθηκε. Ο Ζητώ συγγνώμη που άργησα σήμερα το πρωί. Είχα μία άλλη συνεδρίαση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, αλλά δεν μπορώ να τον ευχαριστήσω για την καλή συνεργασία, διότι μόνο την περασμένη εβδομάδα πήρα αυτά τα μπόρεσα να ακολουθήσω. Συνεπώς αυτή τη στιγμή ε, δεν μπορώ να πω τίποτα επειδή πρόσφατα κοίταξα ε, όλο το θέμα. Έριξα μια ματιά στις τροπολογίες, ορισμένες κατά τη γνώμη μου είναι επικοδομητικές και άλλες όπως είπε η Επιτροπή δημιουργούν προβλήματα όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις. Ακόμα και αν συμφωνώ με την γενική υπευθυνότητα των επιχειρήσεων, νομίζω ότι πρέπει να είναι θελοντική, αφορά κάτι το συγκεκριμένο και κατόπιν η εικόνα των επιχειρήσεων, το να παροτρύνουμε τις βέλτικες πρακτικές. Νομίζω ότι αυτό δεν ενισχύει την ανταγωνιστικότητα. Τώρα, ως προς τις τροπολογίες που αφορούν τους ορισμούς, SG και τα λοιπά, η Επιτροπή ήδη ε, το, γνωρίζει ποια είναι η εκτίμηση των κρατών μελών. Αυτό αφορά τους κανόνες που έχουν σχέση με τις κρατικές ενισχύσεις. Το θέμα είναι πολύ ευαίσθητος πιστεύω και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Ε, αυτό που μας χρειάζεται είναι επιπλέον υποστήριξη, αλλά συγχρόνως να εξασφαλίζουμε την ομαλή λειτουργία της αγοράς. Δεν πρέπει να υπάρχει προστατευτισμός. Πρέπει λοιπόν να βρούμε την καλύτερη, την καλύτερη ισορροπία. Ευχαριστώ. Υπάρχουν άλλοι που θέλουν να μιλήσουν. Ο κύριος Μάν. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον εισηγητή επειδή κατόρθωσε να μειώσει τον ρυθμό των ε, τροπολογιών, πράγμα το οποίο καταδεικνύει ότι η έκθεση ήταν καλή, επειδή δεν χρειάστηκε να διορθώσει πολλά. Το άρθρο 3 το οποίο αναφέρθηκε, ε, για μας πρέπει να υπάρχει κοινωνική υπευθυνότητα από μέρους των επιχειρήσεων το ζητούμενο είναι να δούμε κατά πόσον το μέτρο αυτό θα είναι υποχρεωτικό ή εθελοντικό. Πρόκειται λοιπόν για μια ευθύνη που αναλαμβάνουν οι ευθύνε. Συνεπώ γίνεται εκουσίω. Συνεπώ νομίζω ότι είναι περιττό να αναφερθεί ο δεσμευτικό χαρακτήρα. Αυτά όσον αφορά την τροπολογία. Λοιπόν, η τροπολογία 3 τώρα, για την 22. Εδώ έχουμε ορισμένες δυσκολίες. Αυτή η τροπολογία της έχουμε. Αναφέρεται στην υποχρέωση πώληση της επιχείρηση ορισμένε περιπτώσεις. Πρέπει να το διευκρινίσουμε. Υπάρχει πιθανή παραβίαση ε, του δικαίου περί ανταγωνισμού. Η θέση μας είναι διαφορετική σε σχέση με τις κυρίες Μπερέσε. Άλλωστε, η Επιτροπή εξήγησε ποια είναι η γραμμή που ακολουθούμε. Αυτή είναι η θέση μας. Διότι υπήρχαν ορισμένοι δισταγμοί, αντιδράσεις και πρέπει συνεπώς να δούμε ποια, ποιο είναι το νομικό πλαίσιο στο οποίο κινείται μια επιχείρηση για να μην υπάρχουν πιθανές παραβιάσεις ε, των κανόνων του ανταγωνισμού, όπως υπόθηκε εδώ. Φαντάζομαι ότι θα υπάρξει συμφωνία στην ομάδα μας. Ευχαριστώ. Υπάρχουν άλλοι που θέλουν να μιλήσουν. Σε σχέση με τα όσα είπε ο κύριος Τόμας Μάν, ε, σχετικά με τις ε, συμβαστικές τροπολογίες και τα σχόλιά σας για τις άλλες τροπολογίες που καλύπτονται από τις συμβαστικέ λύσεις. Ποια θα είναι η θέση σας ως εισηγητή. Ήδη τον έφερα. Αναφέρθηκα στις άλλες τροπολογίες. Το μόνο που μπορώ να πω τώρα είναι ότι έλαβα υπόψη τις παρατηρήσεις που έγιναν από τους συναδέλφους και θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ απόλυτα με τη θέση του κυρίου Μαν για την τροπολογία 22. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο είχε προκαλέσει και πολλές συζητήσεις στις προηγούμενες συνεδριάσεις μας. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο. Πολύ καλά. Συνεπώς θα ψηφίσουμε τη γνωμοδότησή σας αύριο προκειμένου η Οικονομική Νομισματική Επιτροπή που θα τοποθετηθεί αύριο να το λάβει υπόψη. Όχι, θα ψηφίσουμε αργότερα στη συνεδρίαση της ψηφοφορίας. Ερχόμαστε τώρα στο σημείο 4 της σημερινής διάταξης και δίνω το λόγο στη συνάδελφό μας Τσάμπα Σόγκορ. Στον συνάδελφό μα, με συγχωρείτε, Τσάμπα Σόγκορ, για να παρουσιάσει τι πέντε τροπολογίε, σημαστικέ τροπολογίε που ε, κατατέθηκαν με βάση τις 41 τροπολογίες για την εκπαιδευτική και επαγγελματική κινητικότητα των γυναικών στην Ευρώπη. Πρόκειται για ένα σχέδιο γνωμοδότησης που έχει σχέση με την έκθεση της Λίξα Ροντζούλη στα πλαίσια της Επιτροπής Γυναικών για το ίδιο θέμα. Προτού όμως προχωρήσω, θα ήθελα να καλωσορίσω την αντιπροσωπεία της Ένωσης ΟΝΣΕ, Ισπανική Ένωση Υποστήριξης μέσω ε, για την εργασία και την ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία, συγκεκριμένα των τυφλών, μια οργάνωση που κάνει εξαιρετική δουλειά και την καλωσορίζω θερμότατα αυτή την αντιπροσωπεία στην Επιτροπή μας. Όπως είπα, θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Σόγκορ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη βοήθειά σας και να ευχαριστήσω και τους ε, συντάκτες των τροπολογιών για τις 42 τροπολογίες που κατέθεσαν, που προσπάθησα να συμπηλήσω σε πέντε συμβαστικέ τροπολογίες. Θεωρώ ότι καταφέραμε να συμπεριλάβουμε στο έγγραφο όλα τα σημαντικά σημεία την κρίση της φτώχειας, τη βελτίωση της παροχής ε, υγειονομικής περίθαλψης, τη, το γεφύρωμα του μισολογικού χάσματος, ε, η ενίσχυση της επαγγελματικής κινητικότητας, η ενίσχυση των αναπήρων γυναικών, η ε, μεταβίβαση των δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης και ούτω καθεξής. Ήταν πολύ στενή η συνεργασία μας με την αρμόδια καθήλια επιτροπή, την Επιτροπή των Γυναικών και θεωρώ ότι η γνωμοδότησή μας είναι πολύ μεστή και αξιόλογη. Ευχαριστώ. κυρία Μπλινκεβιτσούτε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ε, συντάκτη της γνωμοδότησης και τους ε, σκιώδης ηγητές των λοιπόν ε, πολιτικών ομάδων για την διαλλακτικότητα που έδειξαν σε ό,τι αφορά την σύνταξη συμβαστικών τροπολογιών. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε τη συμπερίληψη των γυναικών και την ενσωμάτωσή τους στην αγορά εργασία, στη διαβίου κατάρτιση και την πρόσβασή τους σε όλες τις δυνατότητες που δίνει η εκπαίδευση και η αγορά εργασία. Φυσικά θα πρέπει να δημιουργήσουμε και κάποιες ε, θεμελιώδεις προϋποθέσεις για την ένταξη των γυναικών στην, ε, στα διά, στους διάφορους τομείς της ζωής και την πρόσβασή τους ε, σε επαγγελματική κατάρτιση και άλλου είδους κατάρτιση. Επίσης, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το πρόβλημα των χαμηλότερων συντάξεων που λαμβάνουν οι γυναίκες και το, τη δυσμενή μεταχείριση των πιο ηλικιωμένων γυναικών θα υποβάλω κάποιες προφορικές τροπολογίες και έτσι αντί για γυναίκες μετανάστες να λέμε γυναίκες που αποδημούν στην Ολοδαπή. Moving abroad. Άλλωστε και η έκθεση της Επιτροπής Γυναικών αυτό τον όρο περιλαμβάνει. Θα καταθέσω τροπολογίες ζητώντα διαγραφή κάποιων υποζημιώσεων που θεωρώ ότι μετά τις συμβαστικές τροπολογίες είναι περιτές. Ευελπιστώ ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία και θα μπορέσουμε τελικά να υπερψηφίσουμε τις συμβαστικές τροπολογίες και τη γνωμοδότηση εν γέννη. Ε, ε, Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν θα ήθελα να επαναλάβω τα όσα είπαν οι προαλήσαντες. Ουσιαστικά συμφωνώ μαζί τους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε, που φαίνεται άλλωστε και στις πέντε συμβαστικές τροπολογίες τις οποίες καταλήξαμε και τις οποίες προφανώς υποστηρίζουμε. Ωστόσο υπάρχουν κάποιες τροπολογίες τις οποίες δεν μπορούμε να στηρίξουμε. Πρώτον, τροπολογία παριθμών 7. Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω την τοποθέτηση που έχουμε στην τροπολογία αυτή. Τι ακριβώς λέμε εδώ πέρα. Μιλάμε για ευέλικτες αγορές εργασίας. Επίσης δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με την τροπολογία 36. Οι δύο αυτές τροπολογίες δεν καλύπτονται από τις συμβαστικές τροπολογίες. Πιο συγκεκριμένα, η τροπολογία 36 είναι σωστή ως προς το περιεχόμενό της αναφέρεται ουσιαστικά στην επανένωση των οικογενειών. Έχουμε όμως μια οδηγία στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ασχολείται ακριβώς με το ζήτημα αυτό. Πρόκειται λοιπόν για ένα ζήτημα που αφορά περισσότερο τις εργασίες της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται εμεί κάθε φορά που συντάσσουμε μια έκθεση να επαναλαμβάνουμε πράγματα που έχουμε πει σε άλλε οδηγίε. Αυτό δεν βελτιώνει την, το κείμενο. Προκειμένου να έχουμε μια καλύτερη διατύπωση επίσης, η δική μου πολιτική ομάδα στηρίζει την ε, τροπολογία που έχουν υποβάλει οι σοσιαλιστές Όσον αφορά όμως την τροπολογία 22 συγκεκριμένα, θεωρούμε ότι η αρχική τροπολογία ήταν καλύτερη από αυτή στην οποία τελικά καταλήξαμε. Επίσης, θεωρούμε ότι δεν θα πρέπει να στρεβλώσουμε το περιεχόμενο του ψηφίσματος. Αναφερόμενοι στο πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο, Πρόεδρο, σας ευχαριστούμε για την παρέμβασή σα. Δεν θέλει να πάρει κανείς άλλο το λόγο, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όχι. Επομένω, ο κύριο Σόγκορ για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε να ευχαριστήσω και τους προλύσαντες για τις παρατηρήσεις τους. Σήμερα το απόγευμα μπορούμε να συνεδριάσουμε για να διευθετήσουμε τις τελευταίες αυτές διαφωνίες που υπάρχουν. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, ολοκληρώνουμε το σημείο αυτό. Θα ψηφίσουμε για την γνωμοδότηση αυτήν αύριο και τον Απρίλιο θα ψηφίσει η Επιτροπή Γυναικών για αυτή την έκθεση. Φτάνουμε στο σημείο 5 της ημερήσιας διάταξης και θα ήθελα να δώσω το λόγο στην Ανθέα Μακιντάιρ, για να μας παρουσιάσει τις συμβαστικές της τροπολογίες όσον αφορά τις 12 τροπολογίες που είχαν αρχικά κατατεθεί για την γνωμοδότησή της. Γνωμοδότηση για την οποία ακολουθούμε τη διαδικασία συνδεδεμένης επιτροπή σε σχέση με την Επιτροπή Περιβάλλοντος όσον αφορά τους βασικούς κανόνες ασφαλείας για την υγειονομική προστασία από τους κινδύνους που προκύπτουν από την έκθεση σε ιονίζουσες ακτινοβολίες. Κυρία Συγκήτρια, έχετε το λόγο. 40 τροπολογίες, με συγχωρείτε λέει πρόεδρο, 40 τροπολογίες είχαν αρχικά κατατεθεί για το σχέδιο γνωμοδότησή σα βάσει των 12 αρχικών τροπολογιών που είχατε εσεί καταθέσει. Δεν υπάρχει συμβαστική τροπολογία και σα δίνω ευθύ αμέσω το λόγο να μα παρουσιάσετε την κατάσταση. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Δύο συμβαστικέ τροπολογίε τελικά έχουμε τώρα, τι οποίε θα ήθελα να σα παρουσιάσω. Όπω είπατε πολύ σωστά, πρόκειται για μία έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία προσπαθεί να συνδυάσει πολλές οδηγίες για την προστασία από την έκθεση σε ιονίζουσες ακτινοβολίες. Εν γέννη υποστηρίζω την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρόκειται για μια έκθεση όπου έχουμε συναρμοδιότητα, κοινή αρμοδιότητα με την Επιτροπή Περιβάλλοντος και αυτό το οποίο συνέβη τελικά είναι ότι οι τροπολογίες αναφέρονται σε πολλά διαφορετικά άρθρα και γι' αυτό το λόγο ήταν πολύ δύσκολο να καταλήξουμε σε συμβαστικές τροπολογίες. Καταρχάς πάντως θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους, τους κοιόδης εισηγητές, με συγχωρείτε, για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε και θεωρώ ότι έχουμε φτάσει πλέον πολύ κοντά σε ένα σημείο συμφωνίας. Καταρχάς θα ήθελα να σας πω ότι υπάρχουν ορισμένες τροπολογίες τις οποίες θεωρήσαμε μη αποδεκτές και αυτό γιατί καλύπτουν κάποια τμήματα της έκθεσης επί των οποίων εμείς δεν έχουμε ούτε αποκλειστική ούτε κοινή αρμοδιότητα. Επομένως τροπολογίες 15, 18, 46 και 51 θεωρούνται ως μη αποδεκτές. Και υπάρχουν ε, δύο τομείς οι οποίοι είναι διαφιλονικούμενοι. Η πρώτη έχει να κάνει με τους ανθρώπους οι οποίοι ταξιδεύουν συχνά με αεροπλάνο, όπου οι σοσιαλιστές ήθελαν να συμπεριληφθεί η κατηγορία αυτή στην έκθεση, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ήταν υπέρ. Εγώ δεν μπορούσα να υποστηρίξω την ε, ιδέα αυτή. Και θεώρησα ότι και τα περισσότερα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενδεχομένως να ανησυχούσαν πλέον ιδιαίτερα για τις ε, συχνές αυτές πτήσεις οι οποίες αναγκάζονται να πάρουν για να συμμετέχουν σε συνεδριάσεις, είπαμε ότι θα μπορούσαμε να είχαμε χωριστή ψηφοφορία προκειμένου όσοι υποστηρίζουν την τροπολογία αυτή για τους ε, συχνά επιβαίνοντες αεροπλάνα να μπορούν να στηρίξουν αυτή την τροπολογία εφόσον το επιθυμούν. Αυτό λοιπόν θα το αποφασίσουμε αύριο και οι σελιστές θα ήθελαν να υποβάλουν μια προφορική τροπολογία προκειμένου να γίνει μια εκ νέου αναφορά στους συχνά επιβαίνοντες αεροπλάνα. Εγώ δεν θα υποστήριζα μια τέτοια προφορική τροπολογία, πάντως στο πνεύμα της καλής συνεργασίας δεν πρόκειται να εμποδίσω τους αλιστές στην προσπάθειά τους να υποβάλουν αυτή την προφορική τροπολογία. Ένας άλλος τομέας, στον οποίο συζητήσαμε ε, εκτενέστατα, είναι οι ανώτατε οριακέ τιμέ έκθεση στην ιονίζουσα ακτινοβολία. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτέ οι οριακέ τιμέ να βασίζονται σε επιστημονικά δεδομένα. Τα επιστημονικά δεδομένα τα οποία έχω δει εγώ, και μάλιστα πρέπει να σα πω ότι μετά από τα δεδομένα αυτά αφαίρεσα δύο δικέ μου τροπολογίε όσον αφορά τι οριακέ τιμέ, πράγμα το οποίο μα αφήνει τελικά με κάποιε τροπολογίε του κυρίου Όρη. Μία εκ των οποίων θα μπορούσα να υποστηρίξω, γιατί υπάρχει αιτιολόγηση για αυτήν αλλά οι τροπολογίες 23, 24 και 38 προσπάθησαν επιτυχώς για τις τροπολογίες αυτές να βρω μια αιτιολόγηση και ενδεχομένως να επιθυμούσε ο κύριο Όρη να μα δώσει μια αιτιολόγηση για αυτέ τι τροπολογίε, ενδεχομένω να θέλει να τη σχολιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πάντω, εγώ ήρθα σε επαφή με εμπειρογνώμονε, οι οποίοι μου είπαν το ότι να μειωθούν τα ανώτατα αυτά όρια ουσιαστικά αντιβαίνει σε όλε τι διεθνέ συμφωνίε τι φυστάμενες και δεν θα μπορούσε επίση να γίνει αποδεκτό αυτό ούτε από την Διεθνή Επιτροπή Εκτινοπροστασία. Έχουμε λοιπόν δύο συμβαστικέ τροπολογίε. Η μία έχει να κάνει με τι τροπολογίε του κυρίου Μπένιεν και νομίζω ότι όλοι οι Όλε οι πολιτικέ ομάδε μπορούν να υποστηρίξουν αυτή την πρώτη συμβαστική τροπολογία και έχουμε συντάξει και μια δεύτερη συμβαστική τροπολογία προκειμένου να καλυφθούν οι τροπολογίε του κυρίου Όρη. Και ουσιαστικά εδώ πέρα λέμε ότι κάθε φορά που ένας εργαζόμενος πρέπει να περάσει από ιατρικές εξετάσεις, τότε αυτό θα πρέπει να γίνεται κατά τη διάρκεια του χρόνου εργασίας και όχι εις βάρος του υπόλοιπου χρόνου, του προσωπικού χρόνου του εργαζόμενου αυτού και όχι με δικό του κόστος. Είπαμε λοιπόν ότι η τροπολογία αυτή 34 θα πρέπει να αναφέρεται στο άρθρο 44, ενώ αρχικά αναφερόταν σε κάποιο άλλο άρθρο του κειμένου. Και επ' αυτής όμως τροπολογίας υπάρχει συμφωνία. Κυρία Πρόεδρε, είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη από την κατάσταση στην οποία έχουμε καταλήξει και είμαι στη διάθεσή σας για περαιτέρω σχόλια. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Πραγματικά ανησυχήτρια την πολύ καλή τη συνεργασία και στη συνεδρίαση των σχεδόν εισηγητών και συμφωνήσαμε γενικά επάνω στα βασικά προβλήματα. Όπως ανέφερε η Άνθια, εκεί που δεν συμφωνούμε είναι να περιληφθούν τα άτομα που ταξιδεύουν συχνά. Νομίζω ότι ήταν καλή ιδέα το γεγονός ότι εισήχθη η διαδικασία της ξεχωριστής ψηφοφορίας και υποστηρίζω αυτή την ιδέα της ξεχωριστής ψηφοφορίας και θα πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί εκεί η ψηφοφορία. Είμαι ευγνώμων στους συναδέλφους που ε, συμφώνησα με τη συμβαστική πρόταση ε, της τροπολογίας 29 όσον αφορά τις διαδικασίες ε, αδειοδιώτησης. Για να μην επαναλαμβάνονται οι διαδικασίες, ώστε κάθε φορά που κάνουν κάτι να χρειάζεται ξεχωριστή άδεια. Και αυτό μπορεί να συμβαίνει πάρα πολλές φορές την ημέρα. Ενώ όταν δίνεται μια γενική άδεια δεν επαναλαμβάνεται διαδικασία διαδότησης. Εδώ χρειάστηκε ένα συμβιβασμό. Επειδή υπάρχουν γλωσσικά προβλήματα όταν υπάρχουν πολλές μεταφράσεις και το θέμα ήταν τεχνικό, τελικά ήταν γλωσσικό το πρόβλημα για να βρεθεί η σωστή διατύπωση. Όσον αφορά την ομάδα μας, δεν συμφωνούμε με την ιδέα να επικταθεί αυτό το θέμα και να περιληφθούν οι συχνοί ταξιδιώτες. Αλλά βεβαίω δεν ξέρουμε αν ε, αυτοί, πρέπει να έχουμε υπόψη μας μπορεί να αντιμετωπίσουν κάποιο κίνδυνο. Ευχαριστώ και πάλι του σκιώδη συζητητέ για τον επικοδομητικό διάλογο που είχαμε μαζί. Ρούς και μετά η Επιτροπή. Γιούτα ευχαριστώ. Ευχαριστώ θερμά τον εισηγητή και Ελπίζω να συντάσσουμε πολύ περισσότερες συμβαστικές τροπολογίες και να περιλάβουμε και τους εκπροσώπους των εργαζομένων στη διαδικασία λήψη αποφάσεων. Γιατί έτσι θα καλύπταμε και τους εργαζόμενους, ασκούμενους, θελοντές και ούτω καθεξής. Ούτε το δικαίωμα σε αδειοδότηση θα πρέπει να αποδυναμώνεται. Ελπίζω κυρία Μακεντάρη, η συγγήτρια, να λάβει υπόψη στις τροπολογίες της με μικρές αλλαγές και το όριο της δόσης. Χρήσιμο θα ήταν και αυτό. Και όσοι ταξιδεύουν συχνά, θα πρέπει αν μη τι άλλο να ενημερώνονται ε, για τους κινδύνους, ε, τους πιθανούς κινδύνους στην υγεία τους από τα συχνά ταξίδια. Είναι χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες και δεν είναι πια και τόσο δαπανηρές. Ομολογώ ότι πριν ασχοληθώ με την έκθεση δεν είχα ιδέα για τα θέματα αυτά. Και όταν κανείς είναι ενημερωμένος, κατατοπισμένος για τις ε, ε, ε, επιδράσεις που έχει στην υγεία του μια συμπεριφορά ή μια ουσία, μπορεί να λάβει τα μέτρα του. Οπότε είναι ευπρόσδεκτη η παροχή πληροφοριών, ιδιαίτερα σε όσους είναι αναγκασμένοι να ταξιδέψουν συχνά για επαγγελματικού λόγους. Και φυσικά καλύπτει κάτι τέτοιο και το προσωπικό των αεροπορικών εταιριών. Οπότε στο άρθρο 16 θα καταθέσουμε αύριο μια προφορική τροπολογία. Και θα ήθελα να παρακαλέσω τους συναδέλφους να σκεφτούν αν πραγματικά ενδιαφέρονται σοβαρά για τα επίπεδα προστασίας. Η τελική ψηφοφορία φυσικά και η θέση μας ως προς την έκθεση θα εξαρτηθεί από την έκβαση σε μεμονωμένα στοιχεία, γιατί μας ενδιαφέρει να συμπεριλάβουμε συγκεκριμένα σημεία για να προστατεύσουμε όσοι έρχονται σε επαφή με ιονίζουσα ακτινοβολία. Ευχαριστώ Τσάμπα Ορί. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα είμαι λακωνικός. Η κυρία Μακεντάιρ υπέβαλε προτάσεις που με βρίσκουν σύμφωνο και οι τροπολογίες μου έλευσαν υπόψη συμβαστικές τροπολογίες. Ήταν ε, εξαιρετική η συνεργασία με την συντάκτρια της γνωμοδότησης, την οποία και ευχαριστώ θερμά για το ανοιχτό και συνεργάσιμο πνεύμα της. Σε ό,τι αφορά τους α, ε, συχνούς ταξιδιώτες και την πρόταση των σοσιαλιστών, θεωρώ ότι είναι υπερβολική η απέτησή τους για τη συγκεκριμένη διατύπωση. Γιατί όλοι εδώ έχουμε πείρα με αεροπορικέ εταιρείε γιατί ταξιδεύουμε συχνά και πιστεύω ότι η πείρα μας θα πρέπει να μας οδηγήσει στην κατάθεση ρεαλιστικών και συνετών τροπολογιών. Ευχαριστώ. Θέλει άλλος κανείς το λόγο παρακαλώ. Όχι. Οπότε να δώσω το λόγο στον κύριο Γιάννησεν, τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι και εγώ εξαιρετικά σύντομο γιατί ο συνάδελφος Στέφαν Μάντικελ σχολίασε τι τροπολογίε που εξετάστηκαν στι 20 Φεβρουαρίου. Επιβεβαιώνω ότι η κυρία Μακεντάιρ μα ζήτησε οι, οι οριακές τιμές να, κριθούν, να συμπεριληφθούν από τους διεθνούς κανόνες και προδιαγραφές ε, της ICAB. Αυτό συνήθως κάνουμε άλλωστε. Δεν θα αποκλίνουμε από τα πορίσματα και τις κατευθυντήριες γραμμές της ε, διεθνούς αυτής εταιρείας. Ό,τι αφορά το κόστος και την επίδραση αυτής της ε, πρότασης στις πολιτικές, η ιδέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, με τη νέα οδηγία είναι να προσφέρει μεγαλύτερο περιθώριο λιγμό στα κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά τη... τη ρύθμιση κάποιων πρακτικών, γιατί οι άδειες ε, δίνονται συνολικά και όχι για μεμονωμένες δραστηριότητες. Με την ενισχυμένη ελαστικότητα που προβλέπει η οδηγία επιτρέπει στις ρυθμιστικές αρχές να μειώσουν το κανονιστικό άχθος και όχι να το αυξήσουν. Ελπίζω με την ελάφρυση αυτή που θα έχει αντίκρισμα και στην πραγματικότητα η κατάσταση να βελτιωθεί. Ευχαριστώ κυρία Μακιντάιρ. Θα είμαι πολύ σύντομη, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για την εξαιρετική συνεργασία και την υποστήριξή τους. Θα ήθελα απλώ να διαβεβαιώσω τον κύριο Στάινρουγκ, την κυρία Στάντρουκ, με συγχωρείτε, ότι ο λόγος για τον οποίο δεν υποστηρίζουμε την τροπολογία για την εκπροσώπηση των εργαζομένων είναι γιατί το άρθρο αυτό αναφέρεται στις αρμόδιες αρχές. Και θα ήθελα πάρα πολύ να υποστηρίξουμε την ιδέα των επιστημονικών δεδομένων και την όλη ιδέα ότι υπάρχουν κάποιες εθνικές αρχές οι οποίες λειτουργούν στα πλαίσια της επιτήρησης. Γι' αυτό το λόγο ουσιαστικά δεν υποστήριξα την υποβληθή σε τροπολογία. Και όπου ήταν δυνατό, πραγματικά υποστηρίξαμε άλλες τροπολογίες και κάποιες άλλες ιδέες, πέρα βέβαια από τους συχνά επιβαίνοντες σε αεροπλάνο, που όπως σας εξήγησα υπήρχαν κάποιες διαφωνίες και αποκλήσεις. Ελπίζω πραγματικά ότι θα έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα στην ψηφοφορία αύριο. Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε. Όπως μας είπε η συγγήτρια θα ψηφίσουμε για τη γνωμοδότηση αυτή αύριο. Και η αρμόδια Επιτροπή θα ψηφίσει στις 24 Απριλίου. Περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, εξετάσεις συμβαστικών τροπολογιών όσον αφορά τις 300, 303 τροπολογίες ε, που έχουν κατατεθεί. Ε, παρακαλώ την κυρία Ρούτν, ναι. Ρόιτερ, Κύριε Όμεν θα δώσω τώρα το λόγο στην κύριο Όμεν ρόιτεν για τις συμβαστικές τροπολογίες σχετικά με την έκθεσή της, μια στρατηγική για επαρκής ασφαλής και βιώσιμης συντάξης. Πρόκειται για μια έκθεση με βάση τη λευκή βίβλο της Επιτροπής που δημοσιεύτηκε το Φεβρουάριο 2012, για το οποίο στην Νομισματική και Οικονομική Επιτροπή η συγητής ήταν ο αντιπρόεδρος μας Τόμας Μαν. Κυρία Όμεν Ρότεν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ειλικρινά θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνεργάστηκαν για να προετοιμάσουμε αυτές τις συμβιβαστικέ τροπολογίες. Έγινε, υπήρξε ένα δούνε και λαβίνε. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους από όλες τις ομάδες και τα μέλη της ομάδος μου του ΕΛΚ όπου έχουμε πολλές δυσκολίες μερικές φορές. Αυτό το οποίο σημειώνω είναι το εξής. Θα ήθελα να σας πω ότι τα κεντρικά σημεία παραμένουν επίκαιρα. Αυτό το οποίο θέλουμε είναι να επεξεργαζόμαστε αυτά τα θέματα ενδελεχώς διότι πρέπει να υπάρχει μια οικονομική σχέση ανάμεσα στον ενεργό πληθυσμό και σε εκείνους οι οποίοι δεν εργάζονται πλέον. Πρέπει να υπάρχουν συμπληρωματικές συντάξεις καταρχήν. Αναγνωρίζουμε επίσης ότι καλό θα ήταν στα κράτη-μέλη δεν πρέπει να λησμονούμε την αρχή της στα κράτη-μέλη λοιπόν να δούμε πώς μπορεί να υπάρχει σωστή κάλυψη για τη μελλοντική συνταξιδότηση των ατόμων. Εξασφαλίζοντας αυτά τα άτομα ένα αξιοπρεπές και λογικό επίπεδο ζωής. Είναι εξίσου σημαντικό, πιστεύω, οι επενδύσεις των συνταξιδοτικών ταμείων να καλύπτονται ώστε οι συντάξεις να μην αφορούν μόνο εκείνους που συνταξιδοτούνται, αλλά ένα ευρύτερο χρονικό ορίζοντα. Καταλήξαμε λοιπόν σε αυτούς τους συμβιβασμούς στα πλαίσια του κειμένου που σας έστειλα χθες βράδυ. Ίσως, όπως είπατε κι εσείς, θα πρέπει να γίνουν ορισμένε παρατηρήσεις. Παρακαλώ λοιπόν τους χιώδης συγητές να το δουν με μεγάλη προσοχή. Όσον αφορά τη συμβαστική ε, πρόταση Β. Εδώ ε, δεν είμαστε αρκετά συνεκτικοί. Αναφερόμαστε, ε, πρέπει να εξασφαλίσουμε μία ένα επίπεδο ζωής επαρκές για όλους. Επίσης, αναφέρθηκε το εξής. Το να κινητοποιηθεί η αγορά εργασίας και να ευαισθητοποιηθεί η αγορά εργασίας, η οποία ενοχλείται από σμένα θέματα. θα πρέπει να αντιμετωπιστούν τα εμπόδια ε, ε, που προβάλλονται στην ενιαία αγορά. Αν το αφήσουμε έχει, αυτό σημαίνει ότι το σχέδιο οδηγίας, αν περιοριστούμε μόνο στην ενιαία αγορά, αναφερόμαστε στο άρθρο 115, πράγμα το οποίο θέλουμε να αποφύγουμε. Λοιπόν, ε, τα εμπόδια στην λειτουργία της ελεύθερης διακίνησης. Αν το αναφέρουμε αυτό θα χρειαστεί ειδική πλειοψηφία στο Συμβούλιο. Συνεπώς πρέπει να γίνει μια προσαρμογή στο κείμενο. Πιο πέρα, συμφωνώ με τους συμβιβασμούς στους οποίους καταλήψαμε και υπήρξε ένα ομαδικό πνεύμα που χαρακτηρίζει τις εργασίες μας Επίσης αναφέρουμε ότι πρέπει να είναι δυνατόν να εργάζεται κανείς περισσότερο και μάλιστα μετά την ηλικία συνταξιδότησης. Η... Τα καθεστώτα πρόορης συνταξιδότησης δεν είναι τα ιδανικά, αλλά πρέπει ο πληθυσμό να γυράσκει, αλλά η υγεία του να είναι καλή. Οι προσδοκίε συνταξιδότηση πρέπει να εξεταστούν με γνώμονα το προσδόκιμο ζωή, αλλά πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και η ισότητα μεταξύ φίλων. Αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο για την ομάδα μας. Επίσης υπάρχουν και άλλα τρία σημαντικά θέματα στη Λευκή Βίβλο. Το σκέλος της συνταξιοδότησης δεν νομίζω ότι μπορεί να ρυθμιστεί εδώ μόνον. Τέθηκε ένα ερώτημα σχετικά με τα ταμεία ερευνών. Δεν πρέπει όμως να αναφερόμαστε μόνο στους ερευνητές. Όταν θέλουμε κινητικότητα, η επιθυμία μας είναι ε, να προστατεύουμε τα συνδοσιακά δικαιώματα και τη μείωση των resting periods. Ευχαριστώ. Φρεντερικ και ο κύριος Μπενιόν στη συνέχεια. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρίες ηγήτρια, κυρίες και κύριοι, καταρχάς θα ήθελα να επιβεβαιώσω τα όσα είπε η συγγήτρια Δηλαδή, το ότι προσπαθήσαμε μέσω των επαφών που είχαμε να καταλήξουμε σε κάποιες συμβαστικές λύσεις. Και είναι σαφές βέβαια ότι εξορισμού ένα συμβασμός συνεπάγεται ένα δούνε και λαβήν και βέβαια πρέπει να γίνουν και κάποιες εκχωρήσεις και υποχωρήσεις. Να ευχαριστήσω πάντως την εισηγήτρια η οποία Μα επέτρεψε να εκφράσουμε τη δική μας την προσέγγιση, μερικές φορές διαφορετική από τη δική της. Θα ήθελα ωστόσο να υπογραμμίσω κάποια στοιχεία τα οποία θεωρώ ότι είναι σημαντικά στα πλαίσια του συμβασμού αυτού. Καταρχώς, ο πρώτος πυλώνας δεν μπορεί να φέρεται μόνο στην ε, ελάχιστη σύνταξη. Θεωρούμε εδώ πέρα ότι θα πρέπει να έχουμε και κάποιες διατάξεις για μια καλή σύνταξη, για μια καλή διαβίωση, και θα πρέπει αυτό να γίνει και σε σχέση με το δεύτερο πυλώνα. Όσον αφορά τώρα τον δεύτερο πυλώνα, καταφέραμε μέσω των συζητήσεών μας να πούμε τελικά ότι δεν ήταν υποχρεωτικό να γίνεται εκεί πέρα μια αναφορά όσον αφορά τον τρίτο πυλώνα. Θα μπορούσαμε να δώσουμε εδώ πέρα κάποια κίνητρα, κυρίως όμως όσον αφορά τα χαμηλά εισοδήματα, κυρίως αυτούς οι οποίοι δεν έχουν καταβάλει συνταξιδοτικές εισφορές επαρκής για μια πλήρη σύνταξη. Τώρα, όσον αφορά το προσδόκιμο ζωής, το οποίο αυξάνεται όλο και περισσότερο, το εξτάσαμε αυτό σε σχέση με το περίφημο ζήτημα της ηλικία συνταξιοδότησης και θεωρούμε ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας την εξέλιξη, τη δημογραφική, χωρίς όμως αυτό αυτόματα να πειράζει και την ηλικία συνταξιοδότησης. Θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας και κάποιες οικονομικές παραμέτρους, και ενδεχομένω και κάποιε άλλε προποθέσει και θα πρέπει να δούμε και τη διατύπωση στο σημείο αυτό έτσι ώστε να μετριάσουμε κατά κάποιο τρόπο την αρχική πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία προέβλεπε μια άμεση σύνδεση τελικά ανάμεσα στο προσδόκιμο ζωής και την ηλικία εξοδότηση. Αυτά ουσιαστικά προσπαθήσαμε να περάσουμε μέσω των τροπολογιών. Αναφερθήκαμε επίση στην αρχή τη επικουρικότητα, η οποία αναφέρεται σε κάποια σημεία του κειμένου, και αυτό είναι ένα σημαντικό σημείο. Έπειτα, όσον αφορά την εργασία μετά τη σταξιοδότηση, εφόσον μπορεί κανεί να συνεχίσει να εργάζεται και εφόσον το επιθυμεί, θα πρέπει να προβλέπεται κάτι τέτοιο και γίνανε και κάποιε συζητήσει όσον αφορά το εκτιμώντα Α, αιτιολογική σκέψη Α, όπου αναφερόταν σε κάποια πράγματα τα οποία είχαμε εξετάσει στα πλαίσια τη πράσινη βίβλου. Θα ήθελα εκεί πέρα να γίνεται μία απλή μόνο αναφορά, χωρίς να ξεκινήσει μία ολόκληρη πάλι συζήτηση, χωρί να ξεκινήσουμε, ε, να ανοίξουμε πάλι, συγγνώμη, τη συζήτηση για, τα, για το πώ μπορούμε να προσεγγίσουμε την ε, πράσινη βίβλο και για το περιεχόμενό τη. Μπορώ να πω εν γέννη ότι είμαι ικανοποιημένο από τι συμβαστικέ λήξει τι οποίε ε, καταλήξαμε. Το ζήτημα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο. Ξέρετε ότι έχουμε ένα κατάλογο ψηφοφορία ιδιαίτερα πολύπλοκο στον οποίο προβλέπονται τροπολογίες που καλύπτονται από τη μία ή την άλλη συμβαστική λύση. Πρέπει ακόμα στο εσωτερικό των πολιτικών ομάδων να γίνουν κάποιες περαιτέρω διεργασίες. Θεωρώ πάντως ότι η άποψή μας αντικατοπτρίζεται συμβαστικές λύσεις οι οποίες καταλήξαμε. Ο κύριος Μπενιόν και ο Τόμας Μάν στη συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Φίλιπ Ντεμπάκερ ουσιαστικά θα έπαιρνε το λόγο, αλλά είναι σε μια άλλη συνεδρία επομένω πρέπει απλώ να διαβάσω το σημείωμα το οποίο μου έδωσε. Ουσιαστικά έχει δύο παρατηρήσει. Όσον αφορά την συμβαστική Τζέι φοβάται ότι η τελευταία πρόταση της συμβαστικής αυτής λύσης ενδεχομένως να δίνει την εντύπωση ότι θέλουμε να ενδυναμώσουμε κάποια συστήματα συνταξιοδότησης, πρόορης συνταξιοδότησης, ενώ δεν θα ήθελε ουσιαστικά να λέγεται κάτι τέτοιο, θέλει ουσιαστικά να αλλάξει κάπως η πρόταση εδώ πέρα και να λέγεται ότι θα πρέπει να υπάρχουν ελκυστικά μοντέλα για ομαλή μετάβαση από την εργασία στη συνταξιοδότηση. Να μην δίνεται δηλαδή εντύπωση ότι προωθούμε εδώ πέρα πρόωρα, προγράμματα πρόορη ταξιοδότηση. Όσον αφορά τη συμβαστική Ή, e, πάλι για την τελευταία πρόταση έχει να κάνει μια παρατήρηση. Εδώ πέρα καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην ταχθεί κατά των επενδύσεων που μπορεί να έχουν γίνει στα ταμεία αποταμίευση για τη σύνταξη. Θα ήθελα εδώ πέρα να λέγεται εν γέννη να μην ε, θέσουμε κινδύνο όλες τις επενδύσεις μπορούν να γίνουν στα πλαίσια συνταξιοδοτικών προγραμμάτων. Επομένως, να μην ε, αναφερόμαστε μόνο στα συνταξιοδοτικά ταμεία, στα λεγόμενα pension funds, αλλά γενικότερα στα επενδυτικά προγράμματα, τα συνταξιοδοτικά. Ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία όσον αφορά τι ε, συμβαστικέ αυτέ λύσει και προσβλέπει ε, σε μια θετική εξέλιξη σήμερα το απόγευμα. Ευχαριστώ. Ο Μαν που είναι και ο συντάκτης γνωμοδότησης της ΕΚΟΝ και μετά η Γιούτα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ θερμά και την Ρία Όμεν. Η Ρία είναι από τους συναδέλφους που πραγματικά παλεύουν λιονταρίσια και πολύ αποτελεσματικά. Το θέμα αυτό μας απασχολεί εδώ και πολλά χρόνια. Έχουν γίνει πολλά, ιδιαίτερα για το θέμα της μεταβίβασης ε, του των δικαιωμάτων αυτών και όπως ακούσαμε αρχικά υπήρχε μεγάλη διάσταση απόψεων αλλά τελικά καταλήξαμε σε πολύ αξιόλογες συμβαστικέ τροπολογίες και νομίζω ότι είμαστε σε θέση να καταφέρουμε κάτι. Εγώ συνέταξα τη γνωμοδότηση για την Επιτροπή ΕΚΟΝ. Εκεί υπάρχουν μερικές μικροεπικαλύψεις και μερικές διαφορές αλλά πιστεύω ότι χάρη στη συνεργασία μας καταφέραμε να εξομαλύνουμε τις διαφορές. Μόνο μία αρνητική ψήφο είχαμε στη γνωμοδότηση και αυτό είναι πραγματικά μεγάλο επίτευγμα. Βέβαια τα θέματα αυτά δεν είναι και πολύ συναρπαστικά για τους δημοσιογράφους που θέλουν πραγματικά λησαλέα μάχη. Αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε πια δικαιολόγηση για τους πυλώνες 2 και 3 και κάποια κράτη-μέλη αποστασιοποιήθηκαν από αυτό. Κρίμα. Αλλά αυτό που κάνουν ορισμένα κρατημέρια για τον πρώτο πυλώνα θα πρέπει να παραμείνει ως θεμελιώδη στοιχείο. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι μια αξιοπρεπής διαβίωση, ένα αξιοπρεπές βιωτικό επίπεδο για όσους δικαιούνται σύνταξη και να έχουμε πραγματικά αξιοπρεπείς συντάξεις. Αυτό που μου άρεσε στις συμβαστικές τροπολογίες είναι ότι περιλαμβάνει και την επικουρικότητα, περιλαμβάνουν και την επικουρικότητα. Τα συστήματά μας λειτουργούν πια και δεν θέλουμε να τα αποδυναμώσουμε. Να μπορούν να είναι βιωσιμότητα, να μπορούν να έχουν βιωσιμότητα, να μπορούν να παρέχουν συντάξεις. Σε αυτό το θέμα είμαστε ιδιαίτερα προσιλωμένοι. Επίσης το θέμα της πρόρης συνταξιοδότησης είναι ένα θέμα που προκαλεί μερικές φορές φοδρές συζητήσεις. πολλοί αναγκάστηκαν κατά κάποιο τρόπο σε πρόορη δεξιοδότηση και τελικά είδαν ότι είναι αρνητικό κάτι τέτοιο. Δεν θα πρέπει ε, όσοι είναι ικανοί και επιθυμούν να συνεχίσουν την εργασία τους να αποτρέπονται από κάτι τέτοιο επειδή ήρθε το όριο της συνταξιοδότησης. Θα πρέπει να υπάρχει τέτοια δυνατότητα και τέτοια ελαστικότητα. Και χαίρομαι που τελικά καταλήξαμε στη συμφωνία. Νομίζω ότι το τελικό αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων είναι πολύ θετικό όρια. Ας μην ξεχνούμε ότι πρόκειται για έκθεση ίδια πρωτοβουλία. Πολλοί βέβαια δημοσιογράφοι θα πούν «Ε, και τι αξία έχει μια έκθεση ίδιας πρωτοβουλία. Λάθος όμως, γιατί τέτοιου είδους πρωτοβουλίες ε, και τέτοιου είδους εκθέσεις όπως αυτή στέλνουν χειρά μηνύματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι οι λεπτομέρειες είναι πολύ σημαντικές ε, και η συγκεκριμένη έκθεση της πρωτοβουλίας είναι επίση σημαντική και ελπίζω να αναγνωριστεί η αξία της. Είχαμε πραγματικά και ένα πολύ καλό παράδειγμα προς μίμηση ως προς την αγαστή συνεργασία. Χαίρομαι ε, για τη συνεργασία αυτή και ελπίζω ότι θα έχει αντίκρισμα και στην αυριανή ψηφοφορία. Η Γιούτα Στάινρουκ και μετά ο κύριος Μπέκερ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Συμφωνώ ως προς τα ουσιώδη με τους προλαλήσαντες. Θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο σημεία. Για μας, ε, τους ε, Γερμανούς Σοσιαλδημοκράτες, είναι σημαντικό το όριο συνταξιοδότησης να μην προσδιορίζεται με βάση το προσδόκιμο ζωής, αλλά να προσδιορίζεται με βάση το, τα έτη εργασίας και να μην παρατηρηθούν τα κρατημέλη να τροποποιήσουν τα αξιοδοτικά του συστήματα. Βέβαια μια αναθεώρηση χρειάζεται, αλλά οι επισφαλείς μορφές απασχόληση είναι αυτές που ε, οδηγούν στη φτώχεια τους πιο ηλικιωμένους ε, και τις γυναίκες σε περίπτωση που χρειάστηκε να διακόψουν την εργασία τους ε, για μερικά έτη και να ασχοληθούν με την οικογένειά τους. Και το θέμα της ανεργίας είναι πολύ σημαντικό. Θα πρέπει το θέμα αυτό και τις προσπάθειες εκρίζωσης της φτώχειας να καλυφθούν και οι αξιοπρεπείς μισθοί όπως ε, και οι αξιοπρεπείς συμβάσει. Για τι συμβαστικέ τροπολογίες β και τώρα. Και ε, για την τροπολογία μου 170. Η τροπολογία 170 μιλά για την ε, ειδική προστασία α, για κάποιων συνταξιοδοτικών συστημάτων επιχειρήσεων. Η εισηγήτρια μας είπε ότι η τροπολογία αυτή 270 καλύπτεται από τη συμβαστική τροπολογία νη. Αλλά διαφορά, Γιατί αναφέρεται μόνο στην επικουρικότητα. Αλλά δεν προβλέπει ρητά την προστασία των επιχειρηματικών συντάξεων. Και αυτό το ζήτημα δεν απασχολεί μόνο τη Γερμανία, αλλά και άλλα κρατημέλη. Οι συντάξει των επιχειρήσεων είναι σημαντικές για να αποτραπεί η για τις φτώχειας, ιδιαίτερα για τους ηλικιωμένους. Και αν ε, προβλεφθούν κάποιες αλλαγές σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ε, καταργηθούν αυτές οι επιχειρηματικές συντάξεις, οι συντάξεις που δίνονται από τις επιχειρήσεις, θα έχουν τεράστιο κοινωνικό αντίκτυπο, πολύ αρνητικό, σε όλα τα κράτη-μέλη. Και θα πρέπει τα κράτη-μέλη να καλύψουν το κενό που δημιουργείται από την κατάργηση τέτοιων ε, συνταξιδοτικών συστημάτων που παρέχονται από επιχειρήσεις. Ελπίζω να το λάβουμε αυτό υπόψη, γιατί εμείς ε, ως ε, νομοθέτες που διαμορφώνουν πολιτικές δεν θα πρέπει να καταστρέφουμε ε, εύρυθμα και σωστά λειτουργούντα συστήματα. Θα πρέπει αυτό να το δηλώσουμε ρητά. Κυρία, ο κύριος Μπέκερ και μετά η κυρία Γκουτιέρες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα, θα, Θέλω να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τον εισηγητή. Τώρα θέλω να κάνω ορισμένες προκαταρκτικές παρατηρήσεις. Ορισμένα στοιχεία δεν με ικανοποιούν. Κάποιος από την ομάδα μου θα διατυπώσει τη σκέψη, αλλά δεν με ικανοποιούν ορισμένα σημεία. επομισθήκαμε πολύ μεγάλο βάρος για να προσανατολίσουμε τα κοινωνικά βάρη του μέλλοντος. Αυτή η ευθύνη είναι πολύ σημαντική και ο προσανατολισμός μας θα είναι σημαντικός και για τα μέσα ενημέρωσης. Η θέση μας πρέπει να είναι σαφής για τις επόμενες γενναίες, τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Όχι για όσους έχουν ήδη συνταξιδοτηθεί, αλλά για το μέλλον. Σε όλα αυτά λοιπόν προστίθεται το γεγονός ότι σε ορισμένα κράτη-μέλη, κυρίως του Νότου της Ευρώπης, πρέπει να ενισχυθεί η κατάσταση, επειδή τα συστήματα αυτά δεν είναι επαρκώς ανεπτυγμένα. Και εμείς είμαστε σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνοι Δεν θα πρέπει όλα αυτά να αξιολογηθούν με βάση την σημερινή χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση. Πρέπει να αναγνωρίσουμε το γεγονός ότι θα πρέπει να προβλεφθεί ένα ελάχιστο ποσό για να επιβιώσει κανείς και ίσως δραστηριότητα για τα άτομα μεγαλύτερης ηλικία, ώστε να εξασφαλίζεται ένα καλό επίπεδο ζωής και καλή ποιότητα ζωής. Να υπάρχει αξιοπρέπεια για τα χρόνια της σύνταξης. Ευχαριστώ πολύ για τους, τις συμβαστικές λύσεις τις οποίες ε, καταλήξατε όπου βλέπω και δικές μου τοποθετήσεις ε, το επαναλαμβάνω πιστεύω ότι πρέπει να υπογραμμίσουμε περισσότερο την συμμετοχή των μελλοντικών και των προηγουμένων γενεών, ώστε να υπάρχει μια κοινή λύση, να μην υπάρχει σύγκρουση γενεών. Και θα ήθελα να σας ζητήσω να δείξετε κατανόηση, επειδή υπάρχουν χώρες όπου και στις σκανδιναβικές χώρες, για παράδειγμα, μπορεί κανείς να εργάζεται ελεύθερα μετά τη συντεξιδότηση όχι μόνο υπάρχει μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής που θα είναι μία από τις παραμέτρους για την ηλικία συνταξιδότησης, αλλά πρέπει να έχουμε κατά νου και άλλα κριτήρια. Για παράδειγμα, τη μετανάστευση, ε, την κατάσταση υγείας του πληθυσμού γενικά. Όλα αυτά είναι σημαντικά κριτήρια θα πρέπει να βασιζόμαστε σε κριτήρια λαϊκιστικά, αλλά σε στοιχεία τα οποία έχουν, είναι τα απορίσματα ερευνών. Θα ήθελα λοιπόν να υπογραμμίσω ότι υπάρχουν πολλά στοιχεία που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Ε, σε μάς. Το πρώτο που πρέπει να επιδιώκουμε είναι συνένεση μεταξύ νέων και μεγαλύτερων ανθρώπων. Πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει συνένεση μεταξύ των γενεών και αυτή θα πρέπει να είναι η περιοτεραιότητά μας. Αυτή είναι η βασική μου θέση και χαίρομαι που αντιμετωπίστηκε τόσο επαγγελματικά αυτό το σημαντικό θέμα και σήμερα το απόγευμα θα απόσχω και ζητώ και πάλι την κατανόησή σας και ευχαριστώ τον εισηγητή που κατάλαβε τη θέση μου. Και πάλι σας ευχαριστώ που μου επιτρέψατε να παραθέσω τις απόψεις μου. Ο Σέρχιο Γκουτιέρες παρακαλώ. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ και την εισηγήτρια και τους και οδησηγητές που ασχολήθηκαν με την έκθεση αυτή που είναι πολύ καλή και πολύ σωστό σημείο φετηρίας για να δώσουμε ένα ηχηρό μήνυμα για το είδος των συντάξεων και το μοντέλο των συντάξεων που επιθυμούμε. Αλλά ένα παράπονο θα ήθελα να εκφράσω. Όντως θέλουμε να εμπλουτίσουμε τη Λευκή Βίβλο με τη δική μας θέση για τα συνταξιοδοτικά συστήματα και είπαμε να συντάξουμε κάποιες γενικές αρχές, κατευθυντήριες γραμμές για τα ισχυρά συνταξιοδοτικά συστήματα της Ευρώπης. Από πρώτος πυλώνες θα αφορά την εξασφάλιση ενός ελάχιστου εισοδήματος ε, στους ηλικιωμένους, άνω, άνω των 65 των ε, του συνταξιούχους και δεύτερο και τρίτο πυλώνα που με διαφάνεια θα περιλαμβάνουν ε, μεγαλύτερα, ευρύτερα περιθώρια λιγμών αυτονομίας και προσωπικής ευθύνης για τις μελλοντικές συντάξεις. Και το παράπονο μου είναι ότι φαίνεται ότι μερικές φορές το έργο μας δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, γιατί η πραγματικότητα λέει ότι αυτές οι γενικές αρχές ουσιαστικά είναι παράλληλες με τη... τις εντολές Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τα κράτη-μέλη για τα εθνικά ε, προγράμματα μεταρρυθμίσεων και το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποβάλλουμε κάποιες κατευθυντήριες γραμμές για τα μελλοντικά συνταξιοδοτικά συστήματα, αλλά τα κράτη-μέλη αναθεωρούν τα συνταξιοδοτικά του συστήματα με τρόπο που αντιβαίνει πλήρως ε, στις δικές μας απόψεις και κατευθυντήριες γραμμές. Και πιστεύω ότι θα πρέπει να εκφράσουμε τη λύπη μας για αυτή την ε, απόσταση που υπάρχει. Θα ήθελα τώρα να επικεντρωθώ σε τρεις-τέσσερις βασικές κατευθυντήριες γραμμές της έκθεσης. Την πρώτη την ανέφερε και η συνάδελφος Γιούταρα Στάινμπρουκ. Πολλά κρατημέλη προσπαθούν αυτόματα να συνδέσουν το προσδόκιμο ηλικία, το προσδόκιμο ζωής μάλλον, με το όριο συνταξιοδότησης. Αυτό είναι λάθος και οδηγεί σε μεγαλύτερη αποδυνάμωση των συντάξεων, σε φτώχιση των συντάξεων και τη μη προσαρμογή των συντάξεων στο κόστος ζωής. Δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι η βιωσιμότητα των ε, δημοσίων συνταξιδοτικών συστημάτων ε, εξαρτάται από τα επίπεδα απασχόλησης, από την ποιότητα απασχόλησης και από, το, από την ηλικία ένταξης στην αγορά εργασίας. Δεν θα πρέπει να είμαστε εναλλαστικοί όλες οι αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που κάνουν τα κρατημέλη θα πρέπει να είναι ελαστικές και να προβλέπουν μεγάλες περιόδους προσαρμογής. Ιδιαίτερα στους περιόδους υπολογισμού και στις αδιαδρομίες θα πρέπει να έχουμε μεγάλη ελαστικότητα για να μην οδηγηθούμε de facto σε μια αποδυνάμωση των συνταξιδοτικών μας συστημάτων και μια πίσχνασή τους. Γιατί αυτό θα πλήξει στο μέλλον εκατομμύρια συμπολίτε μας. Οι αλλαγές που θα γίνουν θα πρέπει να είναι ελαστικές και με μακροχρόνιες περιόδους προσαρμογής, ώστε να μπορέσουν οι εργαζόμενοι να προσαρμοστούν στους νέους κανόνες. Και η παρούσα οικονομική κρίση μας έκανε να βιώσουμε σε πολλά κρατημέλη ότι οι συντάξεις δεν είναι απλώς πυλώνας του κράτους πρόνοιας, αλλά σε χαλεπούς οικονομικούς και κοινωνικούς καιρούς έχουν, έχουν μετατραπεί σε ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας στη χώρα, γιατί έχουμε πολλές οικογένειες ανέργων που στη χώρα μας επιβιώνουν χάρη στα ισχυρά στα συστήματα που έχουμε δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια. Ευχαριστώ. Ε, Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα απλώς να σχολιάσω πολύ σύντομα και να προσθέσω πράγματα που έχω πει και σε προηγούμενες συνεδριάσεις. Θεωρώ ότι η έκθεση αυτή πρωτοβουλία θα μπορούσε να αποτελέσει μια καταπληκτική ευκαιρία προκειμένου να εκφράσουμε κάποιες επικρίσεις. Δυστυχώς όμως αυτό το οποίο βλέπω είναι ότι οι δικές μας τροπολογίες έχουν ε, παρακαμφθεί. Γι' αυτό το λόγο δεν είμαστε ικανοποιημένοι με αυτή την έκθεση. Αυτό που θα έπρεπε να μας απασχολήσει είναι τι θα καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε ως σύνταξη στο μέλλον για τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται εκτός απασχόλησης ή σε επισφαλή θέση απασχόλησης. Πολύ φοβάμαι ότι δεν λέμε τίποτα το νέο. Απλώς ε, αναμασάμε πράγματα που έχουμε ξαναπεί στο παρελθόν όσον αφορά το προσδόκιμο ζωής, όσον αφορά την ηλικία συνταξιοδότησης, Προφανώς οι συντάξεις θα πρέπει να προσαρμοστούν σιγά σιγά σε ένα όλο και αυξανόμενο προσδόκιμο ζωής. Ωστόσο τα δεδομένα αυτά μας ήταν ήδη γνωστά και ξέρετε, το λένε άλλωστε και οι ίδιοι επιστήμονες, ότι η προσέγγιση αυτή από μόνη της είναι λυπής. Ξέρετε ότι αν η αυξανόμενη παραγωγικότητα δεν οδηγεί και σε αυξανόμενα εισοδήματα, δηλαδή αυξανόμενες ασφαλιστικές εισφορές, τότε στο τέλος τελικά θα αντιμετωπίσουμε και πάλι τα προβλήματα του παρελθόντος. Θεωρώ ότι τα όσα λέγονται για την πρώτη, δεύτερη, τρίτη σύνταξη δεν είναι ικανοποιητικά και νομίζω ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε ακόμα περισσότερο στο ζήτημα των δημοσίων συντάξεων, στα δημόσια συστήματα αξιταξιοδότησης τα οποία σε κάθε περίπτωση είναι πιο φτηνά από τα ιδιωτικά συστήματα και πολύ πιο ευάλωτα στις εκάστοτε οικονομικές κρίσεις. Και ξέρετε ότι ακριβώς στον τομέα αυτό είναι που οι στεξιούχοι φοβούνται περισσότερο ότι μπορούν να χάσουν τα δικαιώματά τους. Ελοχεύει όμως και ένας κίνδυνος ακόμα βλέπουμε ότι οι προπολογισμοί δεν είναι σχεδιασμένοι κατά τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτουν δημοσιονομικά ελλείμματα. Δείτε το παράδειγμα τη Ισπανία, για παράδειγμα. Βλέπετε ότι υπάρχουν όλο και περισσότεροι ταξιούχοι οι οποίοι χάνουν τελικά τα εξωτικά του δικαιώματα. Υπάρχουν σημαντικότητε περικοπέ στι συντάξει του, αναγκάζονται πολλοί να εργάζονται για περισσότερα χρόνια Καταλαβαίνετε ότι οι άνθρωποι που έχουν εργαστεί σκληρά για ολόκληρε δεκαετίε δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται με αυτόν τον τρόπο. Είναι, αν μη τι άλλο, απαξιωτικό. Θεωρώ λοιπόν ότι η προσέγγιση τη έκθεση αυτή είναι απογοητευτική και δεν μπορούμε να τη στηρίξουμε. Πρόεδρο, υπάρχουν ε, άλλοι που θέλουν να πάρουν το λόγο. Πρωτού δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν βλέπω κανέναν. Εκ μέρου Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπάρχει κάποιο που θα θέλει να πάρει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν είχα ακόμη την ευκαιρία να διαβάσω ε, την διατύπωση που έχουν ε, οι συμβασμοί και θα, θα κάνω λίγα σχόλια σχετικά με τη συζήτηση που έγινε. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πολύ τα αξιότιμα μέλη ε, που αποδέχτηκαν αυτή την έκθεση και τα βασικά μηνύματα και τους γενικούς μας στόχους σε αυτή τη δημογραφική κατάσταση που είναι να παροτρύνουμε τα άτομα να εργάζονται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Τα άλλα ε, εργαλεία πολιτικής όσον αφορά την ηλικία συνταξιδότησης με βάση την μας ζωής είναι όλα αυτά θέματα και πρέπει να έχουμε εργαλεία για να πραγματοποιήσουμε το στόχο μας. Τώρα, σχετικά με το ρόλο των διαφόρων συνταξιδικών πυλώνων για να υπάρχουν επαρκείς συντάξεις στο μέλλον, η Λευκή Βίβλος και η επάρκεια των συντάξεων ε, και οι, εκθέσεις, οι σχετικές εκθέσεις που ε, δημοσιεύτηκαν από την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων τον Μάιο έχουν καταστήσει σαφές ότι ε, το θέμα της συντάξεως είναι πολύ σημαντικό με βάση τις επαρκείς συντάξεις και φυσικά οι συμπληρωματικές συντάξεις θα παίξουν κάποιο ρόλο. Ο σκοπός της, των πρωτοβουλειών της Επιτροπής ε, στην παρότρινση συμπληρωματικών συντάξεων είναι να βελτιωθούν τα δικαιώματα των ε, συνταξιδοτούμενων χωρίς να επιβαρύνουμε υπερβολικά ε, εκείνους οι οποίοι θα επομισθούν τα βάρη και όλα αυτά έχουν ληφθεί υπόψη. Τέλος, σχετικά με το ερώτημα, σχετικά το συνδεσμευτικό ταμείο των ερευνητών, αυτή δεν είναι μια γενική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά μια πρωτοβουλία που ανέλαβε μια ομάδα μεγάλων πανεπιστημίων και Ινστιτούτων Ερευνών, ε, το Κέμπρος παραδείγμα, το ΣΕΡΝ, διαφόρων κρατών μελών, ιδρυμάτων κρατών μελών, που θα ήθελαν να δημιουργήσουν ένα πανευρωπαϊκό ταμείο σύνταξης για τους ερευνητέ τους. Και δεδομένου ότι θα είναι το πρώτο ταμείο αυτής της μορφής στην Ευρώπη, η Επιτροπή υποστηρίζει αυτή την πρωτοβουλία των πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων, ε, παρέχοντας ε, συμβουλές γνωμοδοτήσεις. Δεν αναφερόμαστε τώρα σε μια ε, νομοθετική πρωτοβουλία που δεσμεύει την Ευρωπαϊκή Ένωση ή που προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Αν δεν υπάρχουν άλλες παρατηρήσεις, θα δώσω πάλι το λόγο στην συγκήτρια. Θα ήθελα... Όσον αφορά το Ταμείο Σταξιδότησης των Ερευνητών, Ξέρετε ότι βάσει τη κοινοτική νομοθεσία είναι δυνατόν να ξεκινήσουμε με την ιδέα αυτή. Για ποιο λόγο θα πρέπει να ληφθεί μια νέα κοινοτική πρωτοβουλία. Είναι ήδη δυνατό να στηθεί το ταμείο αυτό. Αν οι ερευνητέ και επιστήμονε επιθυμούν να καταρτήσουν τέτοιο ταμείο, μπορούν να το κάνουν. Δεν χρειάζεται κοινοτική πρωτοβουλία για κάτι τέτοιο. Ήδη προβλέπεται από την υφιστάμενη νομοθεσία. Θα μιλήσω τώρα Ολλανδικά, κυρία Πρόεδρε. Κύριος Μπέκερ. Πήρε το λόγο και αναφέρθηκε στην πτυχή εκείνη στη σχέση ανάμεσα στις διαφορετικές γενναίες. Δεν αναφέρθηκα σε όλα τα σημεία τα οποία ανέπτυξε, γιατί θεωρώ ότι πέρασε σε τόσες πολλές λεπτομέρειες. Για παράδειγμα, είπε ότι θα πρέπει κάθε τρία χρόνια να γίνονται έλεγχοι και είπε ότι θα πρέπει να εμπλέκονται επιστήμονες, ερευνητές και το καθεξής και ότι θα πρέπει η προσέγγισή μας να είναι σαφώς αμερόληπτη. Πολύ φιλόδοξη και καλή η προσέγγιση αυτή, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να ενταχθεί στην έκθεση αυτή. Θεώρησε ότι οι τροπολογίες ήταν ιδιαίτερα λεπτομερείς. Δεν θα μπορούσαν να ενταχθούν σε μια έκθεση σαν τη δική μου. Πάντως αναφέρθηκα στην διαγενεαλογική πλευρά. Ο κύριος Χάντελ, ο οποίος προέρχεται από τη Γερμανία και καταλαβαίνω πόσο σημαντικός είναι για σας ο πρώτος πυλώνας, κύριε Χάντελ. Και η Γιούτα Στάνμπρουκ επίσης μίλησε για τη σημασία του πυλώνα αυτού. Κύριε Πρόεδρε, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι είναι ακριβώς όμως στη Γερμανία που έχουν γίνει οι πιο βάναυσες μεταρρυθμίσεις. Δεν μπορείτε να το προσάπτετε αυτό στην Ευρώπη. Ξέρετε ότι στα πλαίσια της Γερμανίας τελικά είδαμε στον πρώτο πυλώνα μια σημαντικότατη μείωση της συντάξης. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει ενδεχομένω να δείτε τα πράγματα λίγο διαφορετικά, να επανεξετάσετε τους συμβιβασμούς και να δείτε και την αρχική έκθεση. Ο πρώτος πυλώνας είναι πάρα πολύ σημαντικός. ο κύριος Νταρντέν, η Τζιν Λάμπερτ και άλλοι ασχολήθηκαν με το ζήτημα αυτό και με τη δική μου τη συνεργασία και το, ο στόχος μας είναι να μην εξασφαλίσουμε απλώς ένα αξιοπρεπές εισόδημα, αλλά να μπορεί κανείς να ζει αξιοπρεπώς με το εισόδημα αυτό. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει εκ του σύνεγγις να εξετάσετε το ζήτημα εδώ πέρα. Μην πείτε απλώ όχι με την πρώτη ματιά. Θεωρώ ότι εμεί είναι καλύτερο από αυτό το οποίο ήδη διαθέτεται. Μπορείτε να επικρίνετε την πρόταση, αλλά σα ζητώ να την εξετάσετε καλύτερα, με ένα πιο θετικό πνεύμα. Τώρα πιο συγκεκριμένα, απευθυνόμενη στη Γιούτα. Νομίζω ότι η τροπολογία σου καλύπτεται από τη συμβαστική λύση. Νομίζω ότι πρόκειται για τη συμβαστική J, αν δεν κάνω λάθος, όχι την M, διορθώνει ο Αν διαβάσει την ε, συμβαστική τροπολογία θα δεις ότι εκεί πέρα αναφέρεται το εξής. Όχι, διορθώνει ο μιλήτρια, μάλλον δεν είναι η συμβαστική M. Δεν μπορώ να την εντοπίσω. Η N. N. Λέγεται λοιπόν εκεί ότι οι συνταξιούχοι παραμένουν υπό την αρμοδιότητα των κρατών μελών και φοβόμαστε ότι οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία στον τομέα αυτό μπορεί να επηρεάσει τα στεξωτικά συστήματα τεχνικά των κρατών μελών. Αν αυτό δεν είναι επικουρικότητα, δεν ξέρω τι είναι. Επομένως, Γιούτα θεωρώ ότι καλύπτεται η αρχή της επικουρικότητας στην συμβαστική αυτή πρόταση. Μπορούμε να το ξαναδούμε πάντως, αν το επιθυμείς. Κυρία Πρόεδρε, τώρα σε σχέση με τις ε, παρατηρήσεις οι οποίες άκουσα, όντως έκανε υποχωρήσει σε κάποια σημεία, προσπάθησε να προσαρμόσω τη διατύπωση και αυτό έγινε σκεμμένα, προκειμένου να καταφέρουμε να έχουμε μια ξεκάθαρη γραμμή, μια γραμμή με την οποία όλοι θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε. Τα μέλη δηλαδή τα οποία προέρχονται από διαφορετικές πολιτικές ομάδες στα πλαίσια της Επιτροπής μας. Και από ό,τι βλέπω οι φιλελεύθεροι, ο Φίλιπ Ντεμπάκερ και άλλοι, δεν συμφωνούν με το επενδυτικό δυναμικό των επενδυτών στα πλαίσια των συνταξιδοτικών ταμείων. Δεν θα ήθελα όμως να γίνει εδώ πέρα μια διασύνδεση με το IOP. Γι' αυτό το λόγο χρησιμοποίησα τη διατύπωση την οποία βλέπετε στη συμβαστική λύση. Επίσης, κάποιοι είχαν ένα πρόβλημα με τη διατύπωσή μου όταν λέω ότι θα πρέπει να καταπολεμήσουμε τον αθέμητο ανταγωνισμό. Θα πρέπει να δούμε και ποια είναι η άποψη των υπολείπων συναδέλφων. δεν απαραίτητο να χρησιμοποιήσουμε τον όρο καταπολεμό, καταπολεμό τον αθέμητο ανταγωνισμό, γιατί σε άλλα σημεία έχουμε αναφέρει εκτενέστατα τον αθέμητο ανταγωνισμό. Μπορούμε ενδεχομένω στο σημείο αυτό να το διαγράψουμε κιόλα, αν το επιθυμείτε. Πάντως συμφωνώ μαζί σας για τα όσα υπόθηκαν για το H. Τώρα περνάω στο J. Εδώ γίνεται λόγος για τα συνταξιωτικά κοινά προγράμματα τα οποία μπορούν να βοηθήσουν ορισμένους εργαζομένους να χρησιμοποιήσουν περαιτέρω και μετά τη σύνταξη δηλαδή τα επαγγελματικά προσόντα τα οποία έχουν και ζητάμε από τους κοινωνικούς εταίρους να έχουν ένα συγκεκριμένο μοντέλο για μια ευάλωτη μετα... Ε, συγγνώμη, για μια ευέλικτη μετάβαση από την εργασία στη σταξιοδότηση. Τι θέλουμε να πούμε με τη συμβαστική αυτή λύση. Αν υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει εργαστεί σε όλη τη ζωή του, εφόσον φτάσει, εφόσον φτάσει στα 60, δεν θα πρέπει κανείς να μπορεί να αγγίξει ή να επηρεάσει τη σύνταξή του αυτή. Θα πρέπει να καταφέρει μαζί με τον εργοδότη του, εφόσον επιθυμεί να συνεχίσει να εργάζεται, είτε να εργάζεται λιγότερο, είτε να προσαρμοστούν κατά κάποιον τρόπο οι εργασιακές του συνθήκες. Εδώ πέρα δεν αναφερόμαστε σε πρόριστα αξιοδότηση πάντως, αναφερόμαστε σε μία ελαφριά ευέλικτη τροποποίηση των συνθηκών εργασίας. Πάντως το ζήτημα αυτό το καλύψαμε εκτενέστατα. Κυρία Πρόεδρε, θεωρώ ότι με τον τρόπο αυτό καλύπτω και την παρατήρηση της Γιούτα για τις εργασιακές συνθήκες και την πρόριστα αξιοδότηση. Θεωρώ ότι αυτά είχα να σας πω. Θα μπορούσα να αφαιρθώ και σε, κάποια, σε κάποιες άλλες προσωπικές παρατηρήσεις. Μου υπόθηκε ότι θα πρέπει να κάνω κάποιες διευθετήσεις, προσαρμογές σε κάποια σημεία, για παράδειγμα στην συμβαστική Β, θα πρέπει να λέγεται ότι τουλάχιστον εγγυάται ένα αξιοπρεπές επίπεδο ζωής για όλους. Αυτό θα προσθεθεί σαν φράση στο σημείο αυτό, στην συμβαστική αυτή λύση, προκειμένου να υπάρχει μεγαλύτερη συνεκτικότητα με άλλα σημεία της έκθεσης, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι στο 3α η ο Φρεντερίκ με συγχωρείτε έχει δίκιο για το σημείο αυτό θα πρέπει να αφαιρέσουμε την αναφορά η οποία γίνεται στην ηλικία στεξιοδότηση, καθώς επίσης και τον λόγο αναφοράς για τις στεξιοδοτήσεις. Και αυτό το έχουμε συζητήσει και σε προηγούμενη συνεδρίαση. Τώρα όσον αφορά τα όσα είπε ο τα έχω καλύψει θεωρώ. Συμβαστική τροπολογία Q όσον αφορά τα εμπόδια. Εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία Νομίζω ότι και αυτό θα πρέπει να προσθεθεί ως ιδέα. Αυτές είναι οι παρατηρήσεις που είχα να κάνω, κυρία Πρόεδρε. Θα σας διανύμω τις νέες αυτές τροποποιήσεις. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για την προσοχή σας. Και αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το πολύ θετικό πνεύμα συνεργασίας που είχαμε. Ευχαριστώ. Θα ψηφίσουμε αύριο για την έκθεση κυρίας Ρόιτεν, ώστε να μπορέσουμε να την διαβάσουμε στην Ολομέλεια του Μαΐου. Πέραμε στο σημείο 7 τώρα της ημερήσιας διάταξης, να σας κάνω μια ενημέρωση ε, για τα πορίσματα του πρώτου τριμερίου διαλόγου, που έλαβε χώρα στις 14 Μαρτίου. Θέμα ήταν η διαπραγματεύση με το Συμβούλιο σχετικά με τις αρμοδιότητες του κράτους σημαίας. Μετά την απόφαση των συντονιστών και της ε, Επιτροπής μας, θα θυμάστε ότι επικυρώσαμε την διαπραγματευτική εντολή και με ψηφοφορία στην Ολομέλεια που έγινε στις 13 Μαρτίου και μάλιστα στην ψηφοφορία εγκρίθηκαν 69 τροπολογίες Κάτι που επιβεβαίωσαν και την έκβαση στη ψηφοφορία στην Επιτροπή μας και άλλα στοιχεία συμπλήρωσαν την αρχική διαπραγματευτική εντολή. Η Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων ε, ανέθεσε στην ε, Ιρλανδική Προεδρία την εντολή να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να επισημάνω ότι η εντολή της Ολομέλειας επιβεβαιώθηκε και από μια ενδεικτική ψηφοφορία που επικύρωσε αυτή την εντολή με 498 ψήφους, δηλαδή με 120 ψήφους ε, επιπλέον της απαιτούμενης ενισχυμένης πλειοψηφίας, κάτι που δείχνει τη συντριπτική υποστήριξη, τη συντριπτική πλειοψηφία που υποστήριξε αυτή την εντολή ήταν ε, ο εκπρόσωπο του ΕΛΚΑ, Φιλίπ Δεμπακέν για τους Φιλελεύθερου. Τζιν Λάμπερτ για τους πράσινου, Πατρίκ Λεγιαρή για, τους, για, την Κούε και ε, μεταρρυθμιστές ε, κυρία Μακεντάιρ, ένα για του σοσιαλιστέ. Έχω μια σύγκρουση αρμοδιοτήτων γιατί είμαι και σκιωδησηγητρία και η πρόεδρος της ε, διαπραγματευτικής ομάδας. Ο κύριος Ζερσμπακ που είναι ο αρμόδιος συντάκτης Αγρομοδότη Επιτροπής Μεταφορών, προσθέθηκε σε αυτή τη διαπραγματευτική ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στον πρώτο τριμερή διάλογο, λοιπόν, έγινε μια ανταλλαγή απόψεων για το χρονοδιάγραμμα και κοινοποίησαμε στο Συμβούλιο την επιθυμία μας ε, η συζήτηση για το θέμα αυτό να συνδυαστεί με την συζήτηση για την ευθύνη του κράτους ε, λιμένος για να μην υπάρχουν ε, αντιφάσεις μεταξύ των δύο κειμένων. Επίσης, ε, εκφράσαμε μια γενική μας ανησυχία ως προς το κείμενο της ε, συνθήκης για τη θάλασσα. Και περάσαμε και στο κυρίως θέμα της συζήτησης, τουλάχιστον στο πρώτο σκέλος, το θέμα των αιτιάσεων των παραπώνων που γίνονται στη διάρκεια του πλού. Κάτι που δεν είχε ε, περιλάβει στην αρχική πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ το... οι κοινωνικοί εταίροι το ζήτησαν. Βέβαια, κάλιο πέντε και στο χέρι, παρά δέκα και καρτέρι. Ε, και είπαμε ότι ίσως το κείμενο των κοινωνικών εταίρων δεν θα πρέπει εξαντλητικά να περιλαμβάνεται στο κείμενο και ζητήσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τις αναθέσαμε μάλλον, να υποβάλλει μια διατύπωση που θα περιλαμβάνει ρητή μνήα αυτής της δυνατότητας να υποβληθούν αιτιάσεις και ε, στο, στη διάρκεια του πλού. Ώστε το σύνολο το, της συμφωνίας των κοινωνικών εταίρων να ευθυγραμμίζεται με το κείμενο της σύμβασης, να μην υπάρχουν κάποια κενά ή να μην έχουν παραγωνιστεί κάποια θέματα. Επίσης, ε, ασχοληθήκαμε και με το θέμα της πιστοποίησης. Το θέμα είναι πώς τα κράτη-μέλη ελέγχουν ή δεν ελέγχουν τις επιχειρήσεις πιστοποίησης τις επιχειρήσεις που εκδίδουν πιστοποιητικά. Το θέμα είναι, τα κράτη-μέλη έχουν αμοιβαία εμπιστοσύνη ή έχουν το δικαίωμα να ελέγχουν κατά πόσο έγινε η πιστοποίηση στο κράτος προέλευσης. Με βάση τους διαδικαστικούς κανόνες θα σας ενημερώνω τακτικά και για τις επόμενες διαπραγματεύσεις ο επόμενος ε, τριμερής διάλογος θα λάβει χώρα στι 25 Απριλίου, 28 ε, και 29 Μαΐου και η τεχνική συνεδρίαση στι 25 Μαρτίου. Αυτά και περιμένω τις απορίες, τα σχόλια ή τις παρατηρήσεις. Δεν βλέπω να θέλει κανείς το λόγο, οπότε μπορούμε να περάσουμε στο σημείο 8 της ημερήσιας διάταξης που περιλαμβάνει έκθεση για την αντιπροσωπή της Επιτροπής απασχόληση και Κοινωνικών υποθέσεων, υποθέσεως στο Δουβλίνο στις 11 και 12 Φεβρουαρίου 2013. για συνάντηση με την Ιρλανδική Προεδρία. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι αυτή η αντιπροσωπεία την οποία δίφθηνα απαρτίζονται από τον κύριο Όρη, ο συντονιστή του ΕΛΚ, τον κύριο Σερκάς, των Σοσιαλδημοκρατών, την κυρία Ζιν Λομπέρ, υπεύθυνη των Πρεσίνων και επίσης είχαν έρθει και δύο Ιρλανδοί συνάδελφοι, η κυρία Αρκίνα από τους Φιλελεύθερους και η κυρία Μερκέστερολ από ε, το S&D. Στη διάρκεια αυτής της επίσκεψης συναντήσαμε τον αρμόδιο υπουργό για την απασχόληση, τις επιχειρήσεις και τις καινοτομίες, με τον οποίο συζητήσαμε με βάση τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 7 και 8 Φεβρουαρίου, υπενθυμίζοντας την σημασία που αποδίδει το Κοινοβούλιο στη διατήρηση του Ταμείου Προσαρμογής και ε, παγκοσμιοποίησης. Επίσης συναντήσαμε εκπροσώπους οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, το National Youth Council of Ireland, το European Anti-Poverty Network της Ιρλανδίας, γνωρίζουμε τους εκπροσώπους τους εδώ στις Βρυξέλλες, την Εθνική Οργάνωση Ιρλανδίας ε, των Ανέργων και το Σκίνετ. Επίσης συναντήσαμε την κυρία Λούσιντα Κρέτον, Υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, η οποία μας εντυπωσίασε πολύ σχετικά με την κινητικότητά της και τις ικανότητάς της να περιλάβει τους δικούς μας προβληματισμούς ε, στο χαρτοφυλάκιό της. Επίσης, επισκεφθήκαμε ε, την Ακαδημία Digital Skill, ψηφιακών ικανοτήτων, δεξιοτήτων που μας έδειξε μια διαδικασία χρησιμοποίηση ε, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου που προορίζεται κυρίως στην ανακύκλωση ε, στον ψηφιακό κόσμο. Αν δείτε λοιπόν αυτά τα οποία χρησιμοποιεί ο πρόεδρος Μπαρόζο στο scoreboard που παρουσίασε στην ομιλία του την τελευταία φορά ε, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ένα πίνακα τον οποίο σας καλώ να κοιτάξετε που δείχνει τον διαχωρισμό ανάμεσα στα αιτήματα ε, όσον αφορά τα προσόντα στο ψηφιακό τομέα και τον αριθμό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Η μία καμπύλη πηγαίνει προς τα πάνω, έπρεπε να κάνω έτσι μάλλον, είναι ανωδική απόλυτα, ενώ η προσφορά για εκπαιδευτικά προγράμματα ε, είναι μια γραμμή ίσια. Εδώ δεν πρόκειται για αρχική εκπαίδευση, αλλά μετεκπαίδευση, για τα άτομα που έχουν προβλήματα στην αγορά εργασίας. Αυτό το πρόγραμμα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Επίσης έγινε μια επικοδομητική ε, ανταλλαγή απόψεων με την Υπουργό John Burton, Υπουργό Κοινωνικής Προστασίας, όπου μιλήσαμε για ε, τις εργασίες ΕΠΣΚΟ, τις μελλοντικές εργασίες ΕΠΣΚΟ, κυρίως όσον αφορά ε, τις εγγύσεις για τους νέους και την κινητικότητα σε σχέση με τα κοινωνικά διακυβεύματα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, διότι όπως γνωρίζετε το Συμβούλιο ΕΠΣΚΟ συνεδρίασε 28 Φεβρουαρίου με τον πρόεδρο Herman von Rompuy στα πλαίσια της προετοιμασίας ε, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ιουνίου για ε, τον προσανατολισμό προς μια πραγματική Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Κατόπιν συναντήσαμε τους κοινωνικούς εταίρους, ε, σύμφωνα με μια πολύ γνωστή πρακτική. Συγκεκριμένα, την Συνομοσπονδία Απασχόλησης και Irish Congress of Trade Unions, τα συνδικάτα. Στις 12 Φεβρουαρίου επισκεφθήκαμε το Belgian Youth Resource Center που ασχολείται με νέους ε, στα περίχωρα παρουσιάζουν δυσκολίε ε, στα πιο φτωχά περίχωρα του Δουβλίνου και συναντήσαμε τον Υπουργό, τον Αρμόδιο για την εκπαίδευση και τα επαγγελματικά προσόντα με τον οποίο συζητήσαμε διαμακρόν το θέμα της πρωτοβουλίας Επιτροπής ε, για το Use on the Move στις περισσότερες ε, από αυτές τις συναντήσεις υπογραμμίσαμε τις προτεραιότητες της Επιτροπής μας, δηλαδή τη δυνατότητα να ε, έχουμε 25% ε, των δαπανών του Ταμείου Συνοχής για ε, το Ταμείο. Θα το λάβετε γραπτός αυτό το έγγραφο. Αν όσοι με συνόδευσαν επιθυμούν να υπογραμμίσουν ορισμένες άλλες πλευρές αυτής της επίσκεψης, κάτι το οποίο παρέλειψα. Παρακαλώ να το κάνετε τώρα. Η κυρία Έμερ Καστέλ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που ήσασταν επικεφαλής ε, της αντιπροσωπείας αυτή την συνάντηση στο και ήταν πολύ ενδιαφέρουσα άσκηση για μένα. Το γεγονό ότι ασχοληθήκαμε και με του κοινωνικού εταίρου και συναντήσαμε πολλέ άλλε ομάδε. Επίσης ήθελα να πω ότι το feedback ε, και τα, οι αντιδράσει τη ομάδα ήταν όλα πολύ θετικά. Και είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι οι κοινωνικοί εταίροι και οι ΜΚΟ καταλαβαίνουν πολύ καλά ότι τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προβληματίζονται σχετικά με όλα αυτά τα θέματα. Η Ιρλανδία αντιμετωπίζει πολύ μεγάλα προβλήματα και οι ευρωβουλευτές που επισκέφθηκαν το Δουβλίνο αυτές τις λίγες μέρες είδαν την εικόνα και κατάλαβαν το μέγεθος των προβλημάτων μας και τις επιπτώσεις που έχουν στον πληθυσμό γενικότερα. Το θέμα της ε, ανεργίας κυρίως των νέων θίγει ε, ε, επανειλημμένα. Ενώ αναγνωρίσαμε και καταλαβαίνουν και οι υπουργοί και οι ευρωβουλευτές ότι πρέπει να χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά τα κονδύλια του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, Υπάρχουν ορισμένοι προβληματισμοί σχετικά με την εφαρμογή του ΕΣΕΦ και των διαφόρων προγραμμάτων. Γι' αυτό θα ήθελα να επισημάνω ε, τη, χρήση του Ταμείου για τους νέους. Σημείωσα τα θέματα που αναφέρθηκαν σχετικά με την συνεχή επιμόρφωση των νέων, τα προγράμματα τα οποία έχουν οργανωθεί και τη σημασία να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας. Γι' αυτό το ε, λόγο τα προγράμματα επιμόρφωσης είναι πολύ χρήσιμα, καθώς και η εργασία τους μέσα σε επιχειρήσεις. Και πρέπει λοιπόν να εστιάσουμε την προσοχή μας περισσότερο στην δημιουργία θέσεων εργασίας. Υπάρχουν ορισμένα θέματα τα οποία επίσης θα ήθελα να αναφέρω ε, σχετικά με την εφαρμογή αυτής της εγγύησης για τους νέους όσον αφορά το επίπεδο συμμετοχής των νέων, όχι μόνον άλλο ένα πρόγραμμα προκειμένου να προσφερθεί ένα μάθημα, ένα πρόγραμμα και στο τέλος του προγράμματος αναμένεται ότι θα μπορέσουν να βρουν δουλειά. Αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει να λάβουμε υπόψη. Απλά θα ήθελα να πω ότι η επίσκεψη, ε, η επίσκεψή μας έγινε δεχτή Ήταν, η υποδοχή του ήταν πολύ θερμή διότι έγινε αντιληπτό ότι οι ευρωβουλευτέ βρίσκονται κοντά στους πολίτες όχι μόνο ε, να δούμε του υπουργού και του κοινικού εταίρου, αλλά επισκεφθήκαμε τη χώρα και αυτό ήταν πολύ σαφές. Είδαμε ορισμένα προγράμματα και πώς χρησιμοποιούνται τα κονδύλια του Κοινωνικού Ταμείου. Συμφωνώ μετά όσα υπόθηκαν ότι φυσικά ο διάβολος βρίσκεται στις λεπτομέρειες και χρειάζεται πολλά να γίνουν για την εφαρμογή αυτών των προγραμμάτων. Thank you. Any other remark? Υπάρχουν άλλες παρατηρήσεις? Όχι. Ολοκληρώνουμε λοιπόν το σημείο αυτό. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κυρία Κοστέλο και για τα όσα είπατε. και με 7 λεπτά καθυστέρηση φτάνουμε στην ψηφοφορία. Θα ήθελα να σας πω ότι ο συντονιστής από το ΕΛΚΑ παραπονέθηκε γιατί ε, ψηφίζουμε στην στο πρώτο αυτό τμήμα της συνεδρίασης. Σας ε, λέω ότι είναι δικιά μου η πρωτοβουλία αυτή, προκειμένου να καταφέρουμε να δώσουμε τη δυνατότητα στις πολιτικές ομάδες να συνεδριάσουν εκ των προτέρων. Χαίρομαι επίσης ε, πάρα πολύ όταν βλέπω ότι κάθε φορά υπάρχει μια παρέκκληση γίνονται και παρατηρήσεις, γιατί για παρέκκληση πρόκειται αυτή τη φορά. Συνήθως συνεδριάζουμε, όπως σας είπα, την ε, δεύτερη μέρα. Προσπαθήσαμε να περιορίσουμε την ψηφοφορία πάρα πολύ σήμερα. Ξέρω ότι η βασική ψηφοφορία θα γίνει αύριο. Ουσιαστικά εδώ πέρα έχουμε δύο εκθέσεις, την έκθεση του κυρίου Ουγγουρεάνου όσον αφορά την ετήσια έκθεση σχετικά με την πολιτική ανταγωνισμού και μία γνωμοδότηση θα ψηφίσουμε όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για την Ιταλία, για την επιχείρηση Αντώνιο Μερλόνι, αν θέλουμε οι δύο αυτές επιτροπές ε, στις οποίες υποβάλλουμε γνωμοδότηση να λάβουν υπόψη τη γνωμοδότησή μας, πρέπει να ψηφίσουμε σήμερα. Γι' αυτό το λόγο ψηφίζουμε κατ' εξαίρεση σήμερα τις δύο αυτές εκθέσεις. Ο κύριος Όρη έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Όντως ε, παραπονέθηκα για την ακολουθητέα διαδικασία. Το πρόβλημα μου δεν είναι ότι ψηφίζουμε σήμερα ή ότι ψηφίζουμε αύριο, γιατί καταλαβαίνω ότι υπάρχουν περιστάσεις, πολλές φορές μας υποχρεώνουν να ψηφίζουμε διαφορετικές στιγμές από ό,τι ήθιστε. Το πρόβλημά μου είναι ότι το μάθαμε τελευταία στιγμή αυτό. Υπάρχουν κάποιοι συνάδελφοι οι οποίοι ε, έχουν άλλε συνειδημένες υποχρεώσει, επομένω δεν μπορούν να είναι εδώ πέρα σήμερα για να ψηφίσουν. Ξέρετε ότι υπάρχουν ορισμένοι συναδελφοί οι οποίοι θα ήθελαν να βρίσκονται σήμερα στην ε, σημερινή ψηφοφορία, αλλά δυστυχώ ενημερώθηκαν για την αλλαγή στο πρόγραμμα την τελευταία στιγμή. Επ' αυτού ουσιαστικά θέλω να υποβάλω μια παρατήρηση. Επομένω, κάθε φορά που τροποποιείται η ημερήσια διάταξη, κάθε φορά που πρέπει να προσθεθούν νέα σημεία στη ημερήσια διάταξη, κάθε φορά που προβλέπεται μια ψηφοφορία νωρίτερα από ό,τι συνήθω διεξάγεται στην Επιτροπή μας, θεωρώ ότι θα πρέπει να ενημερωνόμαστε εν γέρος προκειμένου να αποφύγουμε τέτοια προβλήματα. Δηλαδή να υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι πολύ απλά δεν μπορούν να παραστούν ακριβώς επειδή έχουν άλλες υποχρεώσεις αλλού. Επομένως θα θέλαμε και η Πρόεδρος αλλά και η Γραμματεία να μας ενημερώνουν ή δυνατόν νωρίτερα. Κύριε Ορή, συγγνώμη που θα σας πω ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως τα παρουσιάζετε. Όλοι οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν ακολουθώντας ένα πολύ αυστηρό χρονοδιάγραμμα. Πολύ εγκαίρος λοιπόν. Ήδη από τη συνεδρίαση των συντονιστών είχαμε πει ότι θα ψηφίζαμε κατά αυτόν τον τρόπο, δηλαδή σήμερα το πρωί, και το είχαμε πει τότε ξεκάθαρα, εγκρίνοντας με τους συντονιστές το χρονοδιάγραμμα για τη σημερινή και τις επόμενες συνεδριάσεις. Η γραμματεία επίσης σε ενημέρωσε εγκαίρως, έτσι ώστε να καταφέρει να προσαρμόσετε το πρόγραμμά σας και να μπορεί να λειτουργεί ομαλά η Επιτροπή μας. Λοιπόν, κατά τη συνεδρίαση συντονισμού ήδη από το Φεβρουάριο είχαμε αποφασίσει για το χρονοδιάγραμμα το οποίο ακολουθούμε. Εν συνεχεία δεν έγινε καμία τροποποίηση στην ημερήσια διάταξη και έτσι λοιπόν σας απεστάλλει η ημερήσια διάταξη ήδη την προηγούμενη εβδομάδα όσον αφορά τη σημερινή μας συνεδρίαση. Λοιπόν, χωρίς άλλη καθυστέρηση θα ήθελα να προχωρήσουμε στο σημείο 9 της ημερήσιας διάταξης και να ψηφίσουμε την έκθεση του κυρίου Ουγγουρεάνου όσον αφορά την ετήσια έκθεση σχετικά με την πολιτική ανταγωνισμού. Εξετάσαμε σήμερα το πρωί λίγο νωρίτερα τις συμβαστικές τροπολογίες τις οποίες έχουν, οι οποίες έχουν κατατεθεί. Αν δεν υπάρχουν άλλες παρατηρήσεις, ας ξεκινήσουμε με την ψηφοφορία της τροπολογίας 2 για την παράγραφο 1. Λουτβίσον Κέρκας Καστέξιπερ, κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 3 Φιλίπ Μπουλόν υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 4 πάντα για την παραγραφό 1 Λουγκδίσον υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία Α από τρεις πολιτικές ομάδες υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 1. Συμβαστική τροπολογία Β από τρεις πολιτικές ομάδες υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 2, τροπολογία 7, Λούντβιτσον Καστέξ, υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 2, τροπολογία 9, διορθώνει η Πρόεδρος, τροπολογία 8, υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτεται. Παράγραφος 2, τροπολογία 9 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 2, τροπολογία 10, Λούντβιτσον σέρκα Κάστεξ, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 2, τροπολογία 11 του εισηγητή υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 12 και 13 αποσύρονται. Περνάμε στην παράγραφο 3, τροπολογία 14, Λούντβιντσον Θέρκας, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 3. Συμβαστική σε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 3. Τροπολογία 16 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 17 έχει αποσυρθεί, 18 για την παράγραφο 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 19 για την παράγραφο 4 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παραγραφος 4 τροπολογία 20 του συγητή υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 5 τροπολογία 21 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 5 τροπολογία 22 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 5 τροπολογία 23 του συγητή υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Εκτιμώντας Παράγραφος Β, τροπολογία 1 από τους Λούτβιτσον Καστέξ, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ψηφίσουμε το σύνολο του κειμένου ηλεκτρονικά. Άρτη ψηφοφορία. Και εγώ δεν έχω την κάρτα μου. Έχετε όλη την κάρτα σας. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. «32 υπέρ, μία ψήφος κατά, μία αποχή. Συγχαρητήρια στον εισηγητή μας. Κύριε συγητά, Α είστε πολύ προσεκτικό τώρα με την Επιτροπή Οικονομικών Θεμάτων προκειμένου να λάβει στο μέγιστο υπόψη τις παρατηρήσει μας, αυτά τα οποία εγκρίναμε με την ψήφο μα Σημείο 10. Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση όσον αφορά την επιχείρηση Αντώνιο Μερλόνι στην Ιταλία. Πρόκειται για μια επιχείρηση Τι ακριβώ κάνει αυτή η επιχείρηση, λέει πρόεδρος. κατασκευάζει οικιακές συσκευές. Όντως, οικιακές συσκευές λοιπόν κατασκευάζει. Ας ψηφίσουμε λοιπόν την επιστολή που αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης και συμφωνίας στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας για το Ταμείο Κινητοποίησης Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση και συνδέεται με την έκθεση του κυρίου Νταρντέν στην Επιτροπή Προπολογισμών, όπου θα γίνει ψηφοφορία σχετική αύριο. Ποιο είναι υπέρ τη επιστολή. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Θέλετε να. Μάλλον, ας κάνουμε μια ηλεκτρονική επαλήθευση, σας παρακαλώ πολύ. Άρτη ψηφοφορία. πέρας. 31 υπέρ, μία ψήφος κατά, δύο αποχές. Δεν εγκρίθηκε ομοφόνος, αλλά εγκρίνεται παρόλα αυτά. Ολοκληρώσαμε λοιπόν με τις ψηφοφορίες. Donc, au point. Περνάμε στο σημείο 11 λοιπόν. Τη δημόσια κρόαση δηλαδή που οργανώνουμε σχετικά με την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων και τις πιθανές διεξόδους. Η οργάνωση δημόσια κρόσης γίνεται στα πλαίσια της έκθεσης ε, ίδιας πρωτοβουλίας ε, της κυρίας Ξιντλεύσκα. Μάλιστα, οι Επιτροπές Γυναικών και Πολιτισμού θα συντάξουν γνωμοδότηση της έκθεσης κυρίας Ξιδλεύσκα. Σας καλωσορίζω όλους στην δημόσια ακρόαση και θα ήθελα να δώσω το λόγο πρώτα στην εισηγήτριά μας, την κυρία Ξιδλεύσκα, για να μας κάνει μια σύντομη εισαγωγή στο θέμα της δημόσιας ακρόασης. Το θέμα αυτό μας απασχόλησε επανειλημμένο στο παρελθόν όταν ε, η Έμιλι Τουρίνεν είχε συντάξει σχετική έκθεση και κατόπιν η υποφαινομένη υπέβαλε προφορική ερώτηση με ψήφισμα στην Ολομέλεια με το ίδιο θέμα. Τελικά η πρωτοβουλία μας απέδωσε καρπούς γιατί στο πρώτο τελευταίο συμβούλιο συνήθιζε και στη Σύνοψη συμφωνία για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων ανέλαβαν την στρατηγική πρωτοβουλία να θεσπίσουν ένα ταμείο εγγύσεων για τους νέους ε, με 6 δισεκατομμύρια ευρώ πρικοδότηση και μάλιστα στα πλαίσια της Μωράν Σαρτιάν για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο εξετάζουμε και το θέμα αυτό του Ταμείου Εγγύσεων για τους Νέους και στα πλαίσια της έκθεσης ε, του συναδέλφου Τεκόζα για το κανονιστικό πλαίσιο το γενικό κανονιστικό πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων. Πέραν του όμως, έχουμε και την δεδηλωμένη βούληση των συντονιστών να συντάξουμε μια ειδική έκθεση για αυτό το πακέτο που αφορά την απασχόληση των νέων. Θα δώσω λοιπόν το λόγο για μια σύντομη εισαγωγή στην ε, εισηγήτριά μας, την κυρία Καταζίνα Σιλεύσκα. Παρακαλώ κυρία εισηγήτρια, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι. Εξετάζοντα εξετάζοντας την έκθεση αυτή και τα μέσα και τους μηχανισμούς που έχουμε για τους νέους, καθώς και τα μελλοντικά μέτρα που θα θεσπιστούν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, όπως το Ειδικό Ταμείο Εγγύσεων για τους Νέους που ανέφερε η Πρόεδρος, ε, συνειδητοποίησα πόσο σημαντική είναι μια πολυδιάστατη προσέγγιση στο πρόβλημα αυτό. Χρειαζόμαστε λύσεις που δεν ε, θα βελτιώσουν ε, γρήγορα και βραχυπρόθεσμα μόνο την κατάσταση, γιατί τέτοια, τέτοια μέτρα είναι ευαλωματικά. Χρειαζόμαστε μακρόπνομα, μακροθο, μακρόπνομα μέτρα για να επιλύσουμε το διαρθρωτικό πρόβλημα της ενεργείας των νέων. Επίσης, θα πρέπει ε, να συνδυάσουμε τα συστήματα κατάρτισης με τις σωστές επαγγελματικές πρακτικές και να προετοιμάσουμε τους νέους ε, ε, για την εργασία με τρόπους που θα εξυπηρετούν και τους εργοδότες και να προσαρμοστούμε στις ανάγκες της αγοράς, να βοηθήσουμε σωστά τον επαγγελματικό τους προσανατολισμό. Γι' αυτό χρειαζόμαστε τη συνεργασία και των πανεπιστημιακών κύκλων, των επιχειρηματιών, των γραφείων ανέβρεση εργασίας, αλλά και των ίδιων των νέων, που είναι οι άμεσα ενδιαφερόμενοι να ενταχθούν το συντομότερο δυνατό στο, στην αγορά εργασίας. Επίσης, χρειαζόμαστε ε, παιδεία ε, που θα δώσει εφόδια στους νέους και τεχνικές δεξιότητες και όχι μόνο μια θεωρητική γνώση που θα τη λαμβάνει στη διάρκεια τη παιδεία. Χρειαζόμαστε και άτυπε ανεπίσημε μορφέ κατάρτιση. Επίση, θα πρέπει οι νέοι να έχουν πρόσβαση στον ε, επαγγελματικό προσανατολισμό, ώστε ήδη να προετοιμάζουν το μέλλον του από το Λύκειο και να συνειδητοποιήσουν πώ οι επαγγελματικέ επιλογέ ε, θα επηρεάσουν το μέλλον του και να γνωρίζουν και πώ λειτουργεί η αγορά εργασία. Επίση, είμαι υπέρμαχο ε, τη ενίσχυση του επιχειρηματικού πνεύματο των νέων. Και μάλιστα εγώ ίδια όταν ήμουν 18 χρονών ξεκίνησα δική μου επαγγελματική δραστηριότητα και σίγουρα δεν μετανιώνω για την επιλογή μου. Ενθαρρύνω λοιπόν τους νέους να αναλάβουν πρωτοβουλίες, να αναπτύξουν τα ταλέντα τους, τις δεξιότητές τους και το επιχειρηματικό τους πνεύμα. Φυσικά για κάτι τέτοιο χρειάζονται μια κρατική βοήθεια με τη, μορφή ίσως επιχορηγήσεων και τη διευκόλυνση των διοικητικών δομών τα κονδύλια που θα αξιοποιηθούν ε, θα πρέπει να βρίσκονται στους κρατικούς προϋπολογισμούς και στον κοινωτικό προϋπολογισμό ε, ε, γιατί θα χρειαστούν πολλά μέσα για να ενισχύσουμε τους νέους προκειμένου να ενταχθούν δραστήρια στην αγορά εργασίας. Όλες αυτές οι δραστηριότητες θα πρέπει να γίνονται παράλληλα με τις δραστηριότητες των κρατών μελών και στόχο θα πρέπει να έχουν την ανάκαμψη της οικονομικής ε, ανάπτυξης και την οικονομική μεγέθυνση. Θα πρέπει να εφοδιαστούμε με πολλά μέσα, να βοηθήσουμε τους νέους να αποκτήσουν και σωστή εκπαίδευση αλλά και σωστή επαγγελματική κατάρτιση και να μην ξεχνούμε τις ανάγκες των επιχειρήσεων, ώστε να προετοιμάζουμε τους ε, νέους, ώστε να προσαρμόζονται στις αγορές ε, ε, στις ανάγκες αγοράς εργασίας. Κύριε γιατί παρακαλώ ε, περιοριστείτε στην υποβολή ερωτήσεων προς καλεσμένους μας, γιατί θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε την παρουσίαση της δικής σας έκθεσης. Τώρα να εκμεταλλευτούμε τη δημόσια κρόση για να υποβάλουμε συγκεκριμένες ερωτήσεις στους καλεσμένους μας. Ναι, χαίρομαι ιδιαίτερο για την ε, οργάνωση αυτής της δημόσιας ακρόασης και την παρουσία των προσκεκλημένων εμπειρογνωμόνων και πιστεύω ακράδαντα ότι οι παρατηρήσεις που θα ακούσουμε και οι συστάσεις τους για την υποστήριξη των νέων ε, και η παρουσίαση των δικών τους εμπειριών θα μας βοηθήσουν και στη σύνταξη της έκθεσης. Θεωρώ ότι οι σημερινοί μας καλεσμένοι εμπειρογνώμονες θα μας δείξουν ε, ποια είναι η σωστή πολυδιάστατη αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, ώστε να μην συντάξουμε απλώς ωραία έγγραφα που θα τα γνωρίζουμε όλοι ότι υπάρχουν, αλλά που θα έχουν και μία έμπρακτη εφαρμογή και που θα μας επιτρέψουν να επιλύσουμε το πρόβλημα της ανεργίας των νέων. Αυτό περιμένω λοιπόν από τους εμπειρογνώμονες και θεωρώ ότι το ζήτημα των ανεργών και της ανεργίας είναι ένα κοινό μέλημα όλων, άσχετα από την πολιτική μας ιδεολογία. Και ελπίζω από κοινού όλοι μαζί με τα μέλη της Επιτροπής Απασχόλησης και με τους εμπειρογνώμους και τη βοήθειά τους θα καταλήξουμε σε έγγραφο που θα είναι αποτελεσματικό και θα μας δώσει κάποιες λύσεις για το μέλλον. Να δώσουμε στους νέους ευκαιρία να γίνει μια γενιά που δεν θα είναι η χαμένη γενιά, αλλά μια γενιά που θα μπορέσει να υλοποιήσει τα όνειρα και τις προσδοκίες της. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Μπορώ να δώσω τώρα το λόγο στους πέντε προσκεκλημένους μας. Χρειάστηκε να τους επιλέξουμε, συμμετείχαν πολλά μέλη της Επιτροπής μας. Θεωρώ ότι έχουμε μία κατάλληλη ισορροπία πλέον εδώ πέρα. Βλέπω ότι μολονότι μιλάμε εδώ πέρα για την ενεργεία των νέων, δυστυχώς προσκεκλημένους μας δεν υπάρχει ούτε μία γυναίκα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Λοιπόν, δίνω ευθύ αμέσω το λόγο για το Πανεπιστήμιο. Συγγνώμη για τον τρόπο που θα το προφέρω τουλάχιστον την πρώτη φορά, θα το διορθώσω μετά, Πανεπιστήμιο Γιατζελόνιαν της Κρακοβίας. Δίνω ευθύ αμέσως το λόγο στον κύριο Γιάροσλαβ Γκόρνιακ. Έχετε το λόγο για πέντε λεπτά. Dziękuję. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι αδιαφυσβήτητα τα γεγονότα ότι έφτασε στα ύψη η ανεργία των νέων και ε, δυστυχώς αυτή η μάστιγα πια έχει χτυπήσει όλες τις χώρες. Είναι ακαθόδες και φλέγον το ζήτημα. Θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με μεγαλύτερη πολιτική ευθύνη λοιπόν. Είναι σημαντικά τα μηνύματα που θα στείλουμε. Καταρχήν θα πρέπει να πιστούμε ότι ε, αξίζει να επενδύσουμε στο ανθρώπινο κεφάλαιο των νέων, που είναι σημαντικό για την οικονομική ανάπτυξη, αλλά και σημαντικό ε, δεδομένων των δημογραφικών απειλών. Επίσης θα πρέπει να δούμε τι γίνεται μετά την ολοκλήρωση των ε, σπουδών των νέων και το, το πρόβλημα της εγκατάλειψης των σπουδών πολλές φορές από τους νέους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε ένα ταμείο εγγυήσεων για τους νέους ε, και την εξασφάλιση σε όλους τους νέους ε, μέχρι τα 25, σωστές, ε, σωστών ευκαιριών πρόσληψης, σωστής παιδείας, δυνατότητες επαγγελματικού στάζ τετράμενου και διαφόρων άλλων μέτρων. Φυσικά αυτή με, η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής δημιουργεί πολλά προβλήματα και πολλά, προβλημα, πολλά ερωτηματικά ως προς την αμοιβή ή όχι των νέων για κάποια επαγγελματικά στάσεις και καταρτήσεις. Υπάρχουν διάφοροι μηχανισμοί που θα πρέπει να περιλαμβάνει η πολιτική. Το σύστημα εγγύσεων των νέων ε, η, λαμβάνει ως τεκμήριο το γεγονός ότι οι, οι νέοι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες των επιχειρηματιών, γιατί οι επιχειρηματίε δεν πρόκειται οι ίδιοι να επενδύσουν σε μέσα για την προετοιμασία των μελών, μελλοντικών τους ε, εργαζομένων. Δεν είναι θέμα δεξιοτήτων και εφοδίων, αλλά η ανεργία των νέων ε, οφείλεται κυρίω ε, στην οικονομική ύφεση, στη μεγάλη ανεργία, αλλά και σε κάποιου θεσμικού παράγοντε Σε πολλέ χώρε, ο συνδυασμό αυτών των τριών παραγόντων οδήγησε σε μια έκρηξη της ανεργίας των νέων. Επίσης, έχουμε την οικονομική κρίση και μια ανεργία που φυσικά αυξάνεται όταν οι οικονομικές συνθήκες είναι χαλεπές. Ε, και οι επιχειρηματίες εξαιτία οικονομικής κρίσης ε, περιορίζουν τις θέσεις απασχόλησης αντί να δημιουργούν νέους. Έτσι προσπαθούν να, να κάνουν μια καλύτερη αξιοποίηση του δυναμικού τους, γι' αυτό και χρειάζεται ένας μηχανισμός υποστήριξης. Γιατί πολύ περισσότεροι χάνουν ε, θέσεις απασχόληση από ό,τι προσλαμβάνονται. αν δεν ε, στηρίξουμε λοιπόν την οικονομική ανάπτυξη δεν πρόκειται να επιλύσουμε το πρόβλημα της ανεργίας. Επίσης θα πρέπει να μην λάβουμε υπόψη μόνο ορισμένου κινδύνου, όπως τη δημογραφική απειλή. Γιατί μερικές ε, χώρες έχουν κάποιες πολιτικές στήριξης ε, της ε, πρόσληψης, αλλά αποκαλύπτουν όλους, όλες τις ηλικιακέ ομάδες, τους νέους, τους ηλικιωμένους, τις γυναίκες και σε περιπτώσεις οικονομικής κρίσης είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστούν όλα αυτά τα μέτωπα. Επίσης υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι σε σχέση με τις πολιτικές που ε, σχέση με τις απειλές ε, ε, για, την, για τους νέους που έχουν σταματήσει τις σπουδέ τους ή που δεν παρακολουθούν κανένα στάζ επαγγελματική κατάρτισης. Αυτοί οι νέοι ε, μερικές φορές παρόλο που αναζητούν εργασία δεν τη βρίσκουν ή μερικές φορές άτομα με ειδικές ανάγκες. Χρειάζονται ιδιαίτερη υποστήριξη προκειμένου να βρουν μια θέση απασχόλησης μερικές φορές ε, ε, και σε ορισμένου τομεί μειώνονται οι θέσει εργασία. Επίση, θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με την παιδεία. Ε, και η παιδεία έχει κάποιο κόστο. Είναι δυστυχώ αναποτελεσματικά κάποια μέτρα πολιτική για για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων. Θα πρέπει στις νέες μας προτάσεις να λάβουμε υπόψη και τη μέχρι τώρα αναποτελεσματικότητα των νέων. Υπάρχουν ε, πολλά, πολλά εμπόδια και για τους επιχειρηματίες, φορολογικά, διοικητικά, θεσμικά. Ε, νέοι που δεν έχουν εμπειρία επαγγελματική αντιμετωπίζουν πολύ μεγαλύτερα εμπόδια γιατί δεν μπορούν να ξεκινήσουν μια επαγγελματική δραστηριότητα ή να αναζητήσουν θέση γιατί οι επιχειρηματίες ζητούν προηγουμένως επαγγελματική πείρα. Ε, Επίσης, ε, δεν θα πρέπει να περιοριστούμε μόνο στου νέου μέχρι 25 χρονών, γιατί ε, έχουμε νέους που σπουδάζουν πολύ περισσότερο. Έχουν πιο ειδικευμένες σπουδέ, αλλά και αυτοί αντιμετωπίζουν ε, τη μάστιγα της ανεργίας. Θα πρέπει λοιπόν να, να λάβουμε υπόψη την υπερβολική δίκευση μερικές φορές των και να τους λάβουμε υπόψη. Οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι καλές, αλλά χρειαζόμαστε νέα προοπτική. Μια σωστή ε, προοπτική ε, και πολιτική απασχόληση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και την πολιτική της οικονομικής ανάπτυξης. Να προετοιμαστούμε και για το θα συμβεί μετά την κρίση. Θα πρέπει να προετοιμάσουμε σωστά τα, ε, τους νέους για, τις, για την αγορά εργασίας Γι' αυτό και χρειαζόμαστε κάποιε πρωτοβουλίε που θα είναι σημαντικέ για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα. Θα πρέπει σε όλα τα κράτη-μέλη να εφοδιάζονται οι νέοι με τα κατάλληλα προσόντα και εφόδια, γιατί θα πρέπει να ξεχνούμε ότι οι νέοι δεν θα περιοριστούν μόνο στη χώρα τους, αλλά θα εργαστούν και στο εξωτερικό. Στην Πολωνία ε, έχουμε στείλει μέχρι και 2 εκατομμύρια νέους στην αλλοδαπή εργασία. Είναι σημαντικό και το θέμα των εγγύσεων για τους νέους. Βέβαια, επικοινωνιακά ίσως δημιουργεί ε, υπερβολικές προσδοκίες ότι ε, οι δημόσιοι φορείς θα εξασφαλίσουν για για τον κάθε νέο αξιοπρεπή απασχόληση. Βέβαια εδώ έχουμε θέμα ποιότητα και ποσότητας της προσφοράς εργασίας από άποψη μισθού και συνθήκων. Θα πρέπει να προτείνουμε κάποια συνετά μέτρα ώστε να αυξηθεί η ποιότητα, αλλά αυτό δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε μείωση των προσφορών εργασίας εκ μέρους των επιχειρηματιών. Βέβαια, εδώ δεν μιλούμε για τις χώρες όπου ε, το διπλό σύστημα εκπαίδευσης και επαγγελματική κατάρτισης λειτουργεί σωστά, αλλά στις χώρες που αντιμετωπίζουν προβλήματα ή ε, σε χώρες που οι νέοι δεν έχουν μεγάλη πρόσβαση ούτε σε παιδεία ούτε σε επαγγελματική κατάρτιση. Επίση θα πρέπει να δίνεται δυνατότητα στου νέου για παράταση των σπουδών και να είναι ποιοτική τέτοια δυνατότητα. Οι προτάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παιδεία και την επαγγελματική κατάρτιση δημιουργεί ένα σημαντικό πακέτο επενδύσεων για τους νέους και ενίσχυση της κινητικότητας. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη της ανάγκης μεγάλης ειδίκευσης, ανάπτυξη των δεξιοτήτων, αλλά και πρόσβαση σε τέτοιου είδους εκπαιδευτικό συστήματα. Δεν αρκούν ούτε τα χρήματα, ούτε οι κανόνες. Θα πρέπει να στηρίξουμε και τη ζήτηση και την προσφορά γιατί ε, αν επικεντρωθούμε, μόνο στη ζήτηση, μόνο στην προσφορά, δεν θα καταλήξουμε σε ε, ικανοποιητικές λύσεις. Ε, βέβαια, μερικές χώρες έχουν πολύ πιο μακροχρόνιες παραδόσεις και πολύ πιο πρόσφατες παραδόσεις, ώστε ο επαγγελματικός προσανατολισμός που προσφέρουν οι σύμβουλοι να είναι πολύ πιο αξιόλογος. Επίσης, θα πρέπει να ε, βελτιώσουμε και τα εκπαιδευτικά συστήματα και τα συστήματα επαγγελματική κατάρτισης, ώστε ε, να δίνουμε δυνατότητα για στάζ ε, πολύμηνα που θα είναι όμως και υψηλή ποιότητα. Χρειαζόμαστε και ποιοτική παιδεία αλλά και επιχειρήσεις που θα μπορούν να προσφέρουν κατάλληλες πρακτικές και στάζ. Θα πρέπει να απαιτούμε την ποιότητα αλλά να μπορούμε να την ελέγχουμε και να τη διαδίδουμε και γι' αυτό χρειάζεται φυσικά διεθνή συνεργασία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πολύ σωστά θέλει να χρησιμοποιήσει το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για να υλοποιήσει αυτέ τι σημαντικέ πολιτικέ, Αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη κυρίως το θέμα της εφαρμογής. Γιατί ε, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την αξιοποίηση των κονδυλίων και την, αποτελεσματικέ δραστηριότητε. Γιατί αν δεν ε, πιάνουν τόπο τα χρήματα, και δεν μπορούμε να ποσοτικοποιήσουμε την, την, την αποτελεσματικότητα αυτών των προγραμμάτων, δεν θα οδηγηθούμε πουθενά. Επίσης θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την ανάγκη πολιτικών που θα στηρίζονται σε ποσοτικοποιημένα αποτελέσματα και φυσικά για κάτι τέτοιο χρειαζόμαστε συστημικές λύσεις και την υποστήριξη τέτοιων συστημικών λύσεων από την διαρθρωτική πολιτική. Ε, φυσικά ε, οι παρεμβάσεις της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ε, ελέγχονται και να ποσοτικοποιούνται. Να δούμε ποια είναι τα αποτελέσματα με βάση κάποιους δείκτες που θα είναι συγκεκριμένοι. Θα πρέπει οπωσδήποτε να ελέγχουμε τον αντίκτυπο των πολιτικών μας. Το πακέτο βέβαια εγγύσεων για τους νέους θα είναι ε, αρκετή πρόκληση για πολλές χώρες, αλλά πιστεύω ότι αξίζει να επενδύσουμε στο δυναμικό αυτό που είναι πολύ σημαντικό, το δυναμικό των νέων. Ευχαριστώ. Bien. Alors, Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Μιούλερ Φόλκαν, ο οποίος αντιπροσωπεύει την Ομοσπονδία τη Γερμανική Ομοσπονδία. Όχι, με συγχωρείτε, λάθο, λάθο τον Οργανισμό Απασχόλησης της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης Γερμανίας, της Βρυξέλλες. Και τον παρακαλώ να μην ακολουθήσει το παράδειγμα ε, του προλαλήσαντος, να είναι λίγο πιο λογικός να μιλήσει πέντε λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, μου ζήτησαν να παρουσιάσω ένα πρόγραμμα του Οργανισμού Απασχόλησης του Αρμόδιου Γερμανικού Υπουργείου, το οποίο έχουμε ετοιμάσει. Θα μπορούσα να μιλήσω για το Ταμείο Εγγύησης για τους Νέους, επειδή ο Οργανισμός Απασχόλησης είναι ένας θεσμός που, εφαρμόζει πολλά από αυτά τα μέτρα και όπως γνωρίζετε ίσως στη Γερμανία η κατάσταση είναι ευνοϊκή. Και ήδη έχουμε εφαρμόσει εγγύησεις για τους νέους αυτής της μορφής. Αυτό το πρόγραμμα λοιπόν ονομάζεται The Job of My Life, η απασχόληση της ζωής μου. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει τριετή διάρκεια, 2013-2016, με χρηματοδότηση 139 εκατομμυρίων ευρώ. Για να εξηγήσω καλύτερα αυτό το πρόγραμμα, πρέπει να σας προσιάσω ορισμένες βασικές υποθέσεις. Πρώτα απ' όλα, πιστεύουμε ε, στην εξισορροπημένη αγορά εργασίας στην Ευρώπη. Γι' αυτό είμαστε υπέρ της κινητικότητας και της κυκλικότητας. Ως επίσημος φορέας, όταν πρόκειται για κινητικότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, χρησιμοποιούμε το δίκτυο EURIS. Το βασικό στοιχείο αυτού του δικτύου είναι να υπάρχει συμφωνία μεταξύ των εταίρων δεν πρόκειται για ανεξάρτητες ε, πρωτοβουλίες όταν μιλάμε για διασυνοριακές δραστηριότητες. Αυτό αφορά και τα επαγγέλματα. Αν υπάρχει δηλαδή ένας υποψήφιος για ένα επάγγελμα, τον προσλαμβάνουμε. Αλλά επίσης αφορά και τις δραστηριότητες τις οποίες θέλουν να αναπτύξουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μία άλλη υπόθεση εργασίας, όπως λέμε, είναι η εξής. Πρέπει να υπάρχει πραγματική ανάγκη. Όχι πιθανή ανάγκη. Πρέπει να υπάρχει μια κενή θέση και ένας υποψήφιος ο οποίος είναι διαθέσιμος για να πληρώσει αυτή τη θέση. Δεν ξέρω πώς θα εκδηλωθεί η κατάσταση απασχόληση στην Ευρώπη. Θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο στοιχεία. Αφενός, δεν υπάρχει μόνο η περίπλοκη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, αλλά και είναι η περίπλοκη πρόσβαση στην κατάρτιση. Κυρίως όταν πρόκειται για συνεχιζόμενη εκπαίδευση. Επίσης, υπάρχουν και οι άνεργοι ε, για μεγάλο χρονικό διάστημα. Το πρόβλημα της κινητικότητας στην Ευρώπη δεν είναι πρόβλημα γνώσεων. Η κατάσταση ε, σήμερα μας δείχνει ότι οι γνώσεις υπάρχουν. Σε πολλές περιπτώσεις δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέτρα πρόθεσης ε, για ε, χώρες που προέρχονται από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά διαμένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφέρονται πολλοί παράγοντες και πολλές αιτίε που κατά την άποψή μας οδηγούν ε, στην κινητικότητα της εργασίας. Το πρόβλημα της επιμόρφωσης και της κατάρτασης των νέων ώστε να μπορέσουν να βρουν εργασία στη Γερμανία βασίζεται σε πολλά στοιχεία. Οι παράγοντες που ανέφερα συνεπάγονται ότι στη χώρα υποδοχής θα πληρούνται και ορισμένε προϋποθέσεις. Η κινητικότητα αρχίζει από τη χώρα προέλευσης, από τη, με βάση τη γλώσσα και τις γνώσεις. Και κατόπιν βλέπουμε ε, ποιες δυνατότητες απασχόλησης υπάρχουν. Ακόμα και αν μας δώσετε 8 λεπτά, ε, εγώ θα, ε, δεν θα προλάβω να καλύψω όλο μου το θέμα, θα τα βρείτε μέσα στα έγγραφα. Αυτές είναι δυνατότητες χρηματοδότησης για τους νέους. Βλέπετε λοιπόν ότι οργανώνονται μαθήματα γλωσσών στη Γερμανία, διότι αυτό είναι ένα από τα βασικά κριτήρια. Πρέπει κανείς να μπορεί να επικοινωνεί, να επικοινωνεί ε, με τους προμηθευτές, ε, με τους εργοδότες. Συνεπώς, πρέπει να υπάρχει μια βασική ε, γνώση της γερμανικής γλώσσας για να μπορούν οι νέοι να παρουσιαστούν σε μια συνέντευξη για να βρουν δουλειά. Υπάρχουν, αυτή είναι μία από τις δυσκολίες. Όλα αυτά τα αντιμετωπίζουμε στο πρόγραμμα και θα δείτε όλες τις δυνατότητες χρηματοδότησης των προγραμμάτων μέσα στο έγγραφο όπως σας έλεγα, αυτό καλύπτει και τη χώρα προέλευσης και όπως βλέπετε εδώ, την παρακολούθηση του ατόμου στη χώρα υποδοχής, συγκεκριμένα στη Γερμανία και κατόπιν ε, την παρακολούθηση του ατόμου αυτού στην επιχείρηση που έχει προσληφθεί. Το θέμα της κινητικότητας των νέων είναι κάτι το αδιαμφισβήτητο. Εδώ θα ήθελα να σας πω δύο λόγια και για τις προοπτικές που υπάρχουν στη χώρα αλλά και στις, στις ενδεχόμενες χώρες προέλευσης. Το βασικό πρόβλημα είναι πάντοτε το πρόβλημα του αποκλεισμού. Εάν υποδεχόμαστε άτομα ορισμένων ειδικοτήτων, Ε, μπορεί κανείς να απασχολήσει και άτομα τα οποία βρίσκονται σε μειονεκτική θέση στη χώρα τους. Εδώ υπάρχει φόβος ε, όσον αφορά τη χώρα προέλευσης. Δεν πρέπει να υπάρχουν αποκλεισμοί. Τώρα, για αυτό το πρόγραμμα θα ήθελα να σας αναφέρω τα δύο επιχειρήματα που βασίζονται στα ίδια κριτήρια. Όπως σας είπα, υπάρχουν 139 εκατομμύρια ευρώ που παρέχονται για αυτό το πρόγραμμα. Αν όμως διαιρέσουμε αυτό το ποσό με τα άτομα που θα φεληθούν, γνωρίζοντας ότι υπάρχουν εκατομμύρια νέων που είναι άνεργοι, ακόμα και αν αξιοποιήσουμε στο έπακρο αυτό το πρόγραμμα, με όλες τις πιθανές χρηματοδοτήσεις, αν μπορούσαμε να υποδεχθούμε όλους ε, τους ενδιαφερόμενους, Αυτό θα δημιουργούσε μια αιμορραγία εγκεφάλου, ένα brain drain στις ε, χώρες προέλευσης και δεν θα, θα μπορούσαμε να καλύψουμε όλες τις ανάγκες στη Γερμανία. Είναι ένα συνοδευτικό μέτρο, αλλά όχι ένα υποκατάστατο. Θα σταματώ εδώ αν έχετε ερωτήσει με στη θέση σας. Ευχαριστούμε. Το λόγο τώρα έχει ο κύριος Μασιμιλιάνο Μασκυρίνη. Μασκυρίνη διορθώνει πρόεδρος. Είστε διευθυντής ερευνών στο Eurofound και αν δεν κάνω λάθος έχετε δώσει ήδη κάποια έγγραφα στους συναδέλφους ενδεχομένως να τα παρουσιάσετε αυτά και στην προφορική σας παρουσίαση. Έχετε πέντε λεπτά σας λέω, τυπικά, αλλά από ό,τι φαντάζομαι θα μιλήσετε κι εσείς ε, οχτώ λεπτά. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Θα ήθελα να παρουσιάσω λίγο τα αποτελέσματα, τα πορίσματα της δημοσίευσης αυτής που έχετε μπροστά στα χέρια σας και θα μιλήσουμε λίγο για την εγγύηση των νέων ως μέσο καταπολέμησης ανεργίας. Βλέπετε πόσο δραματική είναι η εικόνα της ανεργίας των νέων στην Ευρώπη. Το 2011 η Ευρώπη είχε 14 εκατομμύρια νέους οι οποίοι βρίσκονταν εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης. Ουσιαστικά αυτό αντιστοιχεί στο 1 τρίτο του πληθυσμού των μικρών νοτίων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, το γεγονός ότι οι άνθρωποι αυτοί περνάνε πάρα πολύ χρόνο εκτός απασχόλησης έχει ένα τεράστιο κόστος για τον ίδιο τον άνθρωπο αυτόν αλλά και για την κοινωνία. Εμείς θεωρούμε ότι επικεντρωνόμενοι μόνο στα διαφυγόντα εισοδήματα και στους μη κατεβληθέντες φόρους, καταλήγουμε σε ένα ποσό κόστους για την Ευρώπη, το οποίο ξεπερνά τα 153 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή 1,2% του κοινοτικού ΑΕΠ. Βλέπετε λοιπόν ότι η κατάσταση δεν είναι βιώσιμη για την Ευρώπη. Τώρα τα κράτη-μέλη ενεργώς έχουν συμμετάσχει στην κατάρτιση διαφόρων μέτρων και στην ανάληψη πρωτοβουλειών προκειμένου να ενταχθούν οι νέοι στην αγορά εργασίας. Οι παρεμβάσεις αυτές γίνονται σε διάφορα επίπεδα τη πορεία ενό νέου από το σχολείο προ την αγορά εργασία. Υπάρχουν δηλαδή διάφορε πρωτοβουλίε προκειμένου να μειωθεί η ανεργία, προκειμένου να μεταβούν πιο μαλά οι νέοι προ την αγορά εργασία, να βελτιωθούν τα προσόντα και οι δεξιότητέ του και να καταρριφθούν οποιαδήποτε εμπόδια ενδεχομένω υφίστανται, προκειμένου να συμμετέχουν οι νέοι πιο ενεργά στην αγορά εργασία, ιδίω οι πιο ευάλωτοι νέοι. Ωστόσο, αυτό το οποίο βλέπουμε αξιολογώντα την αποτελεσματικότητα αυτών των ε, πρωτοβουλειών, αυτών των μέτρων, βλέπουμε τελικά ότι είναι πολύ δύσκολο να καταλήξουμε στην πιο επιτυχούσα προσέγγιση. Και αυτό το οποίο βλέπουμε τελικά είναι ότι χρειάζεται μια πιο επίσημη αξιολόγηση όλων αυτών των μέτρων υπέρ των νέων και κατά της ανεργίας. Εν γέννη πάντως μπορούμε να πούμε ότι οι περισσότεροι συμφωνούν με την προστιθέμενη αξία της ε, πρωτοβουλίας των νέων προκειμένου να ταχθούν οι νέοι στην αγορά εργασίας, ε, τις εγγύσεις για τους νέους. Και η εγγύηση για τους νέους βοηθά να αποφευχθούν οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις ανεργίας. Όσον αφορά τώρα την εγγύηση για τους νέους, θα ήθελα να αφαιρθώ σε κάποια παραδείγματα τα οποία θεωρούμε ότι είναι τα πιο αποτελεσματικά. Θα ήθελα να αφαιρθώ δηλαδή στη φιλανδική εγγύηση για τους νέους και ο Φιλανδός συνάδελφος φαντάζομαι ότι θα μιλήσει ακόμα περισσότερο για το ζήτημα αυτό. Η φιλανδική εγγύηση για τους νέους απαρτίζεται από δύο τμήματα. Πρώτον, έχουμε μία εξατομικευμένη προσέγγιση όπου καταρτίζεται ένα προσωπικό πρόγραμμα Εξέβρεση εργασία, υποστήριξη ενό νέου και στη συνέχεια έχουμε και την ίδια την εγγύηση όπου βάσει του εξατομικευμένου αυτού προγράμματο δίδεται μία προσφορά προ τον νέο. Αυτή η προσφορά μπορεί να είναι μία μαθητεία, ένα πρόγραμμα κατάρτισης ή μια μαθητεια ενα προγραμμα κατάρτιση η μια θεση εργασία. Το 2010 σύμφωνα με την αρμόδια αρχή αξιολόγηση τη Φιλανδία, η παρέμβαση αυτή κατάφερε να φτάσει σε περισσότερο από 80% των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα αυτό. Το βασικό πλεονέκτημα της εγγύησης για τους νέους έχει να κάνει με το ότι τελικά δίνει μια εξατομικευμένη υπηρεσία προς τους νέους προκειμένου να καταφέρουν να λάβουν πιο συνειδητές αποφάσεις για τη μετάβασή τους από το σχολείο στο χώρο εργασίας και βοηθά η εγγύηση αυτή για τους νέους να καταλάβουν ποιες είναι ενδεχομένω οι αδυναμίες τους και πώς μπορούν να αυξήσουν προσόντα και δεξιότητες για να συμμετέχουν καλύτερα στην αγορά εργασίας. Επίσης υπάρχει μια άμεση δράση προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ενεργεία των νέων προτού οριστικοποιηθεί, προτού παγιωθεί κατά κάποιο τρόπο η απομάκρυνση του νέου από την αγορά εργασία. Ουσιαστικά βλέπουμε ότι οι επιπτώσει είναι πολύ πιο επώδυνε όταν ένα νέο απέχει για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από την αγορά εργασία. Και δεν είναι τυχαίο ότι στη Φιλανδία, και ακολουθεί επίτε η Σουηδία, οι νέοι δεν μένουν για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα εκτό αγορά εργασία. Δηλαδή η ανεργία του είναι σύντομη από χρονική πλευρά. Επίση, μέσω τη εγγύηση αυτή για του νέου, ανοικοδομείται κατά κάποιο τρόπο μια εμπιστοσύνη, επανακτάται η εμπιστοσύνη των νέων προς τα θεσμικά όργανα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ενδεχομένω να είναι και πιο σημαντικό αυτό από το οικονομικό κόστο ανεργία. Θα πρέπει επίση να συνειδητοποιήσουμε ότι η στιγμή, η χρονική στιγμή τη παρέμβαση είναι πάρα πολύ σημαντική. Και η εγγύηση αυτή για του νέου ενδεχομένω να είναι πιο αποτελεσματική για αυτού που είναι έτοιμοι να εργαστούν. Πρέπει λοιπόν οι νέοι να ακολουθούν κάποιες λύσεις μακροπρόθεσμες και να μην επενδύουμε πάρα πολύ σε βραχυπρόθεσμες λύσεις, οι οποίες όμως δεν θα είναι βιώσιμες. Επίσης, οφείλουμε να συνειδητοποιήσουμε ότι η εγγύηση για τους νέους από μόνη της δεν μπορεί να επιλύσει τα διαρθρωτικά προβλήματα της προσχώρησης των νέων στην αγορά εργασίας. Ξέρετε ότι η ένταξη των νέων στην αγορά εργασία εξαρτάται και από πολλέ άλλε δημόσιε πολιτικέ, οι οποίε θα πρέπει ουσιαστικά να εγγυώνται στου νέου προγράμματα μαθητεία, κατάρτιση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό δηλαδή να συνειδητοποιήσουμε ότι θα πρέπει να υπάρχουν αυτές οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης. Απαιτείται η απαραίτητη δημόσια δομή προκειμένου να μπορεί να λειτουργήσει στην πράξη η εγγύηση για τους νέους. Η λειτουργία βέβαια της πρωτοβουλίας αυτής έχει να κάνει πάρα πολύ με την προετοιμασία των κρατών μελών από το επίπεδο ετοιμότητά τους, τους. Θα μπορούσαμε καταρχάς να αξιολογήσουμε την ετοιμότητα αυτή σε δύο σκέλη. Καταρχάς, αν έχουμε μία εξατομικευμένη προσέγγιση και δεύτερον, πώς υλοποιείται τελικά η εγγύηση αυτή. Θα πρέπει να δούμε αν υπάρχει μία δημόσια υπηρεσία για που θα μπορέσει να εφαρμόσει αυτή την εγγύηση για τους νέους και αν υπάρχει καλή συνεργασία ανάμεσα στη δημόσια αυτή υπηρεσία και τις υπόλοιπες δημόσιες υπηρεσίες. Αν πραγματικά θέλουμε να προσδώσουμε μια εξατομικευμένη λύση στους νέους, το κόστος ενδεχομένως για τη δημόσια αυτή υπηρεσία να είναι ιδιαίτερα υψηλό. Η Διεθνή Οργάνωση Εργασία έχει εκτιμήσει ότι η εφαρμογή τη εγγύηση για του νέου αντιστοιχεί περίπου σε 21 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο δικό μου οργανισμό, το Eurofound, θα αξιολογήσει την μεταβιβασιμότητα τη εγγύηση για του νέου σε διάφορες χώρες Ευρωπαϊκή Ένωση. Εν κατακλείδη, κυρίες και κύριοι, βλέπουμε ότι 153 δισεκατομμύρια ευρώ είναι το κόστος το οποίο θα πρέπει να καταβάλουμε αν δεν καταφέρουμε να εντάξουμε τα 14 αυτά εκατομμύρια νέου στην αγορά εργασίας. Τα 153 αυτά δισεκατομμύρια θα πρέπει να καταβληθούν τελικά ως κόστος, ω τίμημα. Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό να μάθουμε μένα από τους ΔΕ, να καταφέρουμε να διαχείουμε περισσότερο τις βέλτιστες πρακτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα πρέπει βέβαια αυτές να προσαρμοστούν έπειτα στο εθνικό πλαίσιο και θα πρέπει η εγγύηση για τους νέους να αποτελέσει μια μακροπρόθεσμη εγγύηση η οποία θα βλέπει πέρα από την καθαρά οικονομική διάσταση και θα είναι σαφώς μακροπρόθεσμη πρέπει να αναλάβουμε δράση επιγόντως. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ποιο είναι το τίμα το οποίο θα πρέπει να καταλάβουμε αν, αν, αν δεν αναλάβουμε δράση εγκαίρως. Δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο πλέον. Σας ευχαριστώ πολύ και με στη διαθεσή σας για τυχόν ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ. Περνάμε τώρα στον επόμενο μας καλεσμένο, στον κύριο Κίμο Ρουθ, που είναι σύμβουλος αγοράς εργασίας στο Υπουργείο Απασχόλησης και Οικονομίας της Φιλανδίας. Και μάλιστα είναι πολύ ενδιαφέρον αυτός ο συνδυασμός γιατί σπάνια έχουμε στο ίδιο Υπουργείο Χαρτοφυλάκια Απασχόλησης και Οικονομίας. Θα μας παρουσιάσει λοιπόν ο καλεσμένος μας τη λειτουργία του φιλανδικού συστήματος. Και μάλιστα είχαμε και την ε, Ευρωπαϊκή Κοινοβουλευτική εβδομάδα ένα από τα θέματα ήταν η απασχόληση στους νέους όπου μας έγινε μια παρουσίαση του φιλανδικού συστήματος ε, με αριστοργηματικό τρόπο. Πολύ επιτυχημένο σύστημα. Κύριε Κίμου, λοιπόν, Ρουθ, έχετε και εσείς το λόγο για 8 λεπτά. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως ακούσαμε, θα σας παρουσιάσω το φιλαδικό μοντέλο εγγύησης για τους νέους που άρχισε να εφαρμόζεται από την αρχή του έτους. Είχαμε κάποιες ε, στοιχειώδεις μορφές ε, του Ταμείου Εγγύησεων πριν από κάποια χρόνια είχαμε κάποια τέτοια ε, κάποιες απαρχές τέτοιου συστήματος, αλλά από φέτος, από την αρχή της χρονιάς, έχουμε ένα συνολικό μοντέλο εγγύησης για τους νέους από τη φιλανδική κυβέρνηση που τηρεί τις ε, κατευθυντήριες γραμμές του Συμβουλίου του Φεβρουαρίου. Θα ήθελα λοιπόν να σας παρουσιάσω τα βασικά στοιχεία του φιλανδικού μοντέλου για την εγγύηση των νέων. Πρώτα όμως να σας δώσω κάποια στοιχεία της κατάστασης ανεργίας στην Ελλάδα. Το ποσοστό ανεργίας των νέων ε, ανέρχεται στο 19% περίπου, δηλαδή λίγο κάτω από τον κοινοτικό μεσόρο, αλλά υψηλό αυτό το ποσοστό ανεργίας για τα φιλανδικά δεδομένα και δυστυχώς ε, αυξάνεται εξαιτίας της ε, ύφεσης από το 2011 και 2012. Πάντως το θετικό είναι ότι η περίοδοι ανεργίας είναι σχετικά βραχίες ε, στη Φιλανδία, ακόμη και για τους νέους. Λιγότερο από 20% των νέων ανέργων περνάνε περίπου τρεις μήνες σε ανεργία γιατί ακριβώ υπάρχουν πολλέ πολιτικέ επανένταξη των νέων στην αγορά εργασία. Τα γραφεία ανέβρεση εργασία ε, πρέπει να συντάσσουν τέτοιο ε, ένα, ένα σχέδιο για την ε, επαναπασχόληση των νέων μετά από δύο εβδομάδες από την έναρξη της περίοδου ανεργίας. Είναι πολύ σημαντικό, όπως σα είπα, αυτό το σχέδιο αγγίσης και βρίσκεται στο κυβερνητικό πρόγραμμα ήδη από το 2011. Θα ήθελα τώρα να δούμε τους στόχους ε, που είναι διτοί. Καταρχήν έχουμε τους νέους ανέργους ε, που τους ε, προσφέρουμε διάφορα στάζ ή διάφορα προγράμματα κατά τους πρώτους τρεις μήνες της ανεργίας τους και έχουμε και το δεύτερο στόχο που περιλαμβάνει εγγύηση της παιδείας. Δηλαδή στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε ε, ένα, μια θέση στην παιδεία όλων των αποφύτων ήδη από τον πρώτο χρόνο αποφύτησής τους. Επίσης ε, ε, έχουμε 60 εκατομμύρια ετησίως την πρικοδότηση αυτής της εγγύησης των νέων από τη φιλανδική κυβέρνηση. Είναι σημαντικά αυτά τα 60 ε, εκατομμύρια, είναι σχετικά μεγάλο ποσό δεδομένης της ε, οικονομικής στενότητας που πλήττει και τη Φιλανδία αυτή τη στιγμή. Επίσης έχουμε επιπλέον 52 εκατομμύρια κάθε χρόνο για το προσωρινό πρόγραμμα ε, για την δημιουργία ε, νέων επαγγελματικών προσόντων, ιδιαίτερα για τους νέους μεταξύ 20 και 29 που έμειναν εκτός του εκπαιδευτικού συστήματος ε, για μερικά χρόνια. Τι περιλαμβάνει η εγγύηση των νέων στη Φιλανδία. Περιλαμβάνει περισσότερες ευκαιρίες επαγγελματική κατάρτισης. Έχουμε αυξήσει τις θέσεις σπουδών κατά 2.000 θέσεις ε, φυσικά λαμβάνοντας υπόψη τις ε, ε, διαφορές της ηλικιακέ. Βέβαια, η Φιλανδία είναι σχετικά αεροκατοικημένη. Ο πληθυσμό συγκεντρώνεται κυρίως στις πόλεις. Επίσης, αλλάξαμε και το κριτήριο αποδοχής της γης. το κριτήριο επιλεξιμότητας δηλαδή για την συμμετοχή στο εκπαιδευτικό σύστημα. Δίνουμε προτεραιότητα στην ε, επιμόρφωση σε όσους ε, δεν έχουν, ε, προς, έχουν, δεν έχουν σπουδές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τώρα, αυξήσαμε το, την χρηματοοικονομική υποστήριξη των επιχειρηματιών. Αυξάνεται σε 800 ευρώ ανά μήνα, κάτι που δίνει έναυσμα στους επιχειρηματίες να προσλαμβάνουν στα σγέρα, σκουμένους στις επιχειρήσεις τους. Επίσης αυξήσαμε και της, ε, τον προϋπολογισμό του, της σχετικής υπηρεσίας. Έχουμε ε, πολύ, περισσότερες, ε, πολύ περισσότερους απασχολούμενους εκεί και επίσης έχουμε προβλέψει κονδύλια για τις μισθολογικές επιχορηγήσεις και την κατάρτιση των νέων. Βέβαια, οι πόροι αυτοί δεν αρκούν. Θα πρέπει ε, να προβλέψουμε και άλλες αλλαγές για να συνδυάσουμε τις, καλύτερα τις υπηρεσίες παιδείας, βρέσος ε, εργασίας ε, και, και την συμμετοχή των επιχειρήσεων. Αυξήσαμε την ευθύνη των τοπικών και περιφερειακών αρχών, ώστε και οι δήμοι και περιφέρειες να αναλαμβάνουν την ευθύνη ε, της καθοδήγησης και του επαγγελματικού προσανατολισμού των νέων μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Και μάλιστα η ευθύνη αυτή θα επεκταθεί ώστε ε, εκτός από τους Δήμους και τις περιφέρειες ε, και οι τοπικοί, τοπικά θεσμικά όργανα να αναλαμβάνουν σχετική ευθύνη. Έχουμε καλά αποτελέσματα σε ό,τι φορά το ειδικευμένο μοντέλο που έχουμε για τους νέους ε, που είναι αποκλεισμένοι, από, δεν ε, παρακολουθούν δηλαδή σπουδές ή δεν παρακολουθούν κανένα στάζ ή ε, πρόγραμμα επαγγελματική κατάρτισης. Και μάλιστα αυτό το σύστημα θα το γενικεύσουμε σε όλη τη χώρα για να βρούμε ποιοι νέοι αποκλείονται από την αγορά εργασίας και από την παιδεία, από το εκπαιδευτικό σύστημα. Και τέλος κύριε Πρόεδρε θα ήθελα να ε, επισημάνω ότι στο μοντέλο εγγύησεων της Φιλανδίας έχουμε επισημάνει την ανάγκη ενός συνολικού σφαιρικού μοντέλου και της ανάγκης συνδυασμού των διαφόρων πολιτικών. Το μοντέλο θα πρέπει να είναι περιεκτικό, ώστε και οι κοινωνικοί εταίροι και οι νέοι, αλλά και όλα τα στρώματα της ε, κοινωνίας να συμμετέχουν στον προγραμματισμό και την εφαρμογή των ε, στόχων του προγράμματος εγγύσεων για τους νέους. Και μάλιστα έχουμε και μια ομάδα εργασίας ε, που εξασφαλίζει το συντονισμό των δράσεων και την εφαρμογή της ε, εγγύησης για τους νέους με συμμετοχή διαφόρων ομάδων της κοινωνίας και μάλιστα έχουμε πολύ ενεργό συμμετοχή των ομάδων της κοινωνίας ε, στην αξιολόγηση, εφαρμογή και τον συντονισμό των δραστηριοτήτων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ερχόμαστε τώρα στο τελευταίο σημείο εξίσου σημαντικό, στους εκπροσώπους του Φόρουμ για τους νέους και δίνω το λόγο στον κύριο Πίτερ Μάτσεσεκ που είναι ο πρόεδρος του Φόρουμ. Ευχαριστώ. Ε, διακεκριμένοι, προσκεκλημένοι και ευρωβουλευτές. Είναι μεγάλη τιμή για μένα που εκπροσωπώ ε, το Φόρουμ, που είναι μια ανεξάρτητη πλατφόρμα των οργανώσεων των νέων στην Ευρώπη, που αντιπροσωπεύει ε, τα Συμβούλια Νεότητας και τις Διεθνείς Οργανώσεις Νέων. Θεωρούμε πολύ σημαντικό το ρόλο μας εργαζόμαστε στα θέματα της απασχόλησης των νέων και της, της ε, κοινωνικής ένταξης. Τα θεωρούμε θέματα προτεραιότητας από το 2008. Σε αυτές τις εποχές λιτότητας όπου οι οργανώσεις νέων είναι τα θύματα των περικοπών στους προπολογισμού, βλέπουμε ότι σήμερα περισσότερο από ποτέ οι νέοι χρειάζονται υποστήριξη επενδύσεις όχι μόνο για να υπάρχει η αξιοπρέπεια του ανθρώπου και να υπάρχει η αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών, αλλά και για την οικονομική και κοινωνική σταθερότητα της Ευρώπης. Θα ήθελα να αναφέρω στατιστικές που ανέφερε ο κ. Μασκερίνη και όλοι τις γνωρίζουν, δηλαδή 153 δισεκατομμύρια ευρώ είναι το κόστος της ανεργίας των νέων όσον αφορά ε, την απώλεια εισφορών, κοινωνικών εισφορών. Όπως είπα, το Φόρουμ των Νέων εργάζεται για τα θέματα τη ανεργία των νέων πολλά χρόνια και είναι απογοητευτικό να διαπιστώνουμε ότι ορισμένα κράτη-μέλη διστάζουν να επενδύουν σε αυτό το χώρο. Ακόμα και πριν από την κρίση, στι καλέ χρονιέ, ήταν ε, διπλάσια η ενεργεία των νέων σε σχέση με τον υπόλοιπο πληθυσμό. Γι' αυτό το Ευρωπαϊκό Φόρουμ χαιρετίζει το πακέτο μέτρων ε, για την επίλυση αυτών των θεμάτων, ώστε οι νέοι ε, να έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα απασχόλησης κυρίως ε, τις προσπάθειες να αντιμετωπιστούν ορισμένα προβλήματα που αντιμετωπίζονται, όπως η ανάγκη βελτίωσης πρόσβασης των νέων στην ε, αγορά εργασίας, ε, την εγγύσια τους νέους και την ομαλή μετάβαση από την εκπαίδευση στην εργανία, κυρίως σε μαθητείες και σε καλύτερη κινητικότητα εργασίας στην Ευρώπη. Οι προτάσεις, προτάσεις από το Συμβούλιο ήταν μια πολύ καλή εξέλιξη και το φόρουμ μας εκτιμά ιδιαίτερως την ευκαιρία που δόθηκε να, για να γίνουν προτάσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Ο τόνος είναι φιλόδοξος. Αναγνωρίζει τη διάσωση σχέση των νέων, τους περιορισμένους οικονομικούς τους πόρους, τις επισφαλείς συνθήκες εργασίας και την περιορισμένη κοινωνική προστασία. Το έγγραφο αναγνωρίζει επίσης ότι οι νέοι έχουν μεγάλες πιθανότητες να αντιμετωπίσουν διακρίσεις στην αγορά εργασίας. Όλα αυτά είναι αιτήματα τα οποία επαναλαμβάνουμε πολλά χρόνια και με τα χαράς βλέπουμε ότι αυτό το γεγονός ε, ε, έχει αναγνωριστεί. Η προσέγγιση της Επιτροπής επίσης άλλαξε ε, σημαντικά τα τελευταία χρόνια και αντικατοπτρίζει τη σοβαρότητα της κατάστασης. Αυτό είναι κάτι το οποίο χαιρετίζουμε. Αναγνωρίζει τη σημασία των υπηρεσιών για τους νέους και των οργανώσεων νέων και αναφέρει ότι θα πρέπει να συμμετέχουν σε όλα τα επίπεδα ε, στην ε, κατάσταση και εφαρμογή των προγραμμάτων για τους νέους. Αυτό το μοντέλο ε, συμμετοχής των πάντων είναι ένα μοντέλο το οποίο θα ακολουθήσουν και τα άλλα κράτη-μέλη. Η σύσταση για την εγγύηση των νέων επίσης καλεί σε συμμετοχή των εκπροσώπων των νέων και των ρόζων των νέων ένα αίτημα το οποίο προωθούμε εδώ και χρόνια, κάτι το οποίο έχει ακουστεί σε αυτό τον οίκο της Δημοκρατίας. Επίσης ζητεί την επικύρωση της επίσημης παιδείας, την αναγνώριση των ικανοτήτων που απαιτούν της συνεργασία. Ε, την ποιοτική εργασία τους νέους και χρησιμοποιεί ε, ε, τον όρο, ορίζει τι είναι το Ταμείο Εγγύης για τον νέο. Επίσης, αναγνωρίζει το γεγονό ότι τα άτομα κάτω των 25 πρέπει να καλύπτουν αυτά τα θέματα, διότι μπορεί, θα, μπορεί να βοηθήσει τους νέους. Ωστόσο, θα πρέπει να πούμε ότι είμαστε απογοητευμένοι από την, τα αποθεματικά των 6 δισεκατομμύρων στο πολιτέ πλαίσιο. Η Παγκόσμια Οργάνωση εργασία έχει συστήσει πολύ περισσότερα δισεκατομμύρια και σημαντικές επενδύσεις για να μπορεί να διατηρηθεί. Αν λάβουμε υπόψη ότι 8,4 δισεκατομμύρια δαπανώνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την κατάρτιση, το το ποσό το οποίο τίθεται για τους νέους είναι σταγόνα το ωκεανό. Δεν θα πρέπει απλώς να επαναλαμβάνονται τα μέτρα που υπάρχουν για να κατανέμονται, αλλά θα πρέπει να γίνουν σημαντικές επενδύσεις και να γίνει μια αναδιοργάνωση των μέτρων ώστε να υπάρχουν υπηρεσίες για τους νέους, τα μέτρα τους και ότι ο κάθε νέος στην Ευρώπη θα μπορεί να βρει μια σωστή δουλειά ή τη δυνατότητα κατάρτισης η εργασία σε επιχειρήσεις. Είμαι ευτυχής που άκουσα ότι μιλήσατε για ποιοτική μαθητεία και ποιοτική κατάρτιση. Αυτό είναι κάτι το οποίο μας αγγίζει, ε, επειδή πρέπει να υπάρχει ένας δομημένος διάλογος. Και πρόσφατα είχαμε μια διάσκεψη για τους νέους και άτομα που λαμβάνουν αποφάσεις ε, στο Δουβλίνο και επανελήφθη ε, επανελήφθη η πλευρά, η ποιοτική πλευρά, να αντιμετωπίζουν δηλαδή ισότιμα στην αγορά εργασία και να μην υπάρχει διάκριση με βάση την ηλικία. Αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο το οποίο είναι σημαντικό ε, και αναγνωρίζεται από τους νέους. Γιατί επειδή οι είναι ρεαλιστικοί, δεν ζητούν κάτι το οποίο δεν είχαν οι γονείς τους ε, θέλουν πραγματικές επενδύσεις και προστασία των δικαιωμάτων τους για εργασία αυτή, αυτό δεν είναι ένα όραμα για το μέλλον της Ευρώπης. Κάτι το οποίο ζητείτε, απαιτείται για να εξασφαλιστεί η σταθερότητα η οικονομική και η κοινωνική της Υπήρου μας. Θα ήθελα να πω και πάλι ευχαριστώ για την ευκαιρία που μας δώσατε να μιλήσουμε εξ ονόματος του Φόρουμ των Νέων και τους νέους που εκπροσωπούμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Χαίρομαι πραγματικά που οι νέοι τελικά είναι αυτοί που δείχνουν πώς μπορούμε να χειριστούμε το χρόνο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δύο λεπτά θα έχουν οι επόμενοι ομιλητές. Όλε Κρίστενσεν και Κλίβικ στη συνέχεια. Όλε Κρίστενσεν στην αρχή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συμμετέχοντες για τις παρουσιάσεις που κάνανε. Όντως το ζήτημα της ενεργείας των νέων είναι μια πρόκληση την οποία θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε και στο μέλλον και πραγματικά οι νέοι πρέπει να είναι σε θέση να ξυπνάνε το πρωί και να πηγαίνουν σε μια δουλειά. είναι πάρα πολύ σημαντική η εργασία και συνδέεται πολύ και με την αξιοπρεπή ζωή. Απευθυνόμενο τώρα στη Eurofound, θα ήθελα να πω το εξή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνδυάσουμε τα γίνονται βραχυπρόθεσμα με αυτά που γίνονται μακροπρόθεσμα. Πώ μπορούμε να συνδυάσουμε λοιπόν την εγγύηση για του νέου με κάποιε μακροπρόθεσμε προσπάθειε, με κάποια μέτρα δηλαδή, τα οποία θα είχαν ω στόχο να μεταρρυθμιστούν κάποιε δομέ εθνικέ. Ποιε προσπάθειε πρέπει να καταβληθούν, τι μέτρα μπορούμε να εγκρίνουμε για να γίνει κάτι τέτοιο. Και μια ερώτηση προ όλο το πάνελ. Οι νέοι αποτελούν πολλές φορές θύμα, θύματα μιας πάρα πολύ βάναυσης, ενός πολύ βάναυσου ανταγωνισμού σε σχέση με πιο ηλικιωμένου εργαζομένους. Τι ρόλο μπορούν να δραματίσουν οι μικρομεσαίε επιχειρήσει, προκειμένου οι νέοι να καταφέρουν να έχουν ε, μια καλύτερη τύχη στην αγορά εργασία, τι κίνητρα μπορούμε να δώσουμε στι μικρομεσαίε επιχειρήσει προκειμένου να προσλαμβάνουν περισσότερου νέου. Επίση, το Συμβούλιο τελικά συνειδητοποίησε εν τέλει ότι θα πρέπει να λάβει υπόψη του το ζήτημα τη ανεργία των νέων. Πώ μπορούμε λοιπόν να εγκρίνουμε συγκεκριμένα κοινοτικά μέτρα στα πλαίσια τη κοινωνική διάσταση για να καταπολεμήσουμε την ανεργία των νέων. Αναφερόμαστε συνεχώ στην περίφημη Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Θα πρέπει πραγματικά να καταδείξουμε ότι μα απασχολεί το ζήτημα αυτό και θέλουμε να δώσουμε μια απάντηση στο σημαντικό του αυτό πρόβλημα. Ευχαριστώ. Η κυρία Κρύβετη. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Μολονότι είναι η εβδομάδα της, α, ε, της θα μιλήσω την ε, γλώσσα μου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω Θα να ευχαριστήσω όλους τους ε, συμμετέχοντες για όλες αυτές τις πάρα πολύ ενδιαφέρουσες ε, παρουσιάσεις. Όλους ιδιαίτερως με ενδιαφέρει η περίπτωση των νέων γυναικών, οι οποίες όπως βλέπουμε είναι οι πρώτες οι οποίες πλήττονται από την ανεργία των νέων. Μολονότι οι περισσότερες εξ αυτών έχουν διπλώματα πανεπιστημιακά και μάλιστα πολύ περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν. Δυστυχώς όμως ο ανταγωνισμός που ασκείται εκ μέρου των συνομήλικών του αντρών είναι πάρα πολύ έντονος, με αποτέλεσμα γυναίκες αυτές τελικά να πλήττονται όλο και περισσότερο από την ανεργία. και στη συνέχεια βέβαια κατηγορούμε και τις γυναίκες αυτές για τις πτωτικές στάσεις στην γεννητικότητα στην Ευρώπη. Θα ήθελα λοιπόν εγώ να μιλήσω περισσότερο για τις νέες αυτές γυναίκες. Θα μπορούσαν να μου πούν οι συμμετέχοντες στην ακρόαση αν έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να βοηθηθούν οι γυναίκες αυτές, προκειμένου να μπορέσουν να ταχθούν περισσότερο στην αγορά εργασίας. Θα μπορούσατε να μου πείτε επίσης πώς ε, θα μπορούσαν να δημιουργηθούν ισότιμες συνθήκες στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. Γιατί ξέρουμε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν ορισμένα κράτη-μέλη τα οποία έχουν ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενταθούν τα μέτρα κινητικότητας των νέων στον τομέα της εργασίας όμως, όχι μόνο της εκπαίδευσης. Προς αυτό τι έχει να μας πείτε κυρία Μπλίνκεβιτσούτε και μετά κυρία Μωρά Σαχτιέ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους καλεσμένους εμπειρογνώμονες και να συμφωνήσω πρώτα απ' όλα με τον εκπρόσωπο του Youth Forum. Φυσικά τα 6-7 δισεκατομμύρια που πρόλευσαν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων για το Ταμείο Εγγυήσεων για τους νέους είναι ένα πενιχρό ποσό. Γνωρίζουμε ότι οι ζημίες μας ανέρχονται σε 153 δισεκατομμύρια το χρόνο εξαιτίας της ενεργείας των νέων. Αν αυτό το διαιρέσουμε σε 27 χώρες, βλέπουμε τι απόλυση έχει κάθε χώρο, χώρα από τη μάστιγα αυτή. Βέβαια θα πρέπει να μείνουμε ενωμένοι και να ελπίζουμε σε αίσιες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Και ευελπιστώ ότι το ποσό αυτό τελικά θα αυξηθεί. Όσοι είναι ανειδίκευτοι, δεν έχουν δουλειά ή δεν είναι ιδιαίτερα καταρτισμένοι, αντιμετωπίσουν πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα να βρουν ε, δουλειά. Αλλά δυστυχώς ακόμη και όσοι είναι ε, απόφοιτοι της εκπαίδευσης, είναι υπερειδικευμένοι, ακόμη και αυτοί αντιμετωπίζουν πρόβλημα στο να βρουν μια θέση απασχόλησης. Και ρωτώ τον καθηγητή από την Κρακοβία. Θα, πρέπει να καταρτίζουμε το, τους νέους μας ώστε να λαμβάνουν τα εφόδια και τα προσόντα που απαιτεί η αγορά εργασία. Έχουμε ένα κατάλληλο μηχανισμό για να προβλέπουμε και τι μελλοντικέ ανάγκες αγορά εργασία ή μήπω θα συνεχίσουμε αυτό που κάναμε μέχρι τώρα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και με ενδιαφέρει η γνώμη σας κύριε καθηγητά για το τι θα έπρεπε να κάνουν και τα κρατημέλη αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να εξισορροπήσουμε το σκέλος της ίτησης με το σκέλος της προσφοράς την προσφορά δηλαδή της ε, παιδείας και τη ζήτηση της αγοράς εργασίας. Σίγουρα οι νέοι είναι το πιο ευκίνητο τμήμα του πληθυσμού και ε, διαπιστώνουμε κίνδυνο σε πολλές χώρες όπως και στην πατρίδα μου, τη Λιθουανία, για αφέμαξη εγκεφάλου. Ένας νέος, ε, ιδιαίτερα αν καταγεται από επαρχία, πολύ πιο εύκολα αφήνει την επαρχία του και πηγαίνει σε μεγάλη πόλη με αποτέλεσμα να περιμόνεται η ύπεθρος και όταν ο νέος αυτός δεν βρίσκει καν δουλειά στην πρωτεύουσα σε μια μεγάλη πόλη, αναγκάζεται σε μετανάστευση. Πηγαίνει στη Γερμανία ή σε άλλες χώρες και αν δεν βρει και εκεί δουλειά, τότε μπορεί να φύγει και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ όλους τους ε, όσους παρενέβησαν ε, μίλησαν πολλά διδάγματα. Τέσσερα ερωτήματα θέλω να θέσω. Πρώτα απ' όλα, μας είπατε πόσο κόστιζε η, η μη πράξη ε, σε δισεκατομμύρια σε όσους νέους δεν έχουν προσόντα. Μπορείτε να προσεγγίσετε τον αριθμό των νέων που δεν έχουν προσόντα ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο με το ποσοστό σε επίπεδο Φιλανδίας. Δεύτερη ερώτηση. η εγγύσια για τους νέους. Λειτουργεί με την επανεκπαίδευση σε τέσσερις μήνες. Για τους νέους που δεν έχουν προσόντα, βλέπουμε ότι σύμφωνα με την εμπειρία μας η επανεκπαίδευση δεν είναι ο, πιο, ο πρώτος και ο πιο σημαντικός κρίκος, διότι εκείνοι που δεν έχουν προσόντα ε, βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση με τα προγράμματα κατάρτισης. Δεν μπόρεσαν να ενταχθούν στο σύστημα, δεν κατόρθωσαν, το σύστημα επίσης δεν ξέρετε πώς να τους απορροφήσει. Όταν λοιπόν στη Φιλανδία ε, λαμβάνονται μέτρα κατά περίπτωση, θα πρέπει να μας πείτε πώς προετοιμάζετε τους νέους ε, να γίνουν πιο υπεύθυνοι όταν δεν έχουν προσόντα, προκειμένου να ενταχθούν καλύτερα. Το τρίτο, είπατε ότι πρέπει να αγγίξουμε εκείνους που βρίσκονται στο περιθώριο, που έχουν αποκλειστεί. Το ερώτημά μου είναι πώς θα το κατορθώσετε, πού θα τους βρείτε, ε, στις ε, φτωχές περιοχές, στα κοινωνικά κέντρα. Αυτό είναι δύσκολο. Ποιο είναι το σύστημα που εφαρμόζετε για να τους προσεγγίσετε. Το τελευταίο ερώτημα έχει σχέση με παρατηρήσεις που έγιναν, αλλά ένα βήμα πιο πέρα. Σήμερα με την κρίση βλέπουμε ότι οι νέες γυναίκες έχουν μεγαλύτερη δυσκολία να βρουν δουλειά παρά οι νέοι, παρά το γεγονός ότι αυτές μπορεί να έχουν καλύτερη κατάρτιση. Στα παραδείγματα της Φιλανδίας και εσείς βλέπετε αυτό το ίδιο φαινόμενο, δηλαδή ότι οι γυναίκες, οι νέες κοπέλες βρίσκουν πιο δύσκολα δουλειά. Σόγκορ, και μετά κύριε Αντζελίλη, ο Τζάμπα Σόκολ. Ευχαριστώ. Κάποιος μίλησε για τα ε, μεγάλα εμβληματικά προγράμματα της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς ε, στις πατρίδες μας έχουμε εμπειρία και από κάποια μικρή εμβέλειες προγράμματα για, τις, για την ηθική επιχειρηματικότητα, γιατί υπάρχουν τεράστια προβλήματα στις τοπικές και περιφερειακές διοικήσεις να τους πείσουμε να βρουν εθελοντέ. Και είχαμε και καλές, αλλά δυστυχώς και κακέ εμπειρίες τα τελευταία χρόνια από το πώς οι κυβερνήσεις ε, ή τα Υπουργεία ε, είναι κατά του εθελοντικού έργου των μη κυβερνητικών ε, οργανώσεων. Και εγώ είμαι υπέρ των μεγαλεπίβολων κοινωτικών προγραμμάτων, αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνούμε και το έργο μικρής εμβέλειας μικρών κυβερνητικών ΜΚΟ που προσπαθούν να εκπαιδεύσουν και να καταρτήσουν τους νέους μεταξύ 14 και 18 ετών. Και το έργο τους είναι πολύτιμο κατά τη γνώμη μας. Η κυρία Αντζελίλη και μετά ο κύριος Σέρκας. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω την Πρόεδρο η οποία διοργάνωσε αυτή την ακρόαση και όλους ιδιαιτέρως θα ήθελα να ευχαριστήσω τους προσκεκλημένους μας. Ένα αίτημα θα ήθελα να υποβάλω προς τους προσκεκλημένους μας. Θα ήταν δυνατόν να μας δώσετε όλα αυτά τα έγγραφα τα οποία παρουσιάσατε και ενδεχομένω ακόμα και τα δεδομένα τα οποία παρουσιάσατε Όλος σε αυτό το που με ενδιαφέρει είναι να γνωρίζω το γερμανικό σύστημα κατάρτισης που από όσο γνωρίζω ναι, μου λένε ότι είναι διαθέσιμα τα έγγραφα, εγώ ένα μόνο είχα λάβει. Πάντως μου λένε ότι το γερμανικό αυτό σύστημα κατάρτισης έχει ουσιαστικά καταλήξει σε πολύ θετικά αποτελέσματα. Μου είναι χρήσιμες όλες αυτές οι πληροφορίες γιατί είμαι η εισηγήτρια για μία γνωμοδότηση όσον αφορά την ανεργία των νέων για την Επιτροπή Γυναικών στην οποία συμμετέχω και επομένω από αυτή την οπτική γωνία θα πρέπει να τονίσουμε ακόμα περισσότερο το ότι ανάμεσα στους άνεργους νέους είναι οι νέες γυναίκες αυτές οι οποίες ε, αντιστοιχούν στο μεγαλύτερο ποσοστό. Επομένως ε, η ανεργία των νέων πλήγει περισσότερο τις νέες γυναίκες από ότι τους νέους άνδρες. Συνεπώς πιστεύω ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε συγκεκριμένα με το ζήτημα αυτό, να μιλήσουμε συγκεκριμένα για το ζήτημα αυτό, λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι στην πραγματικότητα το 60% των νέων πτυχιούχων είναι γυναίκες. Στην πραγματικότητα λοιπόν βλέπουμε ότι είναι οι γυναίκες αυτές οι οποίες πολύ πιο γρήγορα φτάνουν στο πτυχίο, με καλύτερους μάλιστα βαθμούς, αλλά παράλληλα είναι και το τμήμα αυτό του πληθυσμού το οποίο πλήττεται περισσότερο από την ενεργία. Μολονότι ουσιαστικά είναι ένα τμήμα του πληθυσμού το οποίο αξίζει περισσότερο, έχει περισσότερες δεξιότητες. Σας ευχαριστώ. Merci. Ευχαριστώ. Ο Αλεξάνδρ Αλεχάνδρος Σέρκας και μετά η κυρία Γεζοβιέτσκα. Ευχαριστώ. Και για μένα και για τους καλεσμένους είναι προφανές ότι μια τέτοια επιδημία θα έλεγα και ένα τόσο διαρθρωτικό πρόβλημα πολύ δύσκολα θα επιληθεί με κάποια εμβαλωματικά μέτρα ε, με κάποια ημίμετρα ή με κάποια μέτρα που έχουν σε επικοινωνιακό χαρακτήρα. Έχαμε 3 ή λίγα παραπάνω δισεκατομμύρια ευρώ στην πρωτοβουλία για, τον, για τους νέους, αλλά θέλουμε να αξιοποιήσουμε τις βέλτιστες πρακτικές. Θα υποβάλω τρεις ερωτήσεις λοιπόν προς τους καλεσμένους μας, προς εμπειρογνώμενους που ίσως ε, είναι χρήσιμες για τις χώρες ιδιαίτερα που, ε, που έχουν, για τις χώρες που έχουν χτυπηθεί από τη μάστιγα της υψηλής ανεργίας των νέων. θα ήθελα να, πω, να ρωτήσω ε, των εμπειρογνώμων από τη Φιλανδία. Σίγουρα η εξειδίκευση, η εξατομίκευση στα προβλήματα αυτά είναι πολύ σημαντική. Ποια είναι η αναλογία μεταξύ των ανέργων νέων στην Φιλανδία και του προσωπικού που ε, ασχολούνται με τον ειδικό επαγγελματικό προσανατολισμό αυτών των νέων. Σε ό,τι αφορά τον εκπρόσωπο του Φόρουμ για την Νεολαία. Ε, μετά την ανάλυση των εμπειριών της Σουηδίας και της Φιλανδίας ε, που έχουν συγκεκριμένη εμπειρία ε, και δεν ξέρω αν θα μπορούσε το ίδιο το μοντέλο άθικτο να μεταφερθεί στις χώρες του Νότου που έχουν διαφορετικές ανάγκες, να μας πει πώς πιστεύετε ότι μπορούμε αυτό το μοντέλο να το μεταλαμπαδεύσουμε στις χώρες του Νότου, δεδομένων των ιδιαιτεροτήτων που έχουν οι χώρες του Νότου. Γιατί ξέρουμε ότι άλλα προβλήματα έχει η Φιλανδία και άλλα η Ισπανία ή η Ιταλία. Αλλά ποιε είναι οι προτάσει για μια τέτοια δεχόμενη προσαρμογή του σκανδιναβικού μοντέλου προ τον Νότο. Το θέμα τη Γερμανία. Πώ θα προσεγγίσουμε το νέο μοντέλο τη κινηματική της κινητικότητας. Στη Γερμανία έχουμε νέους ε, ε, από την ε, Ισπανία και είχαμε σοβαρότατες ανησυχίες και πολύ ανησυχητικά σχόλια και, παρατη... και πληροφορίες ανθρώπων στη Γερμανία που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν αυτή την ε, δύσκολη στιγμή που αντιμετωπίζουν και την ανάγκη που έχουν οι νέοι από τις χώρες μας να βρουν εργασία. Και ουσιαστικά ε, κάνουν ένα dumping κοινωνικό και εφαρμόζουν ε, low cost ουσιαστικά, να ζητούν low cost, χαμηλού κόστους εργατικό δυναμικό. Οπότε δεν θα πρέπει να ξεχνούμε την μεγάλη ανέχεια που επικρατεί στις χώρες αυτές. Γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αντιμετωπίσει τις χώρες του Νότου οι άνεργοι αυτοί έχουν προβλήματα και δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να υπόκειται επιπλέον σε διακριτική μεταχείριση ή σε κακομεταχείριση από χώρε ε, και ε, άτεκτου επιχειρηματίε που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τη δύσκολη κατάστασή του. Η κυρία Γιαζοβιέσκα, ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να αναφερθώ στο πρόγραμμα αυτό για το Ταμείο των ε, Νέων της Φιλανδίας. Είπατε ότι εφαρμόζεται ένα εξατομικευμένο μοντέλο για κάθε νέο. Πόσους λοιπόν συμβούλους έχετε προσλάβει, πόσους συμβούλους έχετε που ασχολούνται με αυτόν τον επαγγελματικό προσανατολισμό και πώς ετοιμάζονται αυτοί οι σύμβουλοι και πώς σχεδιάζουν αυτά τα ατομικά προγράμματα για τον κάθε μεμονωμένο νέο, γιατί μιλήσατε για εξατομικευμένα προγράμματα επαγγελματικού προσανατολισμού. Επίσης, αναλύσατε την δομή των δαπανών. Ε, ποιες δραστηριότητες απορροφούν περισσότερα κονδύλια και στις, ε, στα εκπαιδευτικά προγράμματα που προτείνεται ή στις καταρτήσεις που προτείνεται. Ε, οι περισσότερες σπουδέ έχουν οικονομικό χαρακτήρα. Ποιο είναι το κεντρικό στοιχείο αυτών των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που προτείνεται. Ε, είπαμε ότι το όλο πρόγραμμα προβλέπει χρηματισμό πάνω από 150 δισεκατομμύρια. Έχουμε μόνο 8 δισεκατομμύρια στο Ταμείο Εγγύσεων για τους νέους. Αυτή η τεράστια διαφορά θα μας οδηγήσει σε ένα περιορισμό ουσιαστικά των δικαιούχων αυτού του προγράμματος ή μήπως θα υποβαθμίσει την ποιότητα γιατί ο καθηγητής από την Πολωνία μίλησε για την ανάγκη της ποιότητας και σίγουρα εν μέσω της κρίσης η ποιότητα αυτού του προγράμματος θα αποτελέσει συνταγή της επιτυχίας του. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ για τις εκπροσωπήσεις που είχατε εδώ. Είχα το ίδιο ερώτημα κι εγώ. Αυτές οι εγγύσεις για τους νέους είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Αυτό που απασχολεί είναι ότι ανεβάζουμε πολύ τις ελπίδες των νέων διότι η υλοποίηση αυτών των εγγύσεων των νέων εξαρτάται από τα κράτη-μέλη. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Ποιες είναι οι βασικές προϋποθέσεις για να μπορούν να λειτουργούν σωστά οι εγγύσει για τους νέους στα κράτη-μέλη. Διότι γνωρίζουμε πώς, πόσο ποικίλουν τα εκπαιδευτικά και κοινωνικά συστήματα στην Ευρώπη. Ποιες είναι οι βασικές προϋποθέσεις ώστε αυτές οι εγγύσεις των νέων να λειτουργούν σωστά. Διαφορετικά, απλώς και μόνο, επαναλαμβάνουμε συνέχεια το ίδιο θέμα. Δηλαδή ότι οι εγγύσεις των νέων κατά κάποιο τρόπο θα λειτουργήσουν θαυματουργά ε, στις ε, αγορές εργασίας των κρατών μελών. Ελπίζω να μην δίνουμε φρούδες ελπίδες στους νέους, όπως ε, είπε εδώ εκπρόσωπος του φόρουμ, ότι έχουν λογικές ελπίδες. Ελπίζω λοιπόν ότι και εμείς θα δίνουμε λογικές απαντήσεις στα προβλήματά τους. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να κάνω ένα ερώτημα στον κύριο Μούλερ, επειδή εξεπλάγει από τον αριθμό των προγραμμάτων που ονομάζονται The Job of My Life, η δουλειά της ζωής μου. Θα πρέπει ίσως να διδάξουμε στους νέους ότι δεν θα έχουν μία δουλειά στη ζωή τους, θα έχουν πολλές δουλειές ε, στη ζωή τους. Ίσως είναι κάτι το οποίο δεν κατάλαβα. Ένα άλλο ερώτημα. Ε, δεν είσαστε εσείς που θα μου απαντήσετε, αλλά εξεπλάγει από την παρουσίαση του προγράμματός σας. Και εσείς προδικάσατε την ιδέα ότι ίσως υπάρχει ένας φόβος, ένας κίνδυνος brain drain. Μία από τι προκλήσει για την Ευρωπαϊκή Ένωση, πιστεύω, είναι να αντιμετωπίσει το θέμα τη κινητικότητα με εκβάθρον διαφορετικό τρόπο από ό,τι έχει κάνει μέχρι σήμερα. Η κινητικότητα ήταν το α και το ω τη συνθήκη τη Ρώμη, πρώτα απ' όλα για τα κεφάλαια, τα οποία υποφελήθηκαν πολύ, το λιγότερο, κατόπιν για τα αγαθά και τι υπηρεσίες, αλλά και για τα άτομα. Βλέπουμε όμω ότι με την κρίση το θέμα τη κινητικότητα των ατόμων τίθεται με διαφορετικό τρόπο. Και υπάρχει ένας κίνδυνος ότι τελικά η κινητικότητα όπως τη βλέπουμε σήμερα ε, φτάνει σε ένα ε, θέμα αντίφασης με την ε, αναγκαστική εργασία, με συγχωρείτε έτσι θα το πω, αλλά ένα οικονομικό μοντέλο που βασίζεται σε μια έξοδο από την κρίση, χάρη σε μια κινητικότητα από οποιασδήποτε προϋποθέσεις. Και οθεί τους πληθυσμούς της περιφέρειας να δουλέψουν στο κέντρο αφού εκπαιδεύτηκαν με χρήματα του κέντρου ε, για να εργαστούν στο κέντρο και μετά να πάρουν σύνταξη στην περιφέρεια είναι ένα μη βιώσιμο μοντέλο. Και αναρωτιέμαι πώς μπορούμε αυτό να ε, το υλοποιήσουμε τη στιγμή που μιλάμε για εγγύηση νέων, γιατί μεταξύ των κινουμένων εκείνοι που μετακινούνται περισσότερο είναι οι νέοι. Αν θέλουμε λοιπόν να αποκαταστήσουμε τις μακροοικονομικές αδικίες, αν θέλουμε να αποκαταστήσουμε ε, τη ζωή, ε, πρέπει να, τα δούμε διαφορετικά τα πράγματα. Στην Λιθουανία ή στην Λετωνία ε, το Διεθνές τα Ταμείο λέει ότι λύνει τα βασικά προβλήματα, αλλά λύνει προβλήματα ε, διώχνοντας τους νέους από τις χώρες τους. Να μην υπενθυμίσουμε τι έλεγε ο Λένιν, έλεγε ότι οι άνθρωποι που έφευγαν ήταν εκείνοι που ψήφιζαν με τα πόδια τους. Δεν είναι αυτό που θέλουμε σήμερα. Πρέπει αυτή η εγγύηση των νέων να είναι ένας τρόπος για να διατηρήσει κανείς τους νέους για να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες οι χώρες που έχουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες. Αυτά που λέω είναι γενικότητες, το ξέρω, αλλά μερικές φορές θέλω να τα υπενθυμίζω, να γνωρίζουμε το πλαίσιο το οποίο κινούμεθα. Δίνω πάλι το λόγο στην εισηγήτρια για δύο λεπτά και μετά όλοι ε, θα μπορέσετε να δευτερολογήσετε, αλλά πολύ σύντομα. Η κυρία Στριβλέσκα. Ευχαριστώ. Όπως και οι προλαλήσαντες, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους ε, καλεσμένους μας για τις πολύ ενδιαφέρουσες ε, συναρπαστικές θα έλεγα παρουσιάσεις τους που συνέβαλαν προς, τον, προς την κοινή διαπίστωση συνέκλεια μάλλον προς την κοινή διαπίστωση ότι θα πρέπει να είναι πολυδιάστατη αντιμετώπιση του προβλήματος ενέργειας των νέων. Και φυσικά τα κράτη-μέλη αναλαμβάνουν ένα μεγάλο τμήμα της ευθύνης και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να δουν τι μπορούν να προτείνουν και να προσφέρουν στους νέους. Και μάλιστα το φιλανδικό μοντέλο που μας παρουσιάστηκε είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση που θα πρέπει να αξιοποιήσουν και οι υπόλοιπε χώρες μέλη και να το προσαρμόσουν στη δική τους πραγματικότητα. Θα ήθελα να αναφερθώ σε κάτι που είπε ο καθηγητής Γκούρνιακ. Ε, είπατε ε, κύριε καθηγητά, ότι αυτό που προέχει πάνω απ' όλα είναι η ποιότητα της παιδείας και η ποιότητα της προετοιμασίας ε, των νέων για να εισέλθουν στην ε, αγορά εργασίας. Αλλά η ανεργία δεν μαστίζει, δεν πλήττει αυτή τη στιγμή μόνο τους νέους, αλλά και τους μεγαλύτερους, άνω των 50 ετών για παράδειγμα, ή τις νεαρές μητέρες. Θα μπορούσατε λοιπόν να μας ε, πείτε πώς μπορούμε να προετοιμαστούμε για να αντιμετωπίσουμε και να λάβουμε υπόψη τις ανάγκες αγοράς εργασίας μετά την κρίση και τι προεργασία θα, θα χρειαστεί στο μέλλον, τι προσπάθειες θα χρειαστούν στο μέλλον ώστε να μπορέσουν καλύτερα οι νέοι να προγραμματίσουν την επαγγελματική του σταδιοδρομία ώστε να βρουν μια δουλειά στη θέση εργασίας και να μην χάνουν όλο τους το χρόνο στην αναζήτηση της αγοράς εργασίας. Επίσης έχω μία ερώτηση προς τον κύριο Μασκερίνη. δεν ξέρω αν προφέρω σωστά το όνομά σας. Διάβασα την έκθεσή σας και έχω μερικές ερωτήσεις. Είπατε ότι ο, ο λόγος και τα αίτια είναι πολύ περίπλοκα Ε, και φυσικά χρειαζόμαστε εξατομικευμένη προσέγγιση για την επαναφορά των νέων στην αγορά εργασία, ιδιαίτερα των μακροχρόνιων έργων. Πιστεύετε ότι μπορούμε στην αγορά εργασία πραγματικά να περιλάβουμε τους πάντες. Σα ευχαριστώ και ευχαριστώ εκ των προτέρων τους διερμηνείς που μου, μας χορήγησαν ένα επιπλέον δεκάλεπτο. Θα προσπαθήσουμε να μην το υπερβούμε και να δώσω το λόγο και πάλι στους εμπειρογνώμονές μας, ε, ζητώντας να απαντήσουν μέσα σε τρία λεπτά και διαβεβαιώνοντας ότι αυτή τη φορά θα είναι πιο αυστηρή στην τήρηση του χρόνου. Θα ξεκινήσουμε με τον καλεσμένο μας από την Κρακοβία, τον καθηγητή Γιαρόσουαφ Γκούρνιακ, για τρία λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμη Ευρωβουλευτέ. Δύο ερωτήσεις μου απέφθηναν τα μέλη της Επιτροπής σας. καταρχήν με ρώτησε η Ευρωβουλευτής από την Λιθουανία αν μπορούμε να προβλέψουμε τις ανάγκες αγοράς εργασίας και για να προγραμματίσουμε καλύτερα και τις σπουδέ. Οι δυνατότητε πρόβλεψης είναι πολύ μικρές, γιατί δεν ξέρουμε τι καινοτομίες θα λάβουν χώρα και τι εξελίξεις θα λάβουν χώρα και στην οικονομία. Συνήθω στην οικονομία μπορούμε να προβλέψουμε σε ένα μακρινό ορίζοντα, αλλά αυτό που μπορούμε να πούμε ότι η υψηλή ποιότητα των προσόντων και τη ικανότητα επίλυση των προβλημάτων, η δημιουργικότητα, το ε, πνεύμα συνεργασία, η συλλογική εργασία και η αξιοποίηση των νέων τεχνολογικών είναι όλα αυτά εφόδια και προσόντα που θα πρέπει να χορηγούνται ήδη από το σχολείο. Κάτι που δυστυχώς δεν γίνεται σήμερα. Πολλέ φορές στις έρευνε που κάνουμε με του επιχειρηματίες, με τους εργοδότες, ακούμε από αυτού, ότι είναι ανεπαρκής η προετοιμασία των νέων όχι μόνο για συγκεκριμένα επαγγελματικά προσόντα, αλλά και κάποιες ε, ικανότητες ε, όπως είναι η δυνατότητα εργασίας σε ομάδας. Είναι κάποια στοιχεία που θα πρέπει να τα μαθαίνουν νέοι από το σχολείο. Και θα πρέπει όχι να αλλάξουμε τους καθηγητές κατά ανάγκη, αλλά να ε, καταρτήσουμε τους καθηγητές ώστε να μπορούν να διδάξουν τέτοιου είδους ε, ε, μαθήματα στους νέους. Επίσης, ε, καινοτομίες είναι συνέχεια απαραίτητε και στην οικονομία και στην απασχόληση και στην πολιτική. Τώρα, για το πώς θα προετοιμαστούμε για την εργασία, για την αγορά εργασίας μετά την κρίση και μάλιστα όχι μόνο ε, στους νέους αλλά και σε άλλες ηλικιακές ομάδες. Κατά τη γνώμη μου, τρέφουμε υπερβολικές ελπίδες και έχουμε υπερβολικές προσδοκίες από ε, κάποιες έμεσες παρεμβάσεις ε, και τι προσφέρουμε τους, ε, στους νέους σε μεγάλο βαθμό, ιδιαίτερα σε χώρες ε, του, του Νότου. Γιατί οι νέοι θα πρέπει να ε, αναζητούν μια θέση ε, εργασίας που θα εξασφαλίζει και επαγγελματική δραστηριότητα και κάποιε μελλοντικέ προοπτικές. Δυστυχώ τέτοιε ποιοτικέ εργασίες δεν υπάρχουν. Είναι υπερβολικές λοιπόν οι προσδοκίες. Οπότε θα πρέπει για να βελτιώσουμε την ποιότητα της προσφοράς να επενδύσουμε περισσότερο και στην παιδεία. Από τις εμπειρίες που έχουμε στην Πολωνία καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η αφιέρωση των πόρων και των εθνικών και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου θα πρέπει να επικεντρωθεί στη βελτίωση της, των δυνατότητων σπουδών που προσφέρονται και των δυνατότητων κατάρτισης στους ανέργους. Γιατί με την καλύτερη παιδεία θα κρατήσουμε τους νέους πολύ πιο κοντά στις ανάγκες αγοράς εργασίας. Θα πρέπει όμως ε, να κάνουμε κάποιες αλλαγές που θα πρέπει να έχουν στόχο και την βελτίωση της οικονομικής κατάστασης για να βελτιώσουμε και την ανεργία. Ο κύριος Μίλλερ από, ε, από, τον από τον Γερμανικό Οργανισμό. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Κοιτάξτε, ακούσαμε διάφορε ιδέε για την ε, κινητικότητα την οποία πρέπει να έχουμε στην Ευρώπη. Θα πρέπει όμω η προσέγγιση μα να λάβει υπόψη τη και την οικονομική κατάσταση. Δεν συμφωνώ πάντω με την άποψη που ακούστηκε. Η κινητικότητα σε κάθε περίπτωση θα αποτελεί προσωπική επιλογή του νέου και ουσιαστικά εξαρτάται από την προσωπική κατάσταση του ανθρώπου και από τις δυνατότητες που του ανοίγονται σε μια συγκεκριμένη χώρα κάπου αλλού. Εμείς πάντα είχαμε ανθρώπους οι οποίοι ερχόντουσαν, μετανάστευαν προς τη χώρα μου, τη Γερμανία. Εξαιτίας της α, διάρθρωσης και της κατάστασης αγοράς-εργασίας στη χώρα μου. Κάτι τέτοιο ενδεχομένω να μην συμβαίνει σε άλλες χώρες. Αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι υπάρχουν αρκετοί Γερμανοί που πηγαίνουν στο εξωτερικό και έχουμε αρκετούς ξένους που έρχονται από την Ελλοδαπή για να εργαστούν στη Γερμανία και γνωρίσαμε κι εμείς κάποιες μεταβατικές περιόδους Νομίζω όμως ότι αντιτίθενται στην ιδέα ότι η κινητικότητα είναι πάντα κάτι το θετικό. Όπου είδαμε μεταβατικές περιόδους, είδαμε ότι υπήρχαν πολύ περισσότεροι νέοι οι οποίοι φεύγαν από τη χώρα, παρά, παρά νέοι οι οποίοι φτάνανε στη χώρα αυτή για να εργαστούν εκεί. Δεν συμφωνώ λοιπόν με την παρατήρηση που εκφράστηκε και να πω και κάτι ακόμα. Υποβλήθηκε μία ερώτηση για, τα βασικά, για τις βασικές απαιτήσει. Νομίζω ότι είναι δύο. Πρώτον, καταρχάς οι νέοι πρέπει να πιστούν θα πρέπει να θέλουν οι ίδιοι να πάνε σε κάποια γραφεία ενεργεία, σε κάποιες αρμόδιες εθνικές υπηρεσίες και να καταχωρηθούν στα εκεί μητρώα. Διαφορετικά δεν θα καταφέρουμε ποτέ να τους εντοπίσουμε. Ενδεχομένως να εντοπίζονται σε κάποιες μελέτες που γίνονται σε κοινοτικό επίπεδο, Όπω η ευρωπαϊκή έρευνα για την αγορά εργασία, αλλά αν πραγματικά θέλουν να μην είναι απλώ στατιστικά δεδομένα, αλλά να βρουν τελικά μια θέση εργασία, θα πρέπει να απευθυνθούν στι αρμόδιε εθνικέ υπηρεσίε, στα αρμόδια εθνικά κέντρα. Βέβαια, πώ θα γίνει κάτι τέτοιο αν οι νέοι δεν έχουν κάποια προσδοκία ότι θα βρουν μια δουλειά. Είναι πολύ δύσκολο να του πείσουμε να ενταχθούν στο σύστημα αυτό. Και βέβαια, πρωταρχικά χρειαζόμαστε προσφορά εργασία. Αυτό είναι το πολύ δύσκολο. Τι γίνεται δηλαδή στι περιπτώσει εκείνες, στι χώρε εκείνε που δεν υπάρχουν θέσει εργασία, που δεν υπάρχουν καινέ θέσει, που δεν προκύπτουν καινέ θέσει. τι θα γίνει. Θα πρέπει το δημόσιο να χρηματοδοτήσει θέσει εργασία και ακόμα και να γινόταν αυτό. Πώ θα μπορούσε να λειτουργήσει στην πράξη. Πολύ συχνά βλέπουμε ότι έχουμε όλο και περισσότερε περιπτώσει που έχουμε μικροεπιχειρήσεις, μικρομεσαίε επιχειρήσει ε, στα κράτη-μέλη και όχι τόσο πολλέ θέσει εργασία στο δημόσιο. Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Μασιμιλιάνο Μασκερίνη, λέει πρόεδρο. Σα ευχαριστώ. Όντω στην έκθεσή μου λέω ότι ε, τα αποτελέσματα τα οποία έχουμε για την ανεργία τελικά έχουν να κάνουν τόσο με το θεσμικό πλαίσιο, την κατάσταση της χώρας και την προσωπική κατάσταση των ε, νέων. Και βέβαια αυτοί που ε, συγκεντρώνουν, αν θέλετε, αρνητικά χαρακτηριστικά σε όλες αυτές τις κατηγορίες, η κατάστασή τους είναι όλο και πιο δύσκολη. Λέμε λοιπόν ότι ε, η εξατομικευμένη προσέγγιση είναι η πιο επιτυχής τελικά και μέσω της εξατομικευμένης προσέγγισης έχουμε ουσιαστικά μία προσέγγιση που αναγνωρίζει τις πραγματικές ανάγκες των νέων και προτείνει στους νέους αυτούς μία λύση η οποία προσαρμόζεται στα προβλήματά τους και στις ανάγκες τους. Γιατί καταλαβαίνετε ότι μία νέα μητέρα και ένας άνδρας ανειδίκευτος έχουν διαφορετικές ανάγκες και κατά διαφορετικό τρόπο θα πρέπει να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Βέβαια δεν μπορούμε να καλύψουμε τους πάντες. Γιατί καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν και ορισμένοι οι οποίοι δεν μπορούν τελικά να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, άλλοι πάλι δεν επιθυμούν, άλλοι πάλι δεν συμμετέχουν στα προγράμματα αυτά και αυτό είναι και μια σημαντική πρόκληση, πώς θα καταφέρουμε να έχουμε πρόσβαση σε περισσότερους νέους. Πρέπει επίση να σα πω ότι η εγγύηση για του νέου δεν γίνεται μία νυχτή να υλοποιηθεί σε όλε τι χώρε. Γιατί ουσιαστικά αυτό το οποίο απαιτείται είναι μία βαθμιαία εφαρμογή τη σε διαφορετικά στάδια. Υπάρχουν ορισμένε χώρε που ήδη έχουν προχωρήσει αρκετά, όπω για παράδειγμα η Φιλανδία και το φιλανδικό μοντέλο, και άλλε πάλι που υπολείπονται. Όσον αφορά τώρα τα προγράμματα κατάρτισης, στην επόμενη έρευνα την οποία θα δημοσιοποιήσουμε, λέμε ότι υπάρχουν ορισμένα κράτη-μέλη, κυρίως στη Νότια Ευρώπη, όπου έχουμε νέους οι οποίοι ένα χρόνο μετά την αποφύτισή τους βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκτός προγραμμάτων μαθητείας ή κατάρτισης και ένα πολύ μικρό μόνο ποσοστό καταφέρει να ενταχθεί στην αγορά εργασίας και αναφερόμαστε σε άτομα τα οποία έχουν πανεπιστημιακή εκπαίδευση άτομα τα οποία λογικά θα πρέπει να ενταχθούν πιο εύκολα στην αγορά εργασία. Για ποιο λόγο όμω συμβαίνει κάτι τέτοιο, Υπάρχει αντιστοιχία ανάμεσα στι ανάγκε τη αγορά και τι δεξιότητέ του, αυτό είναι ένα ζήτημα. Το άλλο πάλι είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι θα πρέπει να αυξήσουμε περισσότερο τις υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού προς τους νέους. Θα πρέπει οι νέοι να κάνουν συνδετές αποφάσεις όσον αφορά το μέλλον τους, προφανώς να γνωρίζουν ποιες είναι οι επιθυμίες τους, αλλά να γνωρίζουν επίσης και ποιες είναι οι επιπτώσεις μιας θετικής ή αρνητικής επιλογής. Αν θέλετε, οι επιλογές θα πρέπει να είναι πιο ενημερωμένες, πιο συνειδητές, τελικά να αναποκρίνονται πολύ περισσότερο στην πραγματικότητα και στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς απασχόλησης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. από την Φιλανδία. Έχετε το λόγο τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι πολλά ερωτήματα τέθηκαν στο φιλανδικό μοντέλο και δεν μπορώ να απαντήσω σε όλες. Αναφέρομαι, αν θέλετε σας ε, παροτρύνω να δείτε την ιστοσελίδα ε, του, των εγγύσεων για τους νέους. Επίσης, ε, εκεί θα βρείτε ορισμένες εκθέσεις και παρουσιάσεις για το φιλανδικό μοντέλο. Αν θέλετε περισσότερες λεπτομέρειες, σας παραπέμπω σε αυτή την ιστοσελίδα. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στα γενικά ερωτήματα. Το ένα ήταν ποιε είναι οι βασικέ προϋποθέσεις για να λειτουργήσει αυτό το Ταμείο Εγγύηση των Νέων με γνώμονα τι ανάγκε των νέων. Τρία σημεία κατά τη γνώμη μου. Πρέπει να υπάρχουν οργανισμοί απασχόλησης που θα λειτουργούν σωστά σε τοπικό επίπεδο. Και γι' αυτό το λόγο χρειάζονται πόροι για να γίνει σωστή δουλειά στα μέτρα των νέων. Δεύτερον, το εκπαιδευτικό σύστημα μπορεί να προσφέρει επαγγελματική κατάρτιση στα μέτρα της αγοράς εργασίας και τρίτον η δέσμευση και η συνεργασία με τους εργοδότες ώστε να υπάρχουν θέσεις απασχόλησης για τους νέους. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Τώρα το πρώτο ερώτημα που τέθηκε ήταν οι δραστηριοτικές αλλαγές για να, βοηθήσει, ε, να βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αυξήσουν την απασχολησιμότητα των νέων. Τι κίνητρα μπορούμε να προτείνουμε. Πρέπει να γίνουν πολλές μεταρρυθμίσεις σε πολλά κράτη-μέλη σε αυτό το τομέα. Καταρχήν, ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν οικονομικό κίνητρο να απασχολήσουν τους νέους θα μπορεί να είναι είτε επιχορηγήσεις, είτε φορολογικά κίνητρα ή άλλα κίνητρα. Επίσης, θα πρέπει να δούμε και το εργατικό δίκαιο. Αυτό το θέμα είναι ευαίσθητο, αλλά συχνά είναι κόλλημα στην πρόσληψη νέων ατόμων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γι' αυτό χρειαζόμαστε ε, νόμους εργατικούς ασφαλείς και ευέλικτους. Επίσης, και το θέμα των μισθών παίζει σημαντικό ρόλο. Αυτό το θέμα όμως είναι πολύ ευαίσθητο και είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή να καταλήξουμε σε συμπεράσματα. Αν έχω ακόμα λίγο χρόνο, θα ήθελα να απαντήσω σε ένα σημαντικό ερώτημα για το πώς ε, αντιμετωπίσουμε εκείνους που, βρίσκονται, που είναι αποκλεισμένοι. Υπάρχει ένα μοντέλο το οποίο αναπτύσσεται στη Φιλανδία αυτή τη στιγμή και θα επεκταθεί σε όλη την επικράτεια. Είναι ένα μοντέλο ε, σύμφωνα με το οποίο οι πλησιάζουν τους αποκλεισμένους νέους ε, βοηθώντας τους να καταρτιστούν. Υπάρχουν ορισμένα εργαστήρια σχετικά όπου μπορούν ε, να δουλέψουν, να κάνουν πρακτική άσκηση οι νέοι για να βρουν μια δουλειά αργότερα. Ένα τρίτο σημείο όσον αφορά τον αποκλεισμό των νέων σημαντική είναι η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των παραγόντων ε, στο εγγύηση των νέων, επειδή οι οργανισμοί απασχόλησης θα πρέπει να γνωρίζουν ποιοι είναι οι νέοι που έχουν τον κίνδυνο να αποκλειστούν. Υπάρχει σχετική νομοθεσία, αλλά πρέπει να δούμε πώς ε, θα ενισχύσουμε την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των ενδιαφερομένων. Για παράδειγμα, ποιοι έχουν ολοκληρώσει την στοιχειώδη εκπαίδευση και μπορούν να καταρτιστούν και κατόπιν χρειαζόμαστε πληροφορίες για τα συγκεκριμένα άτομα. Βεβαίως υπάρχουν και άλλες λεπτομέρειες. Ευχαριστώ πολύ. δώσω τώρα το λόγο στον εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Φόρουμ για τους Νέους. Ευχαριστώ. Από όλα τα σχόλια και τις ερωτήσεις διαπιστώνουμε την περιπλοκότητα αυτού του θέματος τη ανεργίας των νέων. Το θέμα είναι να βρούμε ποιο κάνει τι, ποιο είναι υπεύθυνο γιατί και πού μπορούμε να δραματίσουμε κάποιο ρόλο και εμεί, εκπρόσωποι των νέων. Θέλουμε μια διακλαδική, διατομεακή προσέγγιση, ολιστική, που θα συνδέει την παιδεία με την αγορά εργασία και θα επικεντρώνεται και στη μετάβαση. Θέλουμε ποιοτική εκπαίδευση. Μια παιδεία που θα έχει και τυπικά και ε, μη τυπικά στοιχεία, γιατί υπάρχουν κάποια εφόδια και δεξιότητες που δεν τα λαμβάνω αυτή τη στιγμή από την ε, επίσημη εκπαίδευση, αλλά που είναι απαραίτητα για την αγορά εργασίας. Θα πρέπει λοιπόν ε, να μπορέσει κανείς να αποκτήσει αυτά τα εφόδια, όπως είναι να, μπορεί να εργάζεται σε ομάδες, να μπορεί να εκφράζεται ωραία, ε, είναι σημαντικά όλα αυτά τα θέματα, κάποιες κοινωνικές δεξιότητες. Θα πρέπει ο νέος όταν θέλει ξεκινήσει σπουδές του να ξέρει ε, τι τον περιμένει μετά στην αγορά εργασίας. Πριν τον επαγγελματικό προσανατολισμό λοιπόν ε, να υπάρχουν δυνατότητες ενημέρωση των νέων για τις διάφορες σπουδές. Γιατί μερικέ φορέ πηγαίνουμε εμεί στην, στην ύπεθρο τη Εστονία και δίνουμε τέτοιε συμβουλέ επαγγελματικού προσανατολισμού γιατί δεν υπάρχουν τέτοιε υπηρεσίε. Επίση, μεταβατική περίοδο που θα πρέπει να εξαρτάται από τι δυνατότητε κινητικότητα, Θα επικεντρωθούμε ε, σε αυτό το θέμα και τι δυνατότητε μεταβίβασης των δικαιωμάτων, φορητότητε. Ε, να μπορεί κανεί να κινείται ελεύθερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να ε, μεταφέρει και τα διάφορα δικαιώματα που αποκτά σε κάθε κράτος. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και άλλο ζήτημα της μεταβατικής περίοδου είναι ποιοτικά στάζ ποιοτικέ περίοδοι μαθητείας. Έχουμε κατάλληλη νομοθετική ρύθμιση και κάτι τέτοιο και αν όχι γιατί. Τι ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολύ σημαντικό, γιατί εμείς είμαστε υπέρ των νομοθετικών μέτρων που πρότεινα το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο για την εγγύηση των νέων. Αυτό είναι φυσικά ένας από τους μηχανισμούς, δεν είναι πανάκια, δεν είναι θαυματουργή λύση για όλα, αλλά είναι υπόδειγμα για κάτι που χρειαζόμαστε και θα πρέπει να αξιοποιηθεί πλήρως και να μεταφερθεί όπου γίνεται. Κυρία Σάια, λέτε ποια είναι η βάση για όλα αυτά χρηματοδότηση, αφοσίωση και ανάμιξη. Ανάμιξη εμπλοκή των νέων. Από τη στιγμή που ε, οι νέοι είναι άμεσα ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αναμειγνύονται. Επίσης προσήλωση, δέσμευση των ενδιαφερομένων ε, και κυρίως του κράτους και φυσικά χρηματοδότηση. Αυτές είναι οι τρεις βάσεις, η ακρογωνία, η λύθη ε, του Ταμείου Εγγυήσεων για τους νέους. Και επίσης μία παιδεία που θα αναπτύσσει και το επιχειρηματικό πνεύμα. Να ξέρει ο κάθε νέος τι σημαίνει γίνομαι επιχειρηματίας. Και επίσης ε, να ξέρει ότι αν κάποιος δεν θέλει να γίνει επιχειρηματίας δεν σημαίνει ότι στιγματίζεται. Αλλά να δίνει τη δυνατότητα σε αυτόν που έχει τέτοιες ανάγκες να τις ικανοποιήσει και να τις αναπτύξει το δυναμικό του. Φυσικά ε, να επικεντρωθούμε στην ποιότητα. Ε, να επενδύσουμε στην ανάπτυξη, να επενδύσουμε στους νέους και να δούμε πού μπορούμε να δημιουργήσουμε οικονομική μεγέθυνση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά λοιπόν είναι σημαντικά. Και τέλος, πέρυσι που είχαμε το Ευρωπαϊκό Έτος Ενεργούς Γύρανσης, κάναμε κάποια μελέτη. Δεν θέλουμε οι νέοι να εκτοπίσουν από την αγορά εργασία του ηλικιωμένου, γιατί κάποιο που συνταξιοδοτείται αφήνει μια θέση απασχόληση που δεν μπορεί να πληρωθεί από ένα νέο κατά ανάγκη. Θέλουμε λοιπόν να υπάρχει αλληλεγγύη μεταξύ των γενναιών και αυτό το θέμα δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ που τηρήσατε το χρόνο ομιλία. Θα εξετάσουμε το σχέδιο έκθεση της ε, συναδέλφου Ξηλεύσκα στην ε, συνεδρίαση της 22ης-23ης της Απριλίου. Λέω στην κυρία Αντζελίλη και στους υπολείπους ότι όσα έγγραφα δεν έχουν ε, δοθεί Μάλλον έχουν δοθεί τα έγγραφα της Eurofound, θα σας δοθούν σήμερα το βράδυ ή αύριο. Τα υπόλοιπα έγγραφα θα τα βρείτε στην ιστοσελίδα της Επιτροπής μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους προσκεκλημένους μας για τις παρεμβάσεις τους και θα ήθελα να σα δώσω ραντεβού στι 3 το μεσημέρι για τη συνέχιση της συνεδρίασή μας υπό την Προεδρία του κυρίου Αντιπροέδρου Τόμας Μάν. Σας καλώ όμω τώρα έξω από την αίθουσα αυτή να γιορτάσουμε την πολύ επικοδομητική συνεργασία που είχαμε με την Ιωάννα έξω από την αίθουσα λοιπόν για να πω